Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν να αρχίσουμε εκ νέου τις εργασίες μας, θα ήθελα να εκφράσω την παθιά μου ανησυχία για την καταδίκη σε 38 χρόνια φυλακής και σε μαστίγωμα της του Σουτουτέ, δικηγόρο στο Ιράν, η οποία είχε κερδίσει το βραβείο Ζαχάροφ 2012. Το μόνο της φταίξιμο είναι ότι αγωνίστηκε για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνιού καταδικάζω κάθετα αυτή την παράλογη ποινή και πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνείτε μαζί μου στο να ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωση της νεσρή. Επίσης, την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω ε, τα συλληπιτήρια μας οικογένειας των 76 θυμάτων ε, από τις βροχοπτώσεις στο Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ανθρωπιστική βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η έκτακτη ανάγκη. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι η τελευταία σύνοδος της Ολομέλειας πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έργο σας, για τη δέσμευσή σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μου. Η δουλειά μου είναι να θέτω στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που οργανώσαμε πολλές συνεδριάσεις με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για να δείξουμε ότι βρισκόμαστε στο επίκεντρο του μέλλοντος της Ευρώπης. Πιστεύω ότι όλοι εδώ θέλουν περισσότερη εξουσία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περισσότερες αρμοδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική στην Ευρώπη. δυόμιση χρόνια όλοι μας εργαστήκαμε μαζί και προσπάθησα να τηρήσω ουδέτερη στάση και παράλληλα προσπάθησα να επερασπίσω τα δικαιώματα και τη σημαντική θέση του καθενός σας. Ανεξάρτητα από την πολιτική ομάδα ή από το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκει κανεί. Προσπάθησα να σεβαστώ όλους του ευρωβουλευτέ. Προσπάθησα να επιτρέψω στον καθένα να εκφράσει τη θέση του. Αν έκανα κάπου λάθος, ζητώ συγγνώμη. Και φυσικά πάντοτε μπορούν να γίνουν και λάθη όταν εργαζόμαστε σε τέτοια ζητήματα, αλλά πάντοτε προσπάθησε να είμαι έντιμος και πιστός απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο την... έχω την τιμή να προεδρεύω, όντας εκλεγμένος από την πλειοψηφία ημών. Προσπάθησα να γίνουν σεβαστοί κανόνες, προσπάθησα πάντοτε να τους ακούω όλους σε αυτά τα δυόμιση έτη είχα την τιμή να υπογράψω εκατοντάδες φορές τα αποτελέσματα του έργου σας. Είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα και προσπαθήσαμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Εγώ πάντοτε βέβαια προσπαθούσα να δρω έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγχει την Κομισιόν και όχι να ελέγχεται από την Κομισιόν και να είναι πάντοτε με ψηλά το κεφάλι απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα. Προσπάθησα επίσης να τηρήσω όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβα απέναντί σας την ημέρα της εκλογής μου, όταν παρουσίασα την υποψηφιότητά μου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι για μένα ήταν δύο έτη, δυόμιση έτη εξαιρετικά και πάλι Ευχαριστώ όλους εσάς για όσα πράξατε. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλες τις επικρίσεις, όλες τις επιφυλάξεις. Ακόμη και που με, όσα με αφορούσαν και απέναντί μου. Και άκουσα και όσους είχα και αντίθετες θέσεις από μένα. Μου έδωσαν χρήσιμες συμβουλές, ποτέ δεν υποτίμησα τις επικρίσεις ούτε θέσεις διαφορετικές από τις δικές μου. Προσπάθησα να είμαι ένας αμερόληπτος, ένας ανεξάρτητος πρόεδρος. Προσπάθησα να αξιοποιώ το έργο όλων σας. Και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσω και όλο το προσωπικό και όλους τους διερμηνείς και τους ευχαριστώ από καρδιάς για την υπηρεσία που προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που εμείς εκπροσωπούμε. Δίχως αυτούς ε, δεν ε, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους ε, στόχους που έχουμε θέσει και κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας συνόδου. Σας ευχαριστώ όλους, καρδίας, για το έργο σας. και πάντοτε θα είστε στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ όλους. Σε πολλές γλώσσες. Λέει ευχαριστώ πρόεδρος. Dichiaro Άρχεται η συνεδρίαση που διακόπηκε στις 4 Απριλίου. Τα πρακτικά θα έχουν διανεμηθεί Υπάρχουν παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητέ Αντώνιο, δεν θέλω να χαλάσω αυτή την ε, επίσημη στιγμή. Υπέβαλε ωστόσο μία ένσταση βάση του άρθρου 184 δύο φορές ουδής αντέδρασε στο αίτημά μου. Μήπως θα μπορούσες να, να ζητήσεις από την γραμματεία του να μου απαντήσουν στην ένσταση που υπέβαλα. Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς πρόβλημα είχατε. Έτσι. Ε, είχα υποβάλει ένα αίτημα όταν κάποιος υποβάλει ένσταση βάσει του αντίστοιχου άρθρου και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό μέσα σε 24 ώρες πρέπει να, λάβω γραπτή, πρέπει να λάβει γραπτή απάντηση. Μέχρι τώρα, εδώ και 15 μέρες δηλαδή, κανείς δεν απάντησε στο ερώτημα που υπέβαλα. Θα φροντίσουμε να λάβετε την απάντηση γρήγορα. Άλλε παρατηρήσει για τα πρακτικά. Θεωρούμε ότι εγκρίνονται κατά συνέπεια. Μετά την εκλογή του κυρίου Ιβάρη Πάνταρ ως βουλευτού στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Εσθονία, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χειρία τη θέση από 4η Απριλίου, σύμφωνα με τον κονισμό Οι αρμόδιε αρχέ τη Εστονία ανακοίνωσαν ο κ. Χάνε Χάνσο εκλέγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντικαθιστώντα τον κ. Παντάρα από τι 4η Απριλίου. Το καλωσορίζω τον συνάδελφο και θυμίζω ότι βρίσκεται στο Κοινοβούλιο και τα όργανα του βάση με πλήρη δικαιώματα. Έλαβα από τους σοσιαλιστές αιτήματα ορισμού σε επιτροπές και αντιπροσωπείες που θα, βρεθούν, που θα βρούμε στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μέχρι την έγκριση των πρακτικών, οι αλλαγές αυτές θα θεωρηθούν ότι εγκρίθηκαν. Η ε, συνταγματική επιτροπή πρότεινε μια μηνέα του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερο, δεύτερη παύλα και το άρθρο 149 149α παράγραφος 2 του κανονισμού. Τα κείμενα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας και θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης. Οι ερμηνείε που θεωρούν, θα θεωρηθούν ότι εγκρίθηκαν εάν μέσα σε 24 ώρες καμία πολιτική ομάδα ή ε, ένα αριθμό βουλευτών δεν αντισταθούν σε αυτό. Σύμφωνα με τι διαβουλεύσει που προβλέπει το άρθρο 234 του Χρηματοοικονομικού Ενωσμού, η η Επιτροπή Ανάπτυξη και η Επιτροπή Προλογισμών μου μεταβίβασαν την κοινή του θέση για την επέκταση του Ταμείου τη Ένωση για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που δημιουργήθηκε με απόφαση τη Επιτροπή στι 11 Ιουλίου 2014 και που λήγει στι 30 Ιουλίου 2019. Η κοινή θέση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα τη Ολομέλεια και θα δημοσιευθεί στα πρακτικά τη σημερινή συνεδρίαση αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει από πολιτική ομάδα ή από τα μέλη που φτάνουν το χαμηλό όριο μέσα 24 ώρε, θα μεταβιβάσω επίσημα την κοινή αυτή θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενημερώνω το σώμα ότι μετά την, τις 4, 24 ε, Απριλίου υπέγραψε σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού μαζί με, το, με την Προεδρία του Συμβουλίου τα πρακτικά τη, τη νομοθετική διαδικασία και ενημερώνω το Σώμα ότι μαζί με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου θα υπογράψω 19 νομοθετικά κείμενα που εγκρίθηκαν με την, με την ε, ε, συνήθη νομοθετική διαδικασία. Οι τίτλοι των ε, νομοθετικών αυτών πράξεων θα δημοσιευθούν στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης. Το τελικό κείμενο της ε, διάσκεψης των Προέδρων ε, που εγκρίθηκε με βάση το άρθρο 49 και έχει διανεμηθεί σε όλους. Μετά από διαβουλεύσεις με τις πολιτικές ομάδες θέλω να ενημερώσω το Σώμα για τις ακόλουθες προτάσεις αλλαγής της τελικής μερίσης διατάξεως. Μισό. Μισό λεπτό. Το εγκρίνουμε και μετά σας δίνω το λόγο. Δηλώσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τη Επιτροπή για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 10η Απριλίου 2009 για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνουν την Τρίτη το πρωί, πρώτο σημείο. Υπάρχουν αντιρρήσει, Όχι. Ο κύριος Βάιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και αναφέρομαι στον κανονισμό στο 116α 3. Πρόκειται για μια κοινή συνεδρίαση τη επιτροπή Αναφορών η οποία έλαβε χώρα ε, κατόπιν αιτήματο των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τη Exxon, ε, Mobile, ε, σε ό,τι αφορά ειδήσει για, την, για, για ψευδείς ειδήσει για το κλίμα. Και εκλήθηκε λοιπόν η Exxon Mobile στο, στη συνεδρίαση αυτή. Έχει έξι μπάτζες για λόμπινγκ. Η Mobile δεν ε, ήρθε όμως στη συνεδρίαση και χρησιμοποίησε μια πρόφαση για μια δίκη η οποία έλαβε χώρα. Το 116α όμως καταδεικνύει ότι μια οργάνωση η οποία έχει διαπίστευση ως ε, λόμπι και δεν ε, χρησιμοποιεί παρκώς τις, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, θα πρέπει να τις αφαιρεθούν λοιπόν αυτές οι διαπιστεύσεις. Απεστάλλει λοιπόν επιστολή προς την Mobile Θα απαντηθεί αυτή, η επιστολή, θα αποσυρθούν αυτές οι διαπιστεύσεις ή πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι πλέον καθήκον του Προέδρου ή ενδεχομένως και του Κοινοβουλίου στην τρέχουσα θετία. Ευχαριστώ. Δεν είναι αρμοδιότητα του Προέδρου. Το εξετάζει το θέμα ο Γενικός Γραμματέας. Ε, τέθηκε και στην τελευταία διάσκεψη των Πρόεδρων και θα σα ενημερώσω μόλι ληφθεί η απόφαση. Ο κ. Μαριάς. η αναγνώριση εκ μέρου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της γενοκτονίας των ελλήνων του πόντου αποτελεί πλέον μια ιστορική αναγκαιότητα πολύ δε περισσότερο φέτος που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γενοκτονία των ελλήνων του πόντου. το 1919 μετά την απόβαση του κεμάλ πασά στη Σαμψούντα του πόντου οι νεότουρκοι προχώρησαν σε μαζικές σφαγές και δολοφονίες Αν δεν μου πείτε περί τίνος πρόκειται, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το ερώτημά σας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιο είναι το έτοιμά σας και μετά θα σας δώσω το λόγο. Σας έχει ήδη ενημερώσει η ομάδα μας. Το Πρώτα μιλάω εγώ, μετά εσείς η ομάδα των συντηρητικών ζήτησε να προστεθεί δήλωση της Επιτροπής για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων ποντίων μεταξύ 1914 και 1923. Σαν τελευταίο σημείο στην, στις παρεμβάσεις του ενός λεπτού, η συζήτηση θα κλείσει με ένα ψήφισμα. Ο κύριος Μαριάς, εξηγήστε μας τώρα κύριε Μαριά, γιατί υποβάλλετε το αίτημα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η αναγνώριση εκ μέρους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου της γενοκτονίας των ελλήνων του πόντου αποτελεί πλέον μια ιστορική αναγκαιότητα πολύ δε περισσότερο φέτος που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γενοκτονία των ελλήνων του πόντου. το 1919 μετά την απόβαση του κεμάλ πασά στη σαμψούντα του πόντου οι νεότουρκοι προχώρησαν σε μαζικές σφαγές και δολοφονίες χιλιάδων ελλήνων του πόντου άνδρες γυναίκες και παιδιά ήταν τα θύματα της γενοκτονίας που ξεπέρασαν τις. τριακόσια πενήντα χιλιάδες. εκτελέσεις βιασμοί καταναγκαστικά έργα στα τάγματα εργασίας οδήγησαν στο θάνατο τους ποντίους αδελφούς μας. και πρόκειται για γενοκτονία γιατί οι έλληνες του πόντου δολοφονήθηκαν επειδή ήταν έλληνες και χριστιανοί. ζητούμε λοιπόν σήμερα κύριε πρόεδρε δευτέρα να προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της κομισιόν με θέμα αναγνώριση της γενοκτονίας των ελλήνων του πόντου που έλαβε χώρα το διάστημα 1914 1923 και να εκδοθεί ψήφισμα. επιπλέον ζητούμε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για το αίτημά μας αυτό και καλούμε τους συναδέλφους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου να στηρίξουν αυτή την πρότασή μας ως ένα ιστορικό χρέος ιδίως φέτος που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γενοκτονία των ελλήνων του πόντου. ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που θέλει να λάβει το λόγο κατά της πρότασης. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία το αίτημα τη ομάδα των συντηρητικών για να προσθεθεί δήλωση τη Επιτροπή για την αναγνώριση τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σαν πρώτο σημείο μετά τι παρεμβάσει του ενό λεπτού. Η συζήτηση θα κλείσει με ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Il voto Πέρας ψηφοφορίας. Η πρόταση απορρίπτεται. Τη Δευτέρα η ομάδα της αριστεράς ζήτησε δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις απειρές και τα δικαιώματα καθώς και την ακαιρεότητα των πληροφοριοδοτών την περίπτωση Τζούλιαν Ασάζ να συζητηθεί μαζί με την έκθεση της κυρία Ζωζία για την προστασία των ατόμων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαιώματος της, του νοσιακού δικαίου. Δίνω το λόγο στην κυρία Τόρες για να παρουσιάσει το αίτημα της ομάδας της. Ευχαριστώ δεν είναι το να λέει κανείς την αλήθεια δεν είναι αδίκημα και πρέπει να προστατεύεται. Ο κύριος Ασάνζ διώκεται από τις Ηνωμένε Πολιτείε γιατί παρουσίασε τι έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο Γκουαντάναμο και το Ιράκ. Εμείς πρέπει να προσφέρουμε εγγυήσεις ότι δεν θα επιστραφεί στι ΗΠΑ όπου μπορεί να βασανιστεί. Η επιστροφή του, όπω αναφέρεται, αναφέρει ο ίδιο, αποτελεί κίνδυνο για τη φυσική του ακαιρεότητα και παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει θέση με τη μεριά τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και του κράτου δικαίου. Ζητούμε να συμπεριληφθεί στην μερίσια διάταξη το θέμα αυτό και θέλουμε να να ψηφιστεί με ονομαστική πληροφορία. Παρακαλώ να σεβαστούμε την ελευθερία και την ακαιρότητα του Τζούρινα Σάραντζ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τόρες. Κάποιος θέλει να λάβει το λόγο κατά. Παρακαλώ. Κατά. Please, you the floor. Παρακαλώ. the Greens, we do... Οι εμείς ω πράσινοι θέλουμε σε, ξεχωριστό σημείο συζήτηση για την υπόθεση του κυρίου Ασάντζ. Φοβόμαστε, φοβόμαστε πολύ το θέμα της έκδοσής του στις ΗΠΑ, αλλά θέλουμε αυτό να αποτελέσει ξεχωριστό σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πρόεδρε, ω δικηγόρος υπέβαλα την πρώτη υπόθεση που έγινε δεκτή στην Ευρώπη κατά των βασανιστήριων και της βάρβαρης μεταχείρισης των κρατουμένων στον Κοντάναμο. Αυτό ήταν σε... Εμείς συζητούμε σήμερα ένα γενικό θέμα, την προστασία των ατόμων που καταγγέλουν. Άλλο είναι να περάσουμε μια ειδική περίπτωση μια γενική περίπτωση. Δεδομένης της νομιμότητας που έχω λόγω της υποστήριξής μου στην περίπτωση του Γκαντάναμου, Έχω, ε, είμαι κατά της πρότασης να εντάξουμε ένα ατομικό στοιχείο, μια ατομική περίπτωση στη γενική συζήτηση. Ψηφίζουμε την πρόταση της ομάδας αριστεράς να προστεθεί στη συζήτηση για την, ε, υπό, για την, για προστασία των ατόμων που καταγγέλουν ε, βίες κατά της Ένωσης και την περίπτωση του Julian Assange. Άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστικά. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται η πρόταση. Για την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζήτησε η ψηφοφορία για την έκθεση Γκρέσλε για τι ε, έρευνε τη Όλαφ και τη συνεργασία με, τον, με το Ευρωγραφείο του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα να αποσυρθεί. Παρακαλώ, κύριε Γκρέσλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο αιτήσει ε, για, την για την έκθεση αυτή, για το, την ε, ΦΕΑ περιοχή, σε ό,τι αφορά τα ε, γραφεία των ευρωβουλευτών χωρί άρση τη ασυλίας. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση μόνο εφόσον επιτρέπεται αυτό από τον βουλευτή. Οι ευρωβουλευτέ λοιπόν δεν μπορούν να είναι σε χειρότερη θέση από την εθνική εθνικοί βουλευτέ. Η Όλαφ προφανώ και έχει πρόσβαση στα τεκμήρια αυτά τη δίκηση σε περίπτωση που υπάρχει υποψία απάτη. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ιστορία θα έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στο Κοινοβούλιο που θα πρέπει να την ψηφίσει τελικά το επόμενο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό ζητώ αναβολή τη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο. Αν ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο, είμαστε μια χαρά γιατί δεν έχει διαμορφωθεί θέση στο Συμβούλιο για την νομική αυτή θέση. Και αν απορριφθεί αύριο η πρόταση αυτή, τα πράγματα θα επιδεινωθούν έτσι περαιτέρω. Γι' αυτό λοιπόν σας ε, ζητώ αναβολή προκειμένου να ασχοληθεί με το θέμα αυτό το νέο κοινοβούλιο. Ο για να μιλήσει κατά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, θεωρώ ότι δεν είναι ε, αποδεκτή αυτή η πρόταση αλλαγή τη τροποποίηση τη ημερήσια διατάξη από την αρχή. Για τον κανονισμό τη ΟΛΑΦ είχαμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε κατεπηγόντω. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση και τη δουλειά του ΟΛΑΦ και τη ΕΠΟ, θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια μέχρι το 2020. Η τελευταία αναθεώρηση πήρε 7 χρόνια, δεν έχουμε τόσο χρόνο. Το ΕΛΚ λοιπόν θέλει να αλλάξει την ημερήσια διατάξη γιατί δεν υπάρχει πλειοψηφία στην Επιτροπή για την τροπολογία της. Αυτό είναι μη δημοκρατικό. Αντί να κοιτάμε λοιπόν αυτή την τροπολογία, θα πρέπει να κοιτάξουμε τις συγκεκριμένες υποψίες απάτης και ατασταλιών, τι θα γίνει και τι πρόσβαση θα έχει όλα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει ίση αντιμετώπιση και επειδή είναι κατεπήγον το θέμα αυτό, και δεν μας πείθουν οι λόγοι αντίθετα. Παρακαλώ όλους τους ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν την αλλαγή στην ημερήσια τέταξη. γιατί αν παραταθεί αυτή η κατάσταση θα συνεχιστούν οι απάτες και όχι μόνο στο γραφείο των ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ. Να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση του ΕΛΚ για να αφαιρεθεί από την ημερησή διάταξη η έκθεση Γκρέσλε για τις έρευνε τη Όλαφ και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Η πρόταση απορρίπτεται. Επομένω, παραμένει ω έχει η διάταξη. Η ομάδα Γκου ζήτησε ω τρίτο σημείο το απόγευμα τη Τρίτη να μπει μια δήλωση τη ΥΠΑ ε, τη εκπροσώπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι Εξωτερικέ Αποθέσει και την Πολιτική Ασφαλεία για την αναγνώριση από την πλευρά των ΗΠΑ των ψηπέδων του Γκολάν ω Ισραηλινού εδάφου και την πιθανή προσάρτηση των επικισμών της ε, Δυτικής Όχθης. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ματίας για να παρουσιάσει το αίτημα της ομάδας Γκουέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε οι δηλώσει του Πρόεδρου των Ηνωμένων ε, το να αναγνωρίσουν τα υψίπεδα του Κολάν ε, ω ε, ε, Ισραηλινό έδαφο. Μονομερή δήλωση, όπω και η δήλωση του Ιταμίνη Τενιάχου πρόσφατα επανεκλέγει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη εδάφη της δυτική Αοχθής είναι δύο προθέσεις που αμφισβητούν την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο διακινδυνεύουν την ειρηνευτική διαδικασία, αλλά παραβιάζουν και το διεθνέ δίκαιο και τι ίδιε τι υφιστάμενε συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισραήλ. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι είναι κατεπήγον να συζητήσουμε και να δούμε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ζητάμε η κυρία Μογκερίνη ως είπατε εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος να κάνει μία δήλωση κατόπιν της συζήτησης για τη Λιβύη για να μπορέσουμε όλοι να συζητήσουμε αυτές τις επαράδεκτες προθέσεις είτε του Πρόεδρου Τραμπ είτε του ε, Πρωθυπουργού του Ισραήλ που πρόσφατα επανεξελέγει. Υπάρχει κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί κατά της πρότασης της ομάδας Γκουε. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία της πρότασης για να προσθεθεί η δήλωση. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Η πρόταση εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν θα μπει ως τρίτο σημείο το απόγευμα της Τρίτης μια δήλωση της Αντιπροέδρου και της Εκπροσώπου για την αναγνώριση από την πλευρά των ύπατων ψηπέδων του Γκολάν ως έδαφων της ΟΗΛ και την πιθανή προσάρτηση των αποκλεισμών της Δυτικής Οχθής. Πάλι την Τρίτη ζήτησε η Γκουέ έχουμε μια δήλωση της ΥΠΑ της Εκπροσώπου για την κατάσταση του Σουδάν Ω τρίτο τέταρτο σημείο το απόγευμα. Τελευταίο σημείο για την είπατε εκπρόσωπο. Τώρα ο κύριο Λόπες έχει το λόγο για να παρουσιάσει το αίτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αλμπασίρ είναι επικεφαλής ενός αυταρχικού καθεστώτος εδώ και 30 χρόνια στο Σουδάν. Ένα καθεστώς που άσκησε διώξεις σε πολιτικού, σε κοινωνικά κινήματα και τα τελευταία χρόνια έχει επιβάλει μέτρα λιτότητα στο λαό της, του Σουδάν. Πρόκειται για μια χώρα στην οποία έχει επιβληθεί κυρώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεργαστεί για μεταναστευτικά θέματα. Του τελευταίου μήνε είδαμε ισχυρή λαϊκή κινητοποίηση που αμφισβητεί την κυβέρνηση ε, είχαμε ένα πραξικόπημα την προηγούμενη Πέμπτη και είχαμε την εκδίωξη του δικτάτορα. Ο λαό του Σουδάν συνεχίζει στο δρόμο να διαδηλώνει και απαιτεί την απόσυρση της στρατιωτικής κυβέρνησης και τη σύγκληση εκλογών. Εμείς ε, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο και πρέπει να συζητηθεί στην Ολομέλεια και γι' αυτό ζητάμε την υποστήριξή σας για να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει κατά του αιτήματο της ομάδας Γκουε. Να περάσουμε λοιπόν, παρακαλώ, ο κύριος Μποστινάρου. Κύριε Πρόεδρε, όταν σχεδιάσαμε να καλέσουμε την ύπατη εκπρόσωπο για μια συζήτηση σε σχέση με το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε δεσμευτεί ότι θα ήταν αποκλειστική συζήτηση για το θέμα αυτό για να δώσουμε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να κάνει μια ουσιαστική συζήτηση με την ύπατη εκπρόσωπο και προκειμένου να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα στο Μελλοντικό Κοινοβούλιο. Τώρα, αν έχουμε και άλλα θέματα που θα τα εισάγουμε εδώ, τότε μπορεί να χάσουμε το στρατηγικό σκόπο της συζήτησής μας. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την προσοχή σας ε, στο όχι, να μην επιβαρύνουμε τη συνάντηση με την υπατή εκπρόσωπο γιατί θα χάσει τη στρατηγική της σημασία. Σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στην ψηφοφορία της ομάδας ΓΚΟΕ, να προσθέσουμε μια δήλωση της ύπατης εκπροσώπου για την κατάσταση στο Σουδάν. Στην ουσία διάταξη ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επομένω, προστίθεται η δήλωση τη Επιτροπή για την κατάσταση του Σουδάν ω τρίτο τέταρτο σημείο το απόγευμα. Η ομάδα των Πρασίνων έχει ζητήσει την προσθήκη ω σημείο στην τρίτη το απόγευμα την πιθανή έκδοση του Τζούλιαν Ασάντς. Έτσι λοιπόν, ε, εκφράσατε τη θέση σα στο παρελθόν, πριν λίγο δηλαδή, θέλετε ω ξεχωριστό σημείο να ξαναθέσετε το θέμα. Εμεί είχαμε ζητήσει να μπει στην μέση διάταξη ως ένα κοινό σημείο, ενώ οι πράσινοι τώρα ζητούν να ξεχωριστά αυτό το θέμα. Να ψηφίσουμε, Χωρί ε, να πάρει κάποιο το λόγο. Ποιο είναι υπέρ. Να προσθεθεί μία συζήτηση μια δήλωση του Συμβουλίου και τη Κομισιόν σε σχέση με την πιθανή έκδοση του Ασάνζ. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπεται νομίζω, αλλά να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Λήξη. Εγκρίνεται η πρόταση. Επομένως, την Τρίτη θα προσθέσουμε τη δήλωση Συμβουλίου και Επιτροπή για την πιθανή έκθεση του Julian Assange. Θα μπει ω τελευταίο σημείο για την Τετάρτη. Η ομάδα των Δημοκρατών ζήτησε να μπει ω πρώτο σημείο το πρωί ε, μια συζήτηση για την έκθεση Μπαλάν για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφαλή. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει η σύνοδο στι 8.30. Να δώσω το λόγο στον, στην κυρία Ροντρίγκε για να παρουσιάσει το αίτημα τη ομάδα τη. Uh, Πρόεδρε, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, θέλω να προτείνω η έκθεση μπάλα να συζητηθεί ως πρώτο σημείο την Τετάρτη, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η ανησυχία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε κοινωνική προστασία σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ε, όταν μετακινούνται στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό είναι ε, κάτι, ένα θέμα στο οποίο έχουμε παραχημένους κανόνες. Η έκθεση μπάλα έχει επικαιροποιήσει σημαντικά τους κανόνες αυτούς. Πρόκειται για πολύ σημαντική πρόοδρο από την ε, πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνολικά είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε ακόμη να φτάσει σε μια ενοποιημένη θέση, αλλά αν ψηφίσουμε και συζητήσουμε το κείμενο αυτό στην πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διασφαλίσει την πρόοδο που σημειώσαμε στον τομέα αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για του Ευρωπαίους πολίτε. Γι' αυτό προτείνουμε το σημείο αυτό να μπει ω πρώτο στην ημερησία διάταξη την Τετάρτη. Υπάρχει κάποιο που θέλει να μιλήσει κατά. Ο κύριος Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, να μην αποδεχτούμε αυτή την ε, αίτηση, αυτό το αίτημα. Σωστά το είπε η προηγούμενη η ομιλητρία, ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό για τους πολίτες στην Ευρώπη, αλλά μετά από μακρές διαπραγματεύσεις δεν καταφέραμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα όπου, για παράδειγμα, να συμφωνεί και το Συμβούλιο. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως στην Επιτροπή μας έχουμε την εξή κατάσταση. Είναι μεγάλο ο διχασμό. Δεν υπάρχει καμία πολιτική ομάδα η οποία θα είναι ικανοποιημένη με την έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το χρόνο που θα έχουμε στην αρχή τη επόμενη θητεία, χωρί πίεση να κοιτάξουμε τα θέματα αυτά τα οποία δεν τα έχουμε ολοκληρώσει με σωστό και εύλογο τρόπο. Είναι σημαντικά θέματα, όχι υποχρονική πίεση να πετύχουμε κάτι βιαστικό. Γιατί θεωρώ ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν συμφωνήσουμε με την πρώτη ανάγνωση θα υπονομεύσουμε τα δικά μας δικαιώματα και θα αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δύσκολε. Δεν θα έχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, την δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε και να προασπίσουμε τα δικαιώματά μας. Την επόμενη θητεία λοιπόν και θα ήθελα να μην δεχτούμε το αίτημα αυτό σήμερα. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω ότι μια εντολή ψηφίστηκε στην Επιτροπή. Η εντολή αυτή επιβεβαιώθηκε εδώ στην Ολομέλεια. Υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο ήταν ενωμένο στη συζήτηση από την αρχή στο τέλος και το Συμβούλιο σήμερα ε, Δυστυχώ δεν μπορεί να εγκρίνει, επειδή υπάρχει μια ψηφία εμπλοκής. Νομίζω ότι για το επόμενο κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ισχυρή θέση με ε, μια ευνοϊκή ε, σχέση ισχύ δυνάμεων ε, και αν κάποια μέλη του Συμβουλίου θέλουν ε, να ξαναθέσουν το θέμα επιτάπητος, παραδείγματος χάρη για τα οικογενειακά επιδόματα, αυτό να μπορεί να γίνει. Δημοκρατικά νομίζω είναι λογικό το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί σε μια πρώτη ανάγνωση, γιατί διαφορετικά θα είχαμε κάνει αυτή την κοινή δουλειά και θα πάει χαμένη και θα είναι κρίμα γιατί ήταν αλληλέγγυο το Κοινοβούλιο. Κυρία Τσίμερ. Θα ήθελα να μιλήσω υπέρ του αιτήματο αυτό να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη, γιατί πρόκειται για μια απόλυτα κανονική διαδικασία. Όταν λαμβάνει η χώρα ένα τριμερή διάλογο και δεν οδηγεί σε συμφωνία, γιατί, για παράδειγμα, το Συμβούλιο δεν συμφωνεί ή δεν σχηματίζει πλειοψηφία, συμφωνούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, σε πρώτη ανάγνωση να ορίσουμε την ε, τοποθέτησή μας από πλευρά του Κοινοβουλίου. Τη θέση την οποία προασπίσαμε και στον τρομερή διάλογο. Ακούσαμε το επιχείρημα ότι δεν είναι όριμη η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου και γι' αυτό δεν μπορούμε να την αποφασίσουμε. Να σας υπενθυμίσω ότι ήταν τόσο όριμη αυτή η τοποθέτησή μας που κάναμε πιο πολλούς από έναν τρεμερή διάλογο και αν εμείς αυτό και λέμε ότι α, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία και ομοφωνία στο Συμβούλιο δεν είμαστε κι εμεί σε θέση να τηρήσουμε τη δική μας αρχική θέση, να σας πω ότι τότε αποτυχάνουμε και να σας υπενθυμίσω και τα δικά σας λόγια, γιατί τα είπατε και προηγουμένω πάρα πολύ εύστοχα κύριε Ταγιάννη. Μιλάμε για το ρόλο, την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν απορρίψουμε το αίτημα αυτό, θεωρώ ότι αποδυναμώνουμε την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την πρώτη Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που έχει ζητήσει να μπει ω πρώτο σημείο, τετάρτο πρέμια συζήτηση για την έκθεση μπάλα. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. η πρόταση. Επομένως, θα ξεκινήσει η σύνοδος στις 8 και μισή το πρωί και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Πέμπτη. Η προθεσμία για τις δροπολογίες Τρίτη, 16 Απριλίου στις 10 το πρωί και τμηματική και ξεχωριστή ψηφοφορία την Τετάρτη 17 Απριλίου στις 4 το απόγευμα. Για την Τετάρτη, η ομάδα FTD έχει ζητήσει δήλωση Συμβουλίου και τη Κομισιόν ε, για μια καθολική ψηφιακή ταυτότητα. Ένα θεμελιώδη δικαίωμα για όλου του Ευρωπαίου πολίτε να μπει ω πρώτο σημείο το πρωί. Η συζήτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί με ψήφισμα που θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Να δώσω το λόγο στον κύριο Καστάλτο για να ξεκινήσει τη θέση τη ομάδα του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προτείνω να μπει στην ημερησία διάταξη μια συζήτηση για ένα θεμελιώδε δικαίωμα για το θέμα τη ψηφιακή ταυτότητα. Το δίκτυο είναι ένα χώρο όπου έχουμε και δημόσια αλλά και ιδιωτική δράση και έτσι έφτασε η στιγμή να θέσουμε συγκεκριμένη προστασία στα δικαιώματα των ανθρώπων όταν ε, στο, όσα συμβαίνουν στο ίντερνετ έχουν επιπτώσει στην πραγματική ζωή. Έτσι λοιπόν ε, όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση με τις ίδιες δικλείδες ασφαλείας. Ε, η ιδιαιτερότητα δικτύου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε την ισότητα και στον εικονικό κόσμο. Θα πρέπει η Ένωση να παρέμβει. Δεν πρόκειται πλέον για ένα θέμα που μπορεί να αναβληθεί. Το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο αποτελεί την προϋπόθεση για να εκμεταλλευτεί κανείς τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο. Όμως ε, κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να προστατεύεται και να είναι αναγνωρίσιμος. Γι' αυτό θέλουμε το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει στο το θέμα του θεμελιώδη δικαιώματο στην ψηφιακή ταυτότητα. Και με αυτό συνδέεται μια σειρά θεμελιωδών όπω ε, η προστασία των προσωπικών δεδομένων που αναγνωρίζεται και από το χάρτη τη νίκαια και το ε, δικαίωμα στη λύθη. Έτσι ζητώ να έχουμε μια συζήτηση με ψήφισμα για την επόμενη Τετάρτη το πρωί σα. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο κατά. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση της ομάδας CFDD να προσθεθεί αυτό το θέμα στην μισή διάταξη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίσκεται η πρόταση. Έτσι λοιπόν, ορίστηκε η μερισία διάταξη. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω το θέμα του, των παιδιών που γεννιούνται ε, από γονείς ε, τρομοκρατών της ISIS και ε, κάποιοι από αυτούς βρισκόνται σε φρικτές συνθήκες, σε φυλακές και θα ήθελα να καλέσω εσάς και τα κράτη-μέλη να αναζητήσουμε λύσεις για τη διάσωση των παιδιών αυτών, για να τα φέρουμε στην Ευρώπη, για να έχουν τη φροντίδα που δικαιούνται ω ε, Ευρωπαίοι πολίτε. Γιατί κανένα παιδί δεν είναι τρομοκράτη, δεν γεννιέται τρομοκράτη και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα πάντα και να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του παιδιού και να πρέπει να εξασφαλίσουμε την τήρηση των χάρτη των δικαιωμάτων των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των δικαιωμάτων του παιδιού. Δεν μπορούν να πληρώνουν τα παιδιά για τα εγκλήματα των γονέων. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στην ημερησία διάταξη. Kellemes délutánt kívánok mindannyiuknak. Ez... Καλησπέρα. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε με την σύνοδο με την έκθεση της κυρίας Ροζιέρ για την προστασία των προσώπων που καταγγέλουν, που παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Έχετε το λόγο κυρία Ροζιέρ. Yes, we noticed it. It's a point of order. The floor is yours. Έχετε το λόγο γιατί διαπιστώσαμε όντως ότι είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και λυπούμε που το θέτω μετά την αναχώρηση του κυρίου Ταγιάννη. Ε, το θέμα έχει να κάνει με την συνεδρίαση του Προεδρείου που θα γίνει σε λίγα λεπτά και θα εξετάσει μια πολύ προβληματική έκθεση για το άρθρο 17. Σχέση μεταξύ των θρησκειών και του Κοινοβουλίου. Και στην έκθεση αυτή η... Ε, συζητείται να διευκολυνθεί το λόμπι των θρησκευτικών οργανώσεων μέσα στο Κοινοβούλιο. Η Μίκιο Open Democracy χρηματοδοτεί με 50 εκατομμύρια ευρώ ε, την πολιτική κατά των δικαιωμάτων ατόμων ε, που είναι λεσβείε ομοφυλόφιλοι και που είναι απαράδεκτο να χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να γίνει μια πλήρης συζήτηση για το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Δεν είναι δυνατόν το θέμα αυτό να συζητείται μόνο σε μια συνεδρίαση του Προεδρείου εν αγνία των βουλευτών και χωρίς να γνωρίζουν οι πολίτες. Ευχαριστώ. Καταγράφουμε το έτοιμά σας και το θέτουμε στα πρακτικά. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Ροζιέρ, πάλι, για την προστασία των ατόμων που καταγγέλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης. Έχετε τέσσερα λεπτά, κυρία Ροζιέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, είναι μια συζήτηση πολύ σημαντική αυτή που κάνουμε για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τον, ρόλο που παίζουν τα άτομα που καταγγέλουν παραβιάσεις της Ένωσης σε μια δημοκρατία. Θέτουμε την δημοκρατία και τη διαφάνεια πάνω από τα συμφέροντα. Προστατεύουμε αυτούς που θέλουν, να, που έχουν το θάρρος να μιλούν και που πρέπει να προστατεύονται. Ο στόχος είναι να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες, τους φορείς που είναι οι πιο προηγμένοι στην προστασία των ατόμων που καταγγέλουν. Το κοινο... Αυτό είναι καρπός μεγάλων συζητήσεων στο Κοινοβούλιο που από το 2014 είχε ξεκινήσει να ασχολείται με το θέμα των καταγγελών των αυτών προτείνοντας εν τέλει μια οδηγία. Έκτοτε έχουν αυξηθεί τα σκάνδαλα, Panama Reports, Wikileaks, Football Leaks, δείχνουν πόσο ευάλωτη είναι η κατάσταση των καταγγελόντων αυτών. Έφτασε τώρα η οδηγία δημιουργώντας πολλές ανησυχίες που θέλουμε να διορθώσουμε με την τωρινή οδηγία, αλλά θέλουμε να θέσουμε την οδηγία αυτή υπό την αίρεση μιας πραγματικής προστασίας των ατόμων αυτών. Η συζήτηση στο ημικύκλιο αυτό όταν είχε γίνει, Μα είχαν εξηγήσει από την Επιτροπή ότι δεν ήταν επαρκέ, ότι δεν υπήρχε νομική βάση στην Ένωση για να μπορέσει να αναλάβει δράση η Ένωση. Ωστόσο, τρία χρόνια μετά, σήμερα, συζητούμε το θέμα και αύριο, ελπίζω, θα εγκρίνουμε μια οδηγία που θα προστατεύσει του καταγγέλλοντε σε όλη την Ένωση. Η δέσμευση των συναδέλφων αλλά και τη κοινωνία των πολιτών, των ΜΚΟ που θέλω να καλωσορίσω εδώ, έδωσαν αποτελέσματα. Μετακίνησαν τις θέσεις και κατεύθυνε την Ευρώπη προς ένα δρόμο που δείχνει ότι ακούει τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλω και εγώ να το υπογραμμίσω ότι αν και σπάνιο συγχαίρω την Επιτροπή, την κυρία Γιούροβα και για τη δουλειά που έκανε και για την, ε, τις προσπάθειες που, που κατέβαλε για να βρει λύσεις, να μειώσει τις, ε, τα ερωτηματικά για το θέμα των καταγγελόντων. Έτσι μπορούμε με ένα κείμενο αυτό να προσφέρουμε μια εκτεταμένη προστασία στους ανθρώπους αυτούς, όπως είχαμε ζητήσει στην, ε, στο ψήφισμα που είχαμε υποστηρίξει το 2010. Καλύπτονται και οι μισθωτοί και οι ασκούμενοι και οι συμβασιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θέλησαμε να μην αφήσουμε κενό στην προστασία που θέτουμε και θεσπίζουμε αύριο. Θα θέλαμε επίσης να ε, βοηθήσουμε και άτομα που διευκολύνουν ή βοηθούν τους καταγγέλλοντες και που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπλέκονται από πιθανότητες αντιπίνων. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί στις διαπραγματεύσεις διαφυλάξαμε την αρχική φιλοδοξία του κειμένου της Επιτροπής με εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής ενώ η προστασία των, και στην προστασία των συμφερόντων της Ένωσης, φορολογικά ζητήματα και προστασία του περιβάλλοντος. Και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα ακολουθήσουν τις συστάσεις μας πηγαίνοντας πιο πέρα και από τις ε, τομεακές ε, δυνατότητες εφαρμογής οδηγίες. Ο μηχανισμός ε, σήμανσης που έχουμε υιοθετήσει είναι ένα βασικό κλειδί που υλοποιείται από την υποχρέωση δικτύων ενημέρωσης. Θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι δεν, μάλλον να, διαφωνήσω με ένα από βασικό πρόβλημα, την εσωτερική πληροφόρηση. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα του, του αρχικού κειμένου. Εμείς σαν Κοινοβούλιο βελτιώσαμε το κείμενο, καταργήσαμε την υποχρέωση αυτή που θα ε, οδηγούσε σε σίγουρες κυρώσεις και αντίπεινα κατά, του καταγγέλλοντος. Προτείνουμε ουσιαστική προστασία κατά αντιπίνων, ε, ασυλία για την απόκτηση πληροφοριών που έχουν αποκαλυφθεί και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουν τα κράτη-μέλη αλλά πρέπει να το πετύχουμε. Ε, αντιστροφή του βάρους ε, ε αποδείξεως που προστατεύει τους τους, ψυχολογική και χρηματοοικονομική υποστήριξη. Αυτό το ενισχύουμε για να μην είναι μόνοι τους οι άνθρωποι αυτοί που συχνά αισθάνονται απομονωμένοι ενώπιον των τεράστιων ε, πολυεθνικών. Το φιλόδοξο κείμενο που θα υιοθετήσουμε ενισχύει την δημοκρατία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους και ηγητές που έδειξαν ότι όταν το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο μπορεί να κερδίσει, να δώσει αποτελέσματα και να αντιστρέψει και τις παρελκύουσες μειοψηφίες στο Συμβούλιο, κάτι σπάνιο. Πρέπει να ευχαριστήσω εκ νέου την Επίτροπο γιατί έδειξε ότι πραγματικά ήθελε να πετύχει μια συμβαστική καλή λύση. Ελπίζω αυτό που θα ψηφίσουμε αύριο θα είναι ένα καλό και θετικό αποτέλεσμα για την Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει κ. Βιέκας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Και θα το επαναλάβω. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ είναι το ποσό απάτης και φοροδιαφυγής και ισοδυναμεί έξι φορές τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλές φορές ε, ε, στον προπολογισμό για την παιδεία και την υγεία της Πορτογαλίας και ε, φυσικά χάρη στους καταγγέλλοντες γλιτώνουμε αυτά τα ποσά καταγγέλλοντες σήμερα ε, όπως ε, βλέπουμε και από την περίπτωση Σάνση και την περίπτωση μαζιογράφου στη Μάλτα, ποινικοποιούνται. Είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Πρέπει να εγγυόμαστε την απόλυτη ανωνυμότητα των καταγγελόντων και την πλήρη προστασία τους. Γιατί στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα οι καταγγέλλοντες είναι οι μόνοι που καταδικάζονταν. Και αυτό αποκαλύπτει το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και ε, φυσικά τελικά οι παλιοεθνικές συνεχίζουν με το να παραμένουν ατιμόρυτες. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η οδηγία και είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εκ μέρους ε, της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ, η κυρία Ρουίς έχει το λόγο. Εγώ ήμουν αρμόδια για την εκπόνηση της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ παρά ε, γιατί πρόκειται μόνο για μια γνωμοδότηση, Σκιώτης ε, και εγώ. Κάναμε μια συνολική δουλειά. Ασχοληθήκαμε με το να πάει παραπέρα όλη η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων μας υποστήριξε για να έχουμε μία θέση του νομιλού σύμφωνα με το αίτημα της κοινωνίας. είχαμε να αυξήσουμε την ασφάλεια δικαίου και να μειώσουμε τον κατακαιρματισμό τη προστασία των καταγγελόντων. Σήμερα οι καταγγέλλοντε πολλές ε, φορές ε, δεν μιλούν επειδή φοβούνται τα αντίπεινα. Όμω με την οδηγία αυτή ελπίζουμε ε, να προστατεύονται μέσω ασφαλών διάβλων για την καταγγελία. Επίση προστατεύουμε τις πηγές της ερευνητική δημοσιογραφίας και το αστικό καθήκον της καταγγελία για να μην πρόκειται για μια ηρωική πράξη. Και προσθέτουμε ένα ακόμα στρώμα δικλειδών ασφαλεία για ε, το δημόσιο συμφέρον, ε, γιατί δεν θα ήταν δυνατό να εργαστεί η Επιτροπή Πάνα ε, δίχως τις αποκαλύψεις των Panama Paper και τελικά μπορέσαμε να διφυλάξουμε την ανωνυμία των καταγγελόντων. Μιλάμε για πολύ μεγάλα εγκλήματα που αποδυναμώνουν τις δημοκρατίες μας αλλά και τα δημόσια ταμεία. Γι' αυτό ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε το γενικό συμφέρον και με αυτή την οδηγία όλοι κερδίσουμε. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο έχει η κυρία Γιουροβά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ. Να ευχαριστήσω την ε, κυρία Ροζιέρ, την εισηγητρία, του κοιόδου εισηγητέ και ε, της Προεδρία τη Ευρωπαϊκή ε, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας επέτρεψαν γρήγορη εφαρμογή και συμφωνία σε ό,τι αφορά το σημαντικό αυτό θέμα. Και συμφωνώ με την κυρία εισηγητρία ότι οι διαπραγματεύσει δεν ήταν απλέ και εύκολε. Ωστόσο, όλοι ξέραμε ότι είχαμε στα χέρια μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η συμφωνία η οποία επιτεύχθη είναι ένας ε, σεμιβασμός καλά εσυρεπομένος σε ό,τι αφορά την προστασία των ε, καταγγελόντων και την ενίσχυση της ε, εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Τα πρόσφατα σκάνδαλα όπως το Dieselgate, το LuxLeaks, τα Panama Papers και τη Cambridge Analytica δεν θα είχαν έρθει στο φως αν δεν υπήρχε το θάρρος των καταγγελόντων αυτών. προστατεύοντα λοιπόν τους whistleblowers μπορούμε να ε, αποτρέψουμε την ε, βλάβη ε, του συμφέροντων του κοινού σε ό,τι αφορά την διαφθορά, την απάτη, αθέμητες πρακτικές, αμέλειες κτλ. Και αυτές οι, τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας που υπάρχουν θεωρώ ότι έχουν να κάνουν και ε, την προσωπική σωματική υγεία αλλά και τα συμφέροντά τους. Οι καταγγέλλοντας λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουν πού μπορούν να προστατευτούν ε, στην ε, επιχείρηση που δουλεύουν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στον δημόσιο και δυτικό τομέα, στις επιχειρήσεις, στις εταιρείε που χρειάζεται να προστατεύουν τους καταγγέλλοντες. Ωστόσο, ξέρουμε ότι είναι σημαντικό θέμα αυτό για το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπάρχει και το θέμα της ελεύθερης βούλησης να καταγγέλει κανείς τα περιστατικά αυτά άμεσα στην ανώτατη αρχή αν το θεωρέσουν αυτό απαραίτητο και θα χαίρουν πλήρη ε, προστασία όταν αποφασίσουν να κάνουν τέτοια κίνηση. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ενίσχυση σε βασικούς ε, τομείς ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών. Έτσι αυτό θα υλοποιήσει την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει τέτοια ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, όπως καταγγέλει και η ανακοίνωση του 2016 για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο καλύτερα αποτελέσματα μέσω καλύτερη υλοποίηση. Και μια και πρόκειται για μια οδηγία με κοινά ελάχιστα πρότυπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κλάτη μελη να επεκτείνουν αυτή την οδηγία και σε άλλους τομείς και να δημιουργήσουν ένα συνεχτικό πλαίσιο για την προστασία των ατόμων και των πολιτών. Αυτό πλέον αποτυπώνεται ρητά στο κείμενο. Και ως τμήμα του συμβιβασμού σε ό,τι αφορά το υλικό σκέλος προβλέπουμε αναθεώρηση της ε, οδηγίας το συντομότερο δυνατόν, το 2025 ήτι, τέσσερα χρόνια μετά από την εφαρμογή της οδηγίας. Και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εκτιμηθούν ε, συγκεκριμένα τα θέμα της συμπερίληψης του τομέα της κοινωνικής πολιτικής στην ε, στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Και αυτό θα επιτρέψει μία σε βάθος ανάλυση του πώς θα επηρεάσει η οδηγία το εφιστάμενο κοινωνικό και Και έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει η πολιτική δήλωση αυτή να προσαρτηθεί στην την ε, οδηγία. Παράθεση. Τότε όταν ε, βάσει του άρθρου 27 της οδηγίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα επέκταση του πεδίου εφαρμογή συμπερίληψη ε, κάποιων πράξεων βάσει του 153 και 157 άρθρου της συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικού εταίρους όπου αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με το άρθρο 154 τέλος παράθεσης. Και για να κλείσουμε, συμφωνώντα επί των προτύπων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύει τη δέσμευσή τη στην ε, διαφάνεια, λογοδοσία, καλή διακυβέρνηση και ελευθερία έκφραση, δικαιώματα αναπαρατρίωτα, επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αποτελεί ένα σαφέ και ξεκάθαρο μήνυμα προ του πολίτε, προ του εμπλεκόμενου φορεί, εν ώψη των ευρωεκλογών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει λοιπόν απόλυτα το συμβιβασμό που εξευρέθη μεταξύ των συνομοθετών και προσβλέπει στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρο. Και τώρα το λόγο έχει η κ. Φλάνναγκαν για ένα λεπτό από την Επιτροπή Ελέγχου Προεπλογισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι καταγγέλλοντες, οι whistleblowers είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, πολύ θαραλέοι, οι οποίοι πραγματικά α, παίρνουν μεγάλο ρίσκο. Και αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα ελπίζουμε ότι θα σημαίνει στο μέλλον ότι δεν θα σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι κανείς ε, πάρα πολύ θαραλέος, ε, ασυνήθιστα θαραλέος, για να μπορέσει να κάνει τέτοιες καταγγελίες. Γιατί στην παρόσα φάση στη χώρα μου αν ε, κάποιο κάνει κάποια τέτοια καταγγελία, καλά θα κάνει να φοβάται, γιατί θα τον θα τον βασανίσουν πνευματικά, ψυχολογικά, θα τον καταστρέψουν οικονομικά. Και έτσι θα πρέπει να πετύχουμε να έχει ο κόσμος, όλοι μας δηλαδή, μηδενικό ποσοστό φόβου όταν κάνουν τέτοιες καταγγελίες. Να μην φοβούνται να αναπνεύσουν, να ζήσουν, να κινηθούν. Νομίζω λοιπόν ότι πετύχαμε κάτι καλό εδώ σήμερα. Δεν ε, συμβαίνει πολύ συχνά αυτό και γι' αυτό και το επικροτώ, το χειροκροτώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα, από την Επιτροπή Απασχόλησης, έχουμε τον κύριο Λέι Ιαρίκ για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, επειδή η οδηγία για την τήρηση του απορρίτου ε, δεν αρκεί. Πρέπει να ενισχύσουμε το κείμενο, όπως μας προτείνει δικαίως η κυρία Ροζιέμπρο και για το γενικό συμφέρον έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε συνολική προστασία και ω δυνατόν ευρύτερο πεδίο εφαρμογή ε, και να μην έχουμε πάρα πολύ περιορισμένε εξαιρέσει. Τα κράτη θα έχουν λοιπόν μεγάλο περιθώριο ε, στην εφαρμογή αυτή τη οδηγία, ε, και αυτό μπορεί να μα ανησυχήσει αν σκεφτούμε ότι κάποιε κυβερνήσει προσπαθούν να μπλοκάρουν την νομοθεσία. η Επιτροπή θα πρέπει να επαγρυπνεί προκειμένου να υπάρξει μια καλή και ορθή εφαρμογή της προστασίας που δημιουργούμε. Παραδείγματος χάρη ε, να υπάρξουν και κατευθυντηρίες γραμμές στις οποίες αναφερθήκατε, Επίτροπε, ή να υπάρχει μια ε, ανακοίνωση ερμηνευτική έτσι ώστε όλοι να χαίρουν της μέγιστης προστασίας όταν ε, θέλουν να καταγγείλουν ε, ε, κάποιες πρακτικές που θίγουν το δημόσιο συμφέρον. Νομίζω ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προποθέσει για να προστατεύσουμε και τον Τζούλιαν Ασάντς, στον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί το δίκαιο για τους δημοσιογράφους όπως ρυθμίζεται από τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. ο ομιλητή από την Επιτροπή Ένβη είναι ο κ. Ζωμαρζή. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, λέτε ότι θέλετε να προστατεύσετε τους ε, καταγγέλλοντες. Τι συμβαίνει όμως με τον Τζούλιαν ε, Assange. Η τιμή για τους Ευρωπαίους ήταν να γνωρίσουμε την ε, οφειλή που έχουμε απέναντί του. Γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο Ασάντζ αποκάλυψε μαζική κατασκοπία από τις ΗΠΑ των ευρωπαϊκών χωρών, συμμάχων των ΗΠΑ. Η υποχρέωσή μας σήμερα είναι να του χορηγήσουμε άσυλο. Όπως γνωρίζετε, κινδυνεύει να εκδοθεί. Μέσω αυτού όλοι οι καταγγέλλοντες ε, που θέλουμε να προστατεύσουμε τον κορονισμό τρομοκρατούνται. Ήρθε η ώρα να αλλάξει ο φόβος στρατόπεδο και να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά διώκονται, παρενοχλούνται, δικάζονται και μερικές φορές δολοφονούνται. Αλλά πρέπει να δείξουμε ότι τιμάμε τις υπηρεσίες που, δίνουμε, που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι ξεκινώντας από τον Τζούλιαν Ασάν σήμερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χουντής για την Επιτροπή Πολιτισμού. Ένα λεπτό αγαπητοί συνάδελφοι η σύλληψη του τζούλιαν ασάντζ είναι μια εικόνα από το μέλλον μας ένα μέλλον ανελευθερίας και καταστολής όπου οποιαδήποτε αποκάλυψη της βαρβαρότητας και των παρανομιών του νεοφιλελεύθερου ολοκληρωτισμού θεωρείται έγκλημα της κυβέρνησης του δυτικού κόσμου. η σύλληψη ασάντζ από τη βρετανική κυβέρνηση κατ' εντολή των ηνωμένων πολιτειών έγινε γιατί μέσω της ιστοσελίδας wikileaks αποκαλύφθηκε η βαρβαρότητα των επεμβάσεων των ηνωμένων πολιτειών και των συμμάχων της στη μέση ανατολή και αλλού και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνού δικαίου. με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουν οι υπεριαλιστικέ δυνάμει την ελευθερία τη έκφραση τη μαχόμενη δημοσιογραφία που αποκαλύπτει τι πιο σκοτεινέ τη πλευρέ προ όφελο τη δημοκρατία τη διαφάνεια και τη αλήθεια. η σύλληψη αζάν μα αφορά όλου. οφείλουμε να προστατεύσουμε όσου ξεμπροστιάζουν την πολιτική και οικονομική εξουσία αν θέλουμε ένα διαφορετικό μέλλον για την ευρώπη ένα διαφορετικό μέλλον για τον κόσμο μας οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με το κίνημα υπεράσπισης των ελευθεριών της έκφρασης και της ενημέρωσης. ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά προς όφελος της διαφάνειας, της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος και του δικαίου της Ένωσης. Θα έλεγα ότι κάνουμε και ένα μεγάλο βήμα μπροστά στην δεοντολογία, στην δημόσια δράση. Θέλω να συγχαρώ την Βιζινή Ροζιέρ που έκανε εξαιρετική δουλειά και την Επίτροπο ταυτόχρονα. Να σας πω κυρίες και κύριοι ότι οι καταγγέλλοντες δεν είναι εγκληματίες. Είναι υποδειγματικοί πολίτες θα έλεγα. Δυστυχώς πολλές, πολλά παραδείγματα έχουμε όπου α, τέτοια άτομα υπέστησαν βίαιη αντιμετώπιση. Έχασαν τη δουλειά τους, τη σταδιοδρομία τους, διώχθηκαν μέχρι την οικονομική καταστροφή τους και κυνηγήθηκαν και ποινικά από κάποιες χώρες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να σταματήσει και ευτυχώς η οδηγία που είναι καλή, που είναι πληρέστατη όπως ήδη αναφέρθηκε, που ευνοεί όπως ξεκαθαρίστηκε από τις απόψεις όλες των πολιτικών ομάδων, αποτελεί υποχρέωση των κυβερνήσεων να ενσωματώσουν την οδηγία στο εθνικό του δίκαιο και γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα να ακούσουμε από τις πολιτικές ομάδες ε, τους εκπροσώπους από το ΕΛΚ. Ο κύριος Άξελ Φως έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρα. Ευχαριστώ και την Επιτροπό για τις ε, δηλώσεις σας. Είναι κρίμα το γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται υπό μεγάλη χρονική πίεση στο τέλος της θετίας μας και εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να αφιερώσουμε πιο πολύ χρόνο επί της αρχής σε τέτοια θέματα και να ευχαριστήσουμε και ε, τους ε, σκιώδεις εισηγητές, ε, την εισηγήτρια η οποία πραγματικά έχει σε υδρότα και αίμα για το θέμα αυτό. Εισαγωγικά λοιπόν μιλήσαμε για τις νόμιμες καταγγελίες και νομίζω ότι είναι πραγματικά η στιγμή. Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να υπάρχουν τέτοιες διατάξεις και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται και στο συμβιβασμό που επιτρέφθη σε ό,τι αφορά δηλαδή, την τήρηση του δικαίου και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι νόμιμο, τι είναι με παράτυπο, να μην υπάρχουν ηθικές δεντολογικές κρίσεις και συζητήσεις από αυτόν κάθε φορά. Θα πρέπει να συμφωνούμε σε ό,τι αφορά το δίκαιο ως βάση. Και πιστεύω ότι είναι σωστό το γεγονός αυτό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θεωρώ ότι βρήκαν μια τέτοια βάση γιατί το κόστος εφαρμογής είναι πάρα πολύ υψηλός και με τον τρόπο λοιπόν αυτό μπορούμε να το μειώσουμε και να υπάρχει κάποια συντονισμός μέσα των ενώσεων και των συλλογικών οργανώσεων για να βρεθεί ένα μοντέλο για το οποίο δεν χρειάζεται να πάει κανείς κατευθείαν σε στα, μέσα ενημέρωση ίσω να υπάρχουν εσωτερικέ και εξωτερικέ δυνατότητε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι όλου όσου συμμετείχαν στην διαδικασία αυτή. Από πλευρά του ΕΛΚ θεωρώ ότι μπορούμε να την υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή χωρί πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Κάουφμαν είναι η επόμενη. Για δύο λεπτά. Από του Σοσιαλιστέ και δημοκρατές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα αυτή για μένα. 28 χρόνια μετά την πρώτη συμμετοχή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως παρατρίτρια από την Βυτική Γερμανία. Σήμερα έχω την ε, τιμή για τελευταία φορά να μιλώ στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία και να ευχαριστήσω ιδιαίτερως όλους εσάς. Η συνεργασία μαζί σας αγαπητοί συνάδελφοι πάντα μου έδωσε μεγάλη ικανοποίηση για την κοινή μας αυτή η Ευρώπη. Το κοινοβούλιο αυτό με μέλη από πολλές διαφορετικές χώρες πραγματικά είναι κάτι μοναδικό. Και πραγματικά έχουμε πετύχει πάρα πολλά από κοινού. Αυτό λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας αποτρέψει να συνεχίσουμε τις μάχες και τους αγώνες για το έργο αυτό. Σε καμία περίπτωση λαϊκιστές και εξτρεμιστές δεν θα πρέπει να αφήσουμε να καταστρέψουν ή να αποτιμήσουν αυτό το κοινό έργο μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο θα δώσουμε το πράσινο φως για μια ευρωπαϊκή, πανευρωπαϊκή προστασία των καταγγελόντων. Πανευρωπαϊκή προστασία για τους ανθρώπους οι οποίοι ε, αποκαλύπτουν παρατυπίες προς το κοινό συμφέρον. Μεγάλη πρόοδος, λοιπόν, μεγάλη επιτυχία για τους πολίτες και για μας ως ευρωβουλευτές. Αυτή την προστασία τη ζητούσαμε εδώ και καιρό. Και αγωνιστήκαμε για τον σκοπό αυτό. Και πλέον στέφονται με επιτυχία αυτοί οι αγώνες. Και πιστεύω ότι πολλοί συνέδελφοι οι οποίοι εκ νέου θα κατέβουν στις εκλογές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και το παράδειγμα αυτό της προστασίας των καταγγελόντων αλλά και πολλά άλλα επιτυχημένα παραδείγματα για να τα μεταβιβάσουν προς τους πολίτες και να τα συνδέσουν με το εξής μήνυμα ότι το ευρωπαϊκό έργο αποτελεί υπεραξία για όλους τους πολίτες. Είμαι περήφανη και ευτυχή που είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτό. Ευχαριστώ. Η πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Τόμασιτς έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό που συζητούμε την πρόταση αυτή για την προστασία των μαρτυρών δημοσίου συμφέροντος ακριβώς αυτές τις μέρες ε, ε, οπότε βιώνουμε και τη σύλληψη του Ασάνς και ε, επίσης είμαι πολύ ικανοποιημένη που έχουμε ενώπιόν μας μια πολύ ισορροπημένη έκθεση που θα αυξήσει την προστασία όλων των ατόμων που αποκαλύπτουν πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος Όμω προκειμένου να λειτουργήσει καλά αυτή η προστασία χρειαζόμαστε τις κατάλληλε προποθέσει και στην κοινωνία να εκτιμάται δηλαδή ο αλτρουισμός των καταγγελόντων ε, και οι θεσμοί να ε, λειτουργούν με ένα επαγγελματικό τρόπο για τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Τις πληροφορίες ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες γιατί αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε χειραγώγηση του κοινού. Αλλά θα πρέπει να είναι αντικείμενο περαιτέρω επαγγελματική έρευνα και αποκάλυψη τη αλήθεια. Η δεύτερη απαραίτητη προπόθεση είναι η αποτελεσματικότητα των δικαστικών και διοκτικών αρχών ένα άλλο καυτό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στις χώρες το συντομότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για δύο λεπτά ο κύριος ε, Καβαντά εκ μέρους του Άλντε. Ευχαριστώ. Αν ε, ε, στραφούμε στο να δούμε τι έγινε σε αυτή τη θητεία, θα δούμε ότι έφερε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαίους πολίτες και ε, μάλιστα έδωσε και στους Αμερικάνους βουλευτές ε, την ιδέα να εμπνευστούν από το δικό μας έργο προκειμένου να μην ε, είναι ε, οι πολίτες ε, αντικείμενο εκμετάλλευση από τις ΓΚΑΦΑ. Αν δούμε το έργο αυτής της θητείας των πέντε ετών που πέρασαν, θα αντιληφθούμε σήμερα ότι έγινε μια πολύ μεγάλη δουλειά θεμελιώδης. Αν ο κύριος Σνόντεν ήταν Ευρωπαίος, δεν ε, θα είχε εξοριστεί ε, σε ε, μια μικρή μοσχοβετική γωνιά με να τον παρακολουθούν όλες οι υπηρεσίες να είναι γύρω του διάφοροι κατάσκοποι που θα ήθελαν να εκδοθεί στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έτσι λοιπόν, όταν, ε, μιλά, όταν σας μιλήσουν για την Ευρώπη, συνάδελφοι, να πείτε ότι δεν πρόκειται μόνο για μια αξιόλογη οικονομική εντότητα, αλλά για μια οντότητα που έχει κατορθώσει να προστατεύσει περισσότερο από άλλες οντότητες στον κόσμο τη συλλογική και ατομική ελευθερία. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ροζιέρ, την συγγήτρια, η οποία εξαιρετικά εργάστηκε και την κυρία Γιούροβα ε, για το κείμενο της Κομισιόν ε, πολλές φορές ε, λέμε πολλά κακά για την Κομισιόν, όμως ήταν ουσιαστικό αυτό το κείμενο. Και ε, η δουλειά που κάνετε ε, ουσιαστικά θα βοηθήσει όλους τους καταγγέλλοντες στην Ένωση και τελικά δεν θα υπάρχουν σύνορα στην προστασία. Σας ευχαριστούμε για το έργο αυτό για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ. Πασκάλ για τους πράσινους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια Ευρώπη που προστατεύει το γενικό συμφέρον τους πολίτες της Ένωσης συνολικά είναι κάτι που είναι δυνατό. Δεν χρειάζεται να παρεκβούμε τις ε, συνθήκες ή να περιοριστούμε στα σύνορά μας. Αντίθετα, η Ευρώπη υπάρχει. Αυτή η Ευρώπη είναι σε μία στιγμή που η δημοκρατία κινδυνεύει από την αδιαφάνεια και, τους, ε, και την τεχνοκρατία, χρειάζεται τους ε, πληροφοριοδότες, χρειάζεται τους πολίτες που ξεσηκώνονται και καταγγέλουν αυτά που κάποιοι θέλουν να κλείσουν, να κρύψουν. Αυτό κάνουμε σήμερα. Αυτό κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χάρη στην Επιτροπή. Ευχαριστούμε την κυρία Γιούροβα, τον κύριο Τίμερμαν που θέλησαν να το υιοθετήσουν. Ευχαριστώ τη Βιζινή Ροζιέλ και όλου όσοι δούλεψαν για το ζήτημα αυτό. Να πω ωστόσο κάτι πέραν τη σημασία του κειμένου. Το γεγονός ότι όταν το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο, όταν πραγματικά το Κοινοβούλιο θέλει να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον, δεν το σταματάει τίποτα. Ούτε η συντήρηση, ούτε τα λόμπι και επιτρέπουμε να προχωρήσει η δημοκρατία και το δίκαιο. Ο κύριος Καστάλντο για τους EFTD. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επιτέλους καταφέραμε να εγκρίνουμε μια οδηγία που όλη η Ευρώπη ανέμενε εδώ και χρόνια. Εκτιμάται ότι οι πόροι που έχασε το, η εφορία και η, η έλλειψη επενδύσεων έχουμε χάσει στην Ευρώπη 90 δισεκατομμύρια το χρόνο σε ΑΕΠ και παρά τα αυτά ακόμα και σήμερα δεν υπήρχε ειδική ρύθμιση για την προστασία των καταγγελόντων που είναι μπροστά στη μάχη αυτή. Μεταξύ αυτών είναι οι καλύτεροι πολίτες της Ένωσης, οι καλύτεροι δημοσιογράφοι που προχωρούν τις έρευνες ακριβώς ε, όταν ε, προσπαθούν να ανακατέψουν την κατάσταση για να βγάλουν την, να την αλήθεια. Η στάση μας όμως ε, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους είμαστε οφειλέτες. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε στο περιθώριο της κοινωνίας. Πρέπει να προστατευθούν διότι δεν μπορεί να συμβεί σε αυτούς αυτό που συνέβη στην Τάφνη Καρουάνα πρόπερση, στον Γιακούσνα πέρυσι πρέπει να παράσχουμε προστασία και από τις, τα αντίπεινα και για τον πληροφοριοδότη και για την οικογένειά του, αφήνοντας τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν με καλύτερες και πιο προηγμένες ρυθμίσεις, άμα θέλουν. Είναι παράδοξο, συνάδελφο, την παραμονή της έγκρισης οδηγίας αυτής, και θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό αύριο, να, να συλλαμβάνεται ο Τζούλιαν Ασάν στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ε, αποκάλυψε εξαιρετικές ε, συνδέσεις και πληροφορίες που ουδέποτε θα είχαμε. Ο Ασάνς δεν μπορεί να εκδοθεί, δεν πρέπει να εκδοθεί στη ΣΥΠΑ όπου κινδυνεύει με τη θανατική ε, ποινή. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο όχι. Για το ΕΛΚ, Ζάμιτ Ντίμεχ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι όταν ψηφίσουμε αύριο την αυτή νομοθεσία θα είναι πραγματικά πολύ κατάλληλη ημέρα. Αύριο, βλέπετε, θα έχουμε 18 μήνες, έχουν κλείσει 18 μήνες από την ε, ε, βία δολοφονία της Δάφνης Κορυβάνα Καλίτσια, της ε, δημοσιογράφου αυτή. και πραγματικά στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διαπιστώσουμε τη σημασία της νομοθεσίας αυτής. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο στέλνει ένα σαφές μήνυμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να προστατευτούν οι ερευνητέ ε, δημοσιογράφοι και ήταν τιμή μου από κοινού με τους συναδέλφους να εργαστώ για την ε, κατάρτιση της νομοθεσίας αυτής στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και σε διάφορα θέματα πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω ότι δούλεψα όχι μόνο γιατί η νομοθεσία αυτή παρέχει μεγαλύτερη προστασία σε αυτούς που καταγγέλουν και τους δημοσιογράφους, αλλά γιατί ουσιαστικά αποτελεί και μια δικλίδα ασφαλείας για τα συμφέροντα των πολιτών. Γιατί χάρη στους κατακέλλοντες, χάρη στους δημοσιογράφους αυτούς. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες τις οποίες έχουν δικαίωμα να έχουν. Τα κράτη-μέλη λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα γίνει σωστή εφαρμογή της οδηγίας αυτής ε, για να υπάρχει σωστή προστασία των καταγγελόντων και βάσει των όσων ε, α, προβλέπει ο νόμος, όχι βάσει του κατά πόσον αρέσει αυτό στην εκάστοτε κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες για τους πολίτες πληροφορίες που δεν θα είχε πρόσβαση αλλιώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κ. Κοφεράτη έχει το λόγο για ένα λεπτό από τους Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, όπως είναι γνωστό, η διαφάνεια στην πολιτική και δυναμική αλλά και στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα είναι κάτι θεμελιώδες για να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον. Να κάνουμε ένα βήμα προς το στην κατεύθυνση, πολύ σημαντικό, ήταν ευαίσθητο το ζήτημα. Αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε τους θεραλέους ανθρώπους, αυτούς τους καταγγέλλοντες που έχουν αποκαλύψει κατά τη διάρκεια αυτών των ε, τελευταίων ετών και μηνών πολύ αρνητικά ζητήματα όπως το Panama Paper, το LuxLeaks, το Paradise Papers με την αντίθεση να εργάζονται αυτοί για το, για το γενικό συμφέρον ε, ενώ κανείς δεν τους υπερασπίζει. Για πρώτη φορά εμείς ε, δημιουργούμε ένα δίκτυο προστασίας πολύ σημαντικό για να ε, δώσουμε και κίνητρα στο να εκδηλωθούν τέτοιες συμπεριφορές. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε εσά την συγγήτρια και όλους όσους εργάστηκαν με πεποίθηση εσείς θα έχετε και ένα σημαντικό ρόλο στη συνέχεια να διαδραματίσετε, γιατί εγώ πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να επαγρυπνεί για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής, γιατί τα κράτη που την αντίθετα δεν θα χάσουν την ευκαιρία για να προσπαθήσουν να αμφισβητήσουν αυτά που θα έχουμε ψηφίσει. Σας ευχαριστούμε για τα όσα κάνατε και ελπίζω να μας δώσετε και συγκεκριμένη βοήθεια για την ορθή εφαρμογή. Η κυρία Ρέντα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχεδόν πριν από τρία χρόνια η ομάδα των Πρασίνων παρουσίασε ένα σχέδιο οδηγία για την προστασία των καταγγελόντων. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα συντονισμένη προσπάθεια τη κοινωνία των πολιτών, πολιτικών και δημοσιογράφων και ήταν αντίδραση στην οδηγία για τα εμπορικά μυστικά που είχε ε, υιοθετηθεί και απειλούσε του καταγγέλλοντε από τότε το σχέδιο κειμένου μας έδειχνε ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταγγελόντων είναι πιθανή και συνέπεσε με το σκάνδαλο LuxLeaks. Θέλαμε να δυσφυλίσουμε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθεί το εμπορικό απόρριτο κατά των καταγγελόντων, όπως ήταν και η περίπτωση με το LuxLeaks. Το 2015 δόθηκε το βραβείο των Ευρωπαϊκών Πολιτών, αλλά ε, κατόπιν ε, τον, ο, κατηγορήθηκε ε, ο άνθρωπος αυτός ψευδός και ε, Τώρα, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ε, ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση το σχέδιο της οδηγίας που θέλαμε να υιοθετήσουμε Ακριβώ αναφέρει αυτό που ζητήσαμε το 2016, προστασία των καταγγελώτων να υπερισχύει του εμπερικού απορρίτου. Με αυτή την ε, οδηγία θα μπορέσουν οι καταγγέλλοντε να βασίζονται σε προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Επίτροπο και όλους τους συναδέλφου που εργάστηκαν για το θέμα αυτό. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ κύριο Σβόμποτα για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μια κοινότητα δικαίου και άρα πρέπει να προστατεύει την δική της νομοθεσία. Η έκθεση αυτή είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι σύνθετες κοινωνίες του 21ου αιώνα σέβονται το δίκαιο. Προστατεύουμε αυτούς που προστατεύουν το το δημόσιο συμφέρον και μας πληροφορούν για τις παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Είναι σαφές ότι η κοινωνία δεν μπορεί να αγνοήσει τα σύγχρονα μέσα προστασίας. Ο ρόλος των πληροφοριοδοτών είναι ουσιαστικό σε κάποιες περιπτώσεις για να μπορούν να ανοιχνεύσουν τις σοβαρές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου πρέπει, η προστασία είναι μια ισορροπημένη προστασία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε μια αναλογική προστασία και σε περιπτώσεις συλλογικών δράσεων. Ο στόχος δεν είναι να μετατρέψουμε την κατάσταση αυτή σε μια μάχη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Είναι ωστόσο δυνατό και το είδαμε αυτό στις διαπραγματεύσεις ότι η συμβαστική, που πετύχαμε είναι θετική και τους υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ. Η εξουσία χρειάζεται έλεγχο. Αυτή λοιπόν η οδηγία αποτελεί μια σημαντική λύση. Πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν τους ε, καταγγέλλοντες. Αυτό είναι το θέμα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω και να σας επενθυμίσω ότι πρόκειται για πραγματικούς ήρωες που έχουν πληρώσει με τη ζωή τους ε, τα, τις αποκαλύψεις αυτές και για τα σκάνδαλα του LuxLeaks. Όλη αυτή η πρόοδο μα για τη μεγαλύτερη πρόοδο την οφείλουμε πραγματικά σε αυτούς τους θαραλέους ανθρώπους και αυτοί λοιπόν θα πρέπει να προστατεύονται για να ευχαριστήσω την Βερζινή λοιπόν, να ευχαριστήσω την κυρία Γιούρεβα, την Επίτροπο, να ευχαριστήσω όμως και όλους εκείνους τους ευρωβουλευτές οι οποίοι συνέβαλαν στην ε, νομοθεσία αυτή γιατί πραγματικά χρειάζεται ένα κοινοβούλιο με συνείδηση των καθηκόντων του, το οποίο θα συνεργάζεται και θα αναλαμβάνει πραγματικά το δικαίωμα και της πρωτοβουλίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ζολή για ένα λεπτό από τους πράσινους. Ευχαριστώ. Η οδηγία αυτή αύξαν τις πιθανότητες να βελτιώσουμε τη ε, προστασία των πολιτών στην Ευρώπη. Αυτό χρειάστηκε λοιπόν μεγάλη δουλειά και μεγάλη αισιοδοξία. Η Ευρώπη λοιπόν όπως είναι δεν είναι το όνειρο των οικολόγων, αλλά δεν την απορρίπτουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 είχε δηλώσει ότι ένα κείμενο για την προστασία των καταγγελόντων δεν θα μπορούσαμε να το ε, κοιτάξουμε σε μόνιμη βάση. Εμείς ε, αποδείξαμε το αντίθετο. Καταρτήσαμε λοιπόν τη δική μας οδηγία για να καταδείξουμε προς τον ε, κύριο Γιούγκερ ότι αυτό δεν μπορεί να, αποφασίσει, να αποτελέσει πρόφαση για την αδράνεια. Γιατί κατά βάση θέλουμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας, ε, να μην ε, υποκρινόμαστε ότι πρόκειται για το απόρριτο. Θα πρέπει λοιπόν και ο υπεύθυνο τη αποκάλυψη των LuxLeaks ε, να αποτελέσει ένα παράδειγμα. Να προστατεύσουμε λοιπόν τους καταγγέλλοντες, γιατί αυτό το πετύχαμε χάρη στην επιμονή μας. Μία νίκη η οποία κόστισε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά και εμένα προσωπικά. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι συμφωνούμε με την αρχή ότι όλοι συμπερασπίζουν ε, το κοινό συμφέρον ε, χρήζουν προστασία. Αν συμφωνούν, ε, γιατί συμφωνούμε ότι η πράσπιση του κοινού συμφέροντος αφορά όλους χωρίς εξαίρεση. Αλλά γιατί αν ισχύει αυτό δεν συμφωνούμε το λέω ότι οι καταγγέλλοντες αν βρουν προς το συμφέρον όλων πρέπει να, χρήζουν, να χαίρουν προστασία. Κανένας δεν αμφισβητεί ένα εργαζόμενο να μπορεί να καταγγείλει παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων στην αρχή προστασία τη εργασία. Αυτή είναι διαφοροποιεί λοιπόν αυτό τον εργαζόμενο από έναν άλλο ο οποίο ε, ανακαλύπτει ότι φοροδιαφεύγει η επιχείρησή του. Ε, Προφανώ η, αρχή αυτής, ε, η εφαρμογή αυτή τη αρχή υποχρεώνει στο να έχουμε μια σοβαρή και ισορροπημένη προσέγγιση. Τώρα, η οδηγία που συζητάμε σήμερα είναι ισορροπημένη και λογική και ουσιαστικά στρέφεται σε αυτούς που ε, βλέπουν ε, ότι υπάρχουν ε, κάποιες παρανομίες. Το κείμενο δίνει μία λεπτή ισορροπία μεταξύ του καθήκοντος της καταγγελίας και της προστασίας των συμφερόντων του κράτους χωρίς να υπάρχει εμπλοκή στο εθνικό συμφέρον μεταξύ της δημιουργίας ιστορικών καλλιών για την προστασία των καταγγελόντων και το οικονομικό δικτύπου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα λογικό κείμενο που πρέπει να υποστηρίξουμε και υπερασπίζει το κοινό συμφέρον. Σας ευχαριστώ κυρία Γκόμε. Αυτή η οδηγία ε, αφορά τη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταγγέλλοντες ε, είναι ε, απαραίτητοι για να καταγγέλουν παρανομίες. Το άρθρο 38 της Οδηγίας της νομιμοποίηση Παράνομων Εσόδων ήδη επιχρεώνει τα κρατημέλη να δημιουργήσουν μηχανισμούς προστασίας ακόμη και για καταγγέλλοντες ε, στα πλαίσια τέτοιων οργανισμών. Οι εξεταστικές ε, επιτροπές στο ε, Κοινοβούλιο συζήτησαν τις δολοφονίες του Γιάνν Κούτσακ και της Δάφνης Καρουάνα. Είδαμε ε, την ε, δικαστική δίωξη του Άλμερ στην Ελβετία ε, και στην Πορτογαλία είδαμε το σκάνδαλο του Football Leaks. Υπήρξαν και κάποιοι δικηγόροι που φαίνεται να επηρεάζουν τη δικαιοσύνη και ε, δεν δράει δικαιοσύνη για να τιμωρήσει τους εγκληματίες. Ε, θα ζητηθεί ε, λοιπόν να λογοτήσει ο κύριος Πίντο, όπως έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει ο Ρουι Πίντο να προστατευτεί ως καταγγέλλοντες. Ευχαριστώ Βερζινή, Ροζιέρ και κυρία Επίτροπε και όλους τους συναδέλφους που εργαστήκατε για την οδηγία αυτή. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. πολύ. Η η επόμενη. E ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Βερσινή. Δεν είναι χωρίς ε, συγκίνηση που απευθύνομαι στο σώμα για τελευταία φορά. Κλείνει ένας κύκλος με την έγκριση αυτής της βασικής οδηγίας ε, για την οποία παλέψαμε και στο ίντερνετ από, από την αρχή της θητείας προστατεύοντας με, ελάχιστο, με κατελάχιστον τουλάχιστον τους καταγγέλλοντες όπως οφείλουμε προς αυτούς οι οποίοι ε, κατήγγυλαν μια σειρά παραβιάσεων που είναι άνθρωποι που ε, αξίζουν προστασία όχι αντίπεινα και καταδίκη γιατί προστατεύουν το, το δημόσιο συμφέρον και ελπίζω ότι αύριο το Κοινοβούλιο θα δείξει και συμπαγή στάση και ισχυρή θέση. Ε, είμαι ακόμα πιο πεπισμένη σήμερα για το ότι πρέπει να δώσουμε μια σωστή απάντηση σε αυτό το, ζήτημα και το καλύτερο νομίζω που αυτά τα πέντε χρόνια μου αφήνουν είναι ότι ανακάλυψα πως με πολλούς συναδέλφους συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες, κάνουμε τους ίδιους αγώνες και προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις στα ίδια ερωτήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Προχωρούμε. Ο κύριος Κάζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προστασία των ατόμων αυτών είναι βασικό, βασική επιτυχία του Κοινοβουλίου επιτρέπει να προστατεύουμε τους ανθρώπους αυτούς ανεξάρτητα από το αν καταθέτουν εσωτερικά ή εξωτερικά τις πληροφορίες τους σε ευρωπαϊκές ή εθνικές αρχές. Εγώ ζητούσα να υπάρξει μια τέτοια ευρωπαϊκή ρύθμιση για χρόνια. Χαίρο διότι τώρα θα παρασχεθεί προστασία όταν υποβάλλονται καταγγελίες για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου είχα την ευκαιρία να δω πολλές φορές πόσο σημαντική και πόσο θαραλέοι είναι οι πληροφοριοδότες, ακόμα και οι ε, ερευνητές δημοσιογράφοι μεταξύ αυτών. Προφανώς εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην Ντάφνη Καρουάνο Γκαλίτσια που δολοφονήθηκε και τους πληροφοριοδότες που δεν, που δεν λαμβάνουν προστασία από τη Μάλτα. Περάσαμε πολλά, πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιούροβα για την προστασία που πάλεψε να παράσχει. Θέλω να ευχαριστήσω την Άννα Γκόμενς, την κυρία Μακοβέη και άλλους συναδέλφους που διαπίστωσαν την κατάσταση στη χώρα μας και που κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι να παρασχεθεί προστασία στους δημοσιογράφους. Ευχαριστώ διαδικασία του Catch Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι η προστασία των ε, μαρτύρων οι οποίοι βεβαίως έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τις αρχές και έτσι να μπορέσει να ξεκαθαριστεί η κατάσταση όπου έχουμε απάτες εκεί όπου υπάρχει φόρο διαφυγή εκεί που υπάρχει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. και η συζήτηση αυτή για τους καταγγέλλοντες έχει γίνει επανειλημμένα και εδώ και στην επιτροπή αναφορών και νομίζω ότι τα βήματα που παίρνουμε είναι ιδιαίτερα σημαντικά διότι εάν δεν υπάρξει η προστασία αυτών των ανθρώπων δεν θα αποκαλυφθούν όσα σκάνδαλα έχουν υπάρξει. είχαμε το πρόβλημα των luxleaks είχαμε τεράστια φοροδιαφυγή είχαμε παράνομη λειτουργία των πολυεθνικών. όλες αυτές οι λειτουργίες και οι ενέργειες μπορούν να έρθουν στο φως και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι από τις δημόσιες αρχές μόνο όταν υπάρχει η προστασία των καταγγελόντων. θεωρώ σημαντικές τις ενέργειες που πράττουμε στον τομέα αυτό. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η προστασία των ε, μαρτύρων του δημοσίου συμφέροντος είναι ένα σοβαρό αλλά και ευαίσθητο θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όποιος καταγγέλει μια πράξη η οποία βλάπτει το δημόσιο συμφέρον όπως παραδείγματος χάρη διαφθορά, απάτες, ε, φοροδιαφυγή, ε, μόλυνση περιβάλλοντος, παραβίαση πυρηνικής ασφαλείας και ούτω καθεξής, συμβάλλει αποφασιστικά όχι μόνο στο να αποφευθούν αυτέ οι παράνομε ενέργειε αλλά και να λειτουργήσει ομαλά το κράτο δικαίου. για τον λόγο αυτό πρέπει να προστατεύονται οι μάρτυρε αυτοί. σε διαφορετική περίπτωση αν αποκαλυφθεί η ταυτότητά του υπάρχει κίνδυνο να γίνουν αντικείμενα απειλών επιθέσεων και οπωσδήποτε εκφοβισμού και θα πάψουν από εκεί και πέρα να αναφέρουν οποιαδήποτε παρανομία υποπίπτει στην αντίληψή του. πρέπει όμω να, να λαμβάνεται υπόψη ώστε οι προστατευόμενοι μάρτυρε να μην συκοφαντούν και να μην εκβιάζουν πολύ δε περισσότερο να μην χρησιμοποιούνται ως ψευδομάρτυρες σε δίκες πολιτικού περιεχομένου. με βάση τα προαναφερθέντα θεωρώ ότι η έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να την υποστηρίξουμε. ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Γιούροβα για τρία λεπτά εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρε, Αγαπητοί βουλευτέ, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τι παρεμβάσει σα και θα ήθελα και εγώ να σα ενθαρρύνω να υπερψηφίσετε το συμβιβασμό ο οποίο επιτεύχθη για την πρόταση αυτή και κρίνοντα και από τη συνολική ε, θετική ε, ατμόσφαιρα, ελπίζω να υπερψηφιστεί η πρόταση αύριο. Όπως πολλοί σας αναφέρατε, όντως θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην εξασφάλιση για τη σωστή υλοποίησης και πλήρους υλοποίησης και εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ροζιέρ για να κλείσει τη συζήτηση. Έχετε δύο λεπτά το λόγο και σας ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους, την παρότριση που δίνουν να τους ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, αλλά και την Επίτροπο και την Ρουμανική Προεδρία. Μην ε, νομίζουμε όμως ότι η συνένεση που ακούμε για το κείμενο σήμερα δείχνει ότι δεν υπήρχαν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις. Αναφέρθηκε ήδη. Πρώτα πρώτα είχαμε πίεση χρόνου. Είναι πολύ θετικό το ότι συλλογικά μπορούμε να καυχηθούμε ότι καταφέραμε να συμφωνήσουμε για ένα κείμενο πριν το τέλος της θητείας μας. Δεν ήταν εύκολο και όπως συχνά όλοι λένε ότι είμαστε υπέρ της προστασίας των πληροφοριωτών, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχαμε και κάποιες ε, αντιρρήσεις, ιδίως από κάποια κράτη στο Συμβούλιο. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας και της ενημέρωσης των συμπολιτών μας πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι τα πράγματα δεν ήταν απλά πάντα και κάποια κράτη-μέλη όχι τα μικρότερα, Γαλλία, Αυστρία, Ουγγαρία, προσπάθησαν να μειώσουν την εμβέλεια του κειμένου. Εμείς το κερδίσαμε τον αγώνα χάρη στην κινητοποίηση όλων, ιδίω και των ΜΚΟ, που θέλω εκ νέου να ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν ε, μέχρι τώρα. Ε, πραγματικά ε, να ευχαριστήσω επίσης και τη Ρουμανική Προεδρία για να υπάρξει μια συνένεση από τους συναδέλφους εδώ που άσκησαν πίεση στις κυβερνήσεις τους. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα του ρόλου του Κοινοβουλίου που μιλά ως εκπρόσωπος των πολιτών, παρεμβαίνει στην νομοθετική διαδικασία προς όφελος των πολιτών και αυτό είναι κάτι σημαντικό ιδίως εν ώψη και των ευρωεκλογών. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εκ νέως. Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία συνάδελφοι. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Συνάδελφοι, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Ρουμανία. Δίνω το λόγο πρώτα πρώτα στην κυρία Γιούροβα για να μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Κομισιόν ξεκαθάρισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και παραπέρα, ότι παρακολουθεί εκ του συνεγγύς και με πολύ μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν το κράτος δικαίου στη Ρουμανία. επανειλημμένα έχουμε πει ότι η Ρουμανία θα πρέπει να επιστρέψει στην μεταρρυθμιστική διαδικασία και μάλιστα κατεπηγόντως. Αυτό σημαίνει να πάει προς τα μπρος, όχι προς τα πίσω και να απόσχει από οποιοδήποτε βήμα που ε, ουσιαστικά αναιρεί την πρόοδο των προηγούμενων ετών. Η Κομισιόν και συγκεκριμένα ο πρώτος αντιπρόεδρος, ο Φρανς Τίμερμανς, προσωπικά έχει δεσμευτεί με την Πρωθυπουργό Νταντσίλα και οι εμπειρογνώμονε συναντήθηκαν πολλές φορές για επικοδομητική συζήτηση και διάλογο. Η Κομισιόν πάντοτε ξεκαθάρισε ότι <laughs> ο διάλογος για χάρη του διαλόγου δεν θα αρκεί και ε, αναμένουμε συγκεκριμένε δράσεις από την ρουμανική πλευρά και μάλιστα πολύ σύντομα. Η Επιτροπή συζήτησε την κατάσταση πριν δύο εβδομάδες. Δυστυχώς δεν ε, μπορέσαμε ακόμη να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι έχει επανέλθει στην ορθή οδό η Ρουμανία. Αν ε, δεν ε, διασκεδαστούν οι ανησυχίε μα, θα πρέπει να αναλάβει δράση η Κομισιόν και να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή τη. Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά τεχνικά ζητήματα ή να σα ενημερώσω ε, για ε, την ε, υπαναχώρηση που είδαμε στι συστάσει του μηχανισμού CVM. Εκεί υπάρχει τελμάτωση. Ή να συζητήσουμε ότι οι τελευταίε εξελίξει νομοθετικέ στη Ρουμανία για τη μεταφορά πολλών οδηγιών στο εσωτερικό δικαίωμα δίκαιο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανησυχίε με πιθανή συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο ή να αναφέρουμε περαιτέρω διάβρωση ε, της ε, εμπιστοσύνης ε, και διαφόρες αυθαίρετες διαδικασίες διορισμών. Ε, επίσης, η διαδικασία για την επιλογή της ε, μελλοντική Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, δεν έχει συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήματος. Βλέπουμε επαναχώρηση στο κράτος δικαίου στη Ρουμανία και κυρίως σε ό,τι αφορά την αμεροληψία του δικαστικού σώματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Καταρχήν, οι πιθανέ τροποποίησει του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινική δικονομία. Τέτοια θεμελιώδη ζητήματα χρειάζονται πολύ προσεκτική προετοιμασία, διαβούλευση με το δικαστικό κλάδο και τα ενδιαφερόμενα μέρη και πολύ σαφή κατανόηση των αλλαγών. οποιοδήποτε δράση αναλυφθεί θα πρέπει να συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις καθώς και με τις συστάσεις του μηχανισμού CVM, όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς οι ρουμανικές αρχές ε, θα ε, αναλάβουν κίνδυνο αν προχωρήσουν ε, χωρίς να ακολουθήσουν μια τέτοια διαδικασία και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να έχουμε μια de facto συστημική ατιμορρησία για υψηλούς εξωματικούς που έχουν καταδικαστεί για διαφθορά. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο ε, και μία πιθανή συνέχιση μίας ε, δικαστικής απόφασης ε, που ζήτησε στον να αλλάξει σύνθεση πέντε δικαστικών σχηματισμών δεν ε, μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτό το θέμα από τις ε, σημαντικές ε, συνέπειες του να ξανανοίξουν παλιές υποθέσεις. Κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική παρέμβαση στην αμεροληψία της δικαιοσύνης. Ο κίνδυνος μαζικών προβλημάτων στο ρουμανικό ποινικό σύστημα και πάρα πολλών περιπτώσεων διαφθοράς δεν μπορεί να γνωριθεί. Τρίτον, το θέμα των διορισμών των εισαγγελέων και συγκεκριμένα η ανάγκη για ένα εύρωστο και αμερόληπτο σύστημα του διορισμού των επικεφαλής εισαγγελέων. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα, όμως ο μηχανισμός ελέγχου και ισορροπιών έχει καταψηφιστεί επιτυχώς. Το αποτέλεσμα είναι ε, μία επίμαχη διαδικασία για το να διεριστούν οι ενότατοι εισαγγελεί. Ο Γενικός Εισαγγελέας ε, και ε, ο επικεφαλής εισαγγελέας καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης, τα τμήματα ε, της εισαγγελία που έχουν να κάνουν ε, με το διορισμό των ε, ανακριτών. Έχουν αναφερθεί ανησυχίε στην έκθεση CVM από την Επιτροπή της Βενετίας και από τον Γκρέκο. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση ενισχύει τη δομή αυτή. Όλα τα στοιχεία αυτά, όλα τους, προκαλούν μεγάλες ανησυχίες ε, αν τα δούμε και μονομένα. Ενώ όλα μαζί ουσιαστικά δημιουργούν μια ιδιαίτερα ανησυχητικό. Να τους τελευταίους μήνες ε, είδαμε μια ιδιαίτερα σταθή κατάσταση στη Ρουμανία με μια σειρά βιασμένων αποφάσεων ε, που ελήφθησαν και ουσιαστικά ζητήματα. Αν οι ανησυχίε αυτέ δεν διασκεδαστούν, η Κομισιόν θα πρέπει να δράσει και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή τη. Επομένω, η Κομισιόν παροτρύνει τη Ρουμανία να ε, διαβουλευθεί και να φτάσει σε μία συνένεση, να ακολουθήσει τις συμβουλές της Επιτροπής της Βενετίας, ε, καθώς και τις διαδικασίε του CVM. Δεν είναι πολύ αργά για τη Ρουμανία για να ε, επανέλθει στις μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε, δύο λεπτά για το ΕΛΚ έχει το λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώ δεν μπορούμε να καλωσορίσουμε και την Προεδρία παρά το γεγονό ότι θα ήταν ε, πάρα πολύ ε, καλή λόγη να, παρα, να παραστεί εδώ η Προεδρία. Θα πρέπει να σα πω ότι ανησυχώ, ανησυχώ, γιατί ποτέ δεν έχουμε τόσο γρήγορα δει κατάρρευση του κράτου δικαίου όπω στη Ρουμανία και αυτό δεν έχει παρουσιαστεί σε κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω η Ρουμανία να αποτελέσουν την εξαίρεση. Και καλό θα ήταν να είχαμε ε, δράσει και να έχει δράσει η Ρουμανία πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα. Αυτό που έχουμε να προτείνουμε προτείνουμε βάσει του άρθρου 7 να σταματήσουν οι πόροι, γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε του πόρου αυτού δεδομένη και τη κατάρρευση του κράτου δικαίου, γιατί η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την είναι από ό,τι φαίνεται υπερβολικά επιβαρημένη η Προεδρία ή η ρουμανικη κυβέρνηση είναι και θύμα και θήτης. Και το πρώτο θύμα είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί ουσιαστικά προωθείται έτσι η διαφθορά. βλέπουμε λοιπόν έναν πρόεδρο α, της, από τους σοσιαλιστές του Κοινοβουλίου, ο οποίος α, κατηγορείται και α, η, αυτή η ιστορία θα πρέπει να ακολουθηθεί και από του σοσιαλιστέ και δημοκράτε, γιατί αυτά τα δύο μέτρα και σταθμά είναι κάτι πολύ αρνητικό. Και βλέπουμε λοιπόν α, α, τη διαδικασία της εισαγγελέως, της πρώην εισαγγελέως, η οποία κατηγορείται με διάφορα προσχήματα διαρκώς για εκδίκηση. Είναι υποψήφια των δύο α, μα, μεγάλων κομμάτων για τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα για να προστατευτεί η εισαγγελέας, υποψήφια εισαγγελέας και υπάρχει διάθεση να ανταμείψουμε ακόμα για την Ρουμανία για την παρτυπή αυτή. Αυτό πραγματικά δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί γιατί η Η υποψηφιότητα αυτή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί μήνυμα φιλοσοφική σε ό,τι αφορά κατάφορες παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Κυρίε και κύριοι, το θέμα λοιπόν είναι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το θέμα είναι η αξιοπιστία και της Επιτροπής, του πρώτου, πρώτη Αντιπροέδρου και όλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και έχουμε μία μπλε κάρτα, κυρία Κρέσλε. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την μπλε κάρτα. Θα ρωτήσω λοιπόν την εξή ερώτηση στα αγγλικά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ερμενία. Είπατε στην παρέμβασή σας ε, κάποια τρομερά πράγματα για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πώς μπορείτε να εξηγήσετε στους Ρουμάνους ότι στη δική σας χώρα τα μέλη του συνταγματικού δικτύου μπορούν να είναι και κομματικά στελέχη, μέλη του κόμματος. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή. Δεν είπα ότι το συνταγματικό δικαστήριο έχει πολιτικά κίνητρα. Το θέμα είναι αν οι πολιτικοί τηρούν το δίκαιο εγώ προασπίστηκα τι αποφάσει του συνταγματικού δικαστηρίου για την υποποίηση από του πολιτικού. Αυτό είναι το θέμα. Και έχει έρθει το πρόβλημα του χρόνου οι σοσιαλιστέ να, να τοποθετηθούν από αυτόν. Γιατί να ψηφίσουν λοιπόν οι Ρουμάνοι όταν πρόκειται για ρουμανικά ζητήματα. Αυτό είναι θέμα ολόκληρη τη Ευρώπη. Εγώ το είδα και στην υποψήφια του Εθνικού Συνεδρίου δεν μας είπε την αλήθεια τουλάχιστον. Το λιγότερο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που είχε. Το είδαμε για τους υποψηφίους, την υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πότε επιτέλους ε, οι σοσιαλιστές θα αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά σαν ευρωπαϊκά θέματα. Δεν είναι ρουμάνικο το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συντό συγγνώμη, λέει η πρόεδρο. Συνεχίζεται η συζήτηση. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο Ιωζεφ Βάιντεν Χόλτσερ από του Σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ πολύ. Αντίθετα με αυτά που είπε η προελαλήσασα, πιστεύω ότι η Ρουμανική Προεδρία η οποία έχει πετύχει πάρα πολλά στο σύντομο χρονικό διάστημα που είχε στη διαθέσή τη. Πολλά κατάφερε λοιπόν να πετύχει παρά τις αντίξωε συνθήκε. Γι' αυτό λοιπόν, μα κύριε Πρέντα, ακούστε με, σας παρακαλώ λίγο ε, πειθαρχία. Γι' αυτό λοιπόν είναι τόσο περίεργο το γεγονός ότι σήμερα αυτή η κατεπίγουσα συζήτηση πρέπει να γίνει. Αυτό το θέμα δεν το συζητάμε για, σε πρώτη φορά, για πρώτη φορά. Το Νοέμβριο το Κοινοβούλιο ξεκαθάρισε σε ψήφισμα ότι το θέμα της δικαιοσύνης και των ποινικών διώξεων στην ε, Ρουμανία δεν ε, μπορεί να απειλεί την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος αν θέλουμε να καταπολεμούμε την διαφθορά. Ο έλεγχος και ο έλεγχος θα πρέπει να εγγυώνται και ο κοινοβουλευτικό έλεγχος ε, των ε, μυστικών υπηρεσιών. Δυστυχώ, ε, οι αξιώσει μα δεν ε, λήφθησαν σοβαρά υπόψη. Αυτό μα λυπεί ιδιαίτερω. Το θέμα λοιπόν δεν είναι συγκεκριμένα να στραφούμε κατά τη Ρωμανία. Το θέμα είναι η κοινή ερμηνεία του δικαίου. Ένα εύρυθμα λειτουργών κράτο αποτελεί πυλώνα τη κοινή Ευρώπη. Και αυτό σαφώς θα τα ορίζεται στα κριτήρια της Χάγης. Η τήρηση λοιπόν των κριτηρίων αυτών και η αιμονή στην τήρηση των κριτηρίων δεν αποτελεί θέμα ιστορικό ενό κράτου μέλους, αποτελεί ε, κάτι που αφορά όλους μας και φυσικά δεν μπορεί να γίνεται μονομερός και να αποφασίζεται μονομερός, αλλά τα κοινά αυτά, οι κοινέ αυτές αρχές θα πρέπει να καθορίζονται μέσω διαλόγου. Αυτό είναι το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε προ το Βουκουρέστι. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί από κοινού η Ανατολή και η Δύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο, και τώρα το λόγο έχει η Μόνικα Μακοβέη από το ECR. Σήμερα στη Ρουμανία μια ομάδα διαφθαρμένων πολιτικών ε, με επικεφαλή στον καταδικαστέντα Ντράγκνε, ο οποίο τελεσίδικα έχει καταδικαστεί και έχει και νέε δίκε. Ε, κρατάει όμοιρο ε, τη χώρα. Δεν σέβεται το πρόγραμμα διακυβέρνηση που είχαν ανακοινώσει στι εκλογέ. Αλλάζουν τον νόμο, σβήνουν παραβιάσει και ουσιαστικά πολιτικά ασκούν έλεγχο στου δικαστέ και χρησιμοποιούν χρήματα από τι επενδύσει για να δίνουν μίζες, καταστρέφουν την έννοια τη δημοκρατία. προκειμένου αυτή η διεφθαρμένη πολιτική να την κλειτώσουν από τη δικαιοσύνη ε, και ε, τελικά κρατούν ε, όμοιρο 20 εκατομμύρια ανθρώπους για να σωθεί μόνο ένας οι Ρουμάνοι ε, δεν είναι αδρανείς. Εδώ και δύο χρόνια βγαίνουμε στο δρόμο, ε, μας ρίχνουν δακρυγόνα, μας χτυπάνε, μας ρίχνουν πλαστικές ε, σφαίρες ή χειροβομβίδες. Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να κατεβαίνουμε στο δρόμο. Και στη συνέχεια ο δρόμος μας είναι η Ευρώπη βλέπουμε με απελπισία την καταβήθηση της χώρας ε, που ε, τη χτυπούν ο Ντράγνε, ο Ταριτσάνου και άλλοι. Εγώ όμως δεν μπορώ να σιωπάσω, δεν μπορώ να ε, μας κρατούν όμοιροι κάποιοι εκατοντάδες πολιτικοί που ασκούν την εξουσία σας. Ζητώ να βοηθήσετε την ε, Ρουμανία γιατί η Ρουμανία σήμερα ζει μια εγκληματική δικτατορία και την τραγωδία του αδειάσματος της χώρας. 4 εκατομμύρια Ρουμάνοι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Η απομάκρυνσή μας από την Ευρώπη είναι ο εφιάλτης που ζήσαμε εδώ και δεκαετίες. Αυτό είναι το τελευταίο τρένο το οποίο μπορούμε να πάρουμε. Θέλουμε να είμαστε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Η κυρία Έντφελ. Για τρία λεπτά. Yes, thank you. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Επίτροπο. Ξεκινώ λέγοντας ότι συμφωνώ με την ενόχληση της κυρίας Γκρέσλε για την απουσία του Συμβουλίου. Πόσο μάλλον που η Προεδρία είναι η χώρα την οποία συζητούμε. Μην χειροκροτάτε ακόμα, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που θα πω μετά. Λυπάμαι επίσης διότι δεν είναι εδώ ο κύριος Τίμερμανς δεν θέλω να σας προσβάλλω κύριε Επίτροπε, αλλά είναι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για το θέμα. Τι έκανε για το θέμα αυτό τα τελευταία πέντε χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα μόνο υπέβαλε η Επιτροπή μία ανακοίνωση για το κράτος δικαίου που στην ουσία δεν άξιζε το χαρτί που ήταν πάνω στο οποίο ήταν ε, γραμμένη και δεν εμφανίστηκε καν ο κύριος Τίμερμαν στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών για να το παρουσιάσει. Πού είναι σήμερα. Ε, τι έκανε τελευταία πέντε χρόνια. Εγώ πραγματικά κουράστηκα να συζητώ σήμερα για την Ρουμανία, λείπει το ΕΛΚΑ. Αύριο Ουγγαρία, οι σοσιαλιστές θα κριτικάρουν, θα επικρίνουν τους, ε, το, ε, το, το, το ΕΛΚΑ Ξέρω, κάποιοι φωνάζουν γι' αυτό, δεν θέλω να το πω όλου. Ε, η κυρία Γκρέσλε διαμαρτύρεται, αλλά το θέμα γίνεται τελικά πάντα κομματικό. Δεν είναι κομματικό το θέμα. Το θέμα είναι για τις αξίες που περιλαμβάνει το άρθρο 2 της συνθήκης, που μας αφορούν όλους, ανεξάρτητα από το πολιτικό μας χρώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δυόμιση χρόνια πριν το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μία θέση, μία, υπέβαλε μία πρόταση για ένα γενικό μηχανισμό κράτους δικαίου που καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, όλες τις κυβερνήσεις. Η Επιτροπή και δεν με με εσά, κύριε Επίτροπε, ο κύριος Τίμερμανς είναι ο υπεύθυνο. είπε δεν το χρειαζόμαστε γιατί έχουμε όλα τα εργαλεία στην εργαλειοθήκη που χρειαζόμαστε. Δεν τα έχουμε. Ο κύριος Τίμερμανς είναι Spitzenkandidat και ο κύριος Βέμπερ το ίδιο, υποψήφιοι για πρόεδρο της Επιτροπής και οι δύο. Γιατί λείπουν και οι δύο υποψήφοι. Τι προτίθεται να κάνουν όταν, αν γίνουν πρόεδροι της Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής κύριος Βέμπερ θα κάνει αυτό που υπερψήφισε ως ευρωβουλευτής. Δηλαδή θα προτείνει πλήρη μηχανισμό προστασίας του κράτους δικαίου που θα αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Τελειώνω, πρόεδρε. Η ομάδα μου, η φιλελεύθερη, σαφώς και ξεκάθαρα απομακρύνθηκε από το αδελφό Ρουμανικό κόμμα. Όχι μόνο για παραβιάσεις ε, των, ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου, αλλά για μια σειρά άλλων νομοθετικών κειμένων ε, γάμο για όλους. Ε, είμαστε εξαιρετικά απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά και την προσπάθειά τους να εμποδίζουν την ε, καταχώρηση και τις υποψηφιότητες νέων, ευρω... νέων κομμάτων που θέλουν να κατέβουν στις ευρωεκλογέ. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα κύριε Πρέντα. Συμφωνώ με την επίκρισή σας για την Επιτροπή και τον κύριο Τίμερμανς, κύριε Ιντερνβέλτ, και δεν θέλω να κάνω κομματική συζήτηση, αλλά ο κύριος Φερχόφστατ, επικεφαλής της ομάδας σας, δεν είπε τίποτα μέχρι. Σιώπησε. Ε, το πρόβλημα δεν ξεκίνησε πριν από τρεις μήνες. Όταν είχαμε ζητήσει να κάνετε κάτι, μείνατε ε, στο περιθώριο. Τώρα μετράτε την, κατάσταση εν ώψη των εκλογών και εσείς κυρία μου. Γιατί ο κύριος Φεχόφστατ, πείτε μου, δεν είπε τίποτα τότε από πολιτική φιλία ε, με τον κύριο Τριτσάνο, από, μετράνε περισσότερο οι προσωπικές φιλίες από την πραγματικότητα, πείτε το μου. Λάθος κάνετε. Δείτε τα πρακτικά της Ολομέλειας. Η στάση της ομάδας μας ήταν πάντα ξεκάθαρη. Αν ήταν εξίσου ξεκάθαρη και η θέση του ΕΛΚ, δεν θα είμαστε στην κατάσταση που είμαστε τώρα με την Ουγγαρία. Είμαστε εξαιρετικά αρνητικοί και κριτικοί σε αυτά που συμβαίνουν στη Ρουμανία. Επίσημα απομακρυνθήκαμε από το κόμμα των φιλελευθέρων που είναι στην συγκυβέρνηση σαν Ευρωπαϊκό Κόμμα και ζητήσαμε την απομάκρυνσή τους από την πολιτική μας οικογένεια. Το κάνουμε με βαριά καρδιά διότι έχουμε πολλά χρόνια πολιτικής φιλίας όντως, αλλά εμείς τιμούμε τις αρχές μας αντίθετα από το ΕΛΚ που ακόμα και τώρα δεν απομακρυνθήκε πλήρως από τον κύριο Όλμπαν. Διαβάστε λοιπόν τα πρακτικά της Ολομέλειας. Εγώ προσωπικά κύριε Πρέντα είχα συμμετάσχει στις συζητήσεις για τη Ρουμανία και ήμουν εξαιρετικά επικριτική. Να είστε κι εσείς εξίσου σε ό,τι φέρω το δικό σας μέλος, τον κύριο Όρμπαν. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σερτζαντίνη. Ο... Ε, έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Μποστινάρο και στην κυρία Ενετφέλτ. Θα δέχεστε. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη συνάδελφε, δύο σύντομες ερωτήσεις για σας. Ξέρετε πόσες φορές ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας χαρακτήρισε τις πράξεις της κυρίας ε, Κεβίση ως αντισυνταγματικέ. Ξέρετε πόσες φορές διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε το Ρουμανικό Σύνταγμα και μετά έχουμε την υπόθεση που γνωρίζετε τις κατηγορίες ε, περί κατάχρησης αξιώματος. Οι σημαντικότερε μαρτυρίε προέρχονται από δύο εισαγγελείς τη εθνική Διευθύνσης Καταπολέμηση τη διαφθορά. Αυτοί μαρτυρούν κατά αυτή, είναι οι βασικοί μάρτυρε. Πώ μπορείτε λοιπόν να μιλάτε για πολιτική πίεση σε τέτοιε περιπτώσει. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για δικαστικών υποθέσεων, αλλά πόσο ξέρω πρόσφατα το δικαστήριο αποφάσισε ότι η κυρία Κεβίση, μπορεί να τελειώσω. Θέλετε να με ακούσετε. Σας ενδιαφέρει η απάντηση. Έχω 30 δευτερόλεπτα και τα μισά πέρασαν ήδη. Αυτό που ξέρω είναι ότι πρώτα απ' όλα το δικαστήριο ήδη επέτρεψε στην κυρία Κιόβεση να ταξιδέψει και να εκφραστεί. Το θέμα είναι ότι τα επιχειρήματα που ακούω πάντα είναι... δεν κάνουν τα πράγματα καλύτερα, διότι η εικόνα που έχουμε εδώ είναι ότι υπάρχει ένα απόλυτο χάο. Και χρειαζόμαστε ένα κράτο δικαίου, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το ρουμανικό λαό, διότι οι νέοι άνθρωποι στη Ρουμανία διψούν για μια χώρα σταθερή, ε, για μια κυβέρνηση αξιόπιστη, μη διεφθαρμένη. Και ακούμε όλες τις ιστορίες, ε, ένα στο δικαστήριο, ε, οι μυστικές υπηρεσίες που παρεμβαίνουν. Όλα αυτά κάνουν τα πράγματα καλύτερα, δεν νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση κυρίας Αρτζεντίνα από τους Πράσινους δεν, το κράτος δικαίου δεν είναι αριστερό ή δεξιό και είναι πολύ οδυνηρό που βλέπουμε ότι η ρουμανική κυβέρνηση στηρίζει την Ουγγρική μην βάζοντα στην ημερήσια διάταξη στην έκθεση για την Ουγγαρία. Όλοι το είπαν, αλλά είναι πολύ απογοητευτικό. Η Ρουμανική Προεδρία δεν είναι εδώ. Απίστευτα πράγματα. Επίση, η Προεδρία απονομιμοποιεί τον υποψήφιο του Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και έτσι απονομιμοποιεί όλη τη διαδικασία. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι κρίσιμη στο κράτος δικαίου. Και έχουμε μια χώρα η οποία συνεχώς υπαναχωρεί και προεδρεύει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τούτη την ώρα. Άλλο παράδειγμα. Ξέρω τον Ιανουάριο του 2011 όταν η Ουγγρική κυβέρνηση είχε την προεδρία του Συμβουλίου Πάλι ένα εξάμεινο δεν έγινε τίποτε. Πραγματικά πρέπει να ντρέπονται γι' αυτό. Έξι εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογέ και έχουμε αυτή την κατάσταση εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώ ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι. Εκ μέρου του ΙΕΝΕΦ, ο κ. Μπάτεν. Ο κ. Μπάτεν δεν είναι εδώ. Περνάμε στον κύριο Λενάρ για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση χωρών που έχει συμπράξει για να δώσει έναν, μια μάχη ε, και να συνενώσει δυνάμεις. Αυτό γίνεται πάνω στη βάση ισχυρών θεμελίων κοινών αξιών μόνο. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση σήμερα. Και είδαμε έλλειμμα στις αντιδράσεις της Κομισιόν και η Πολωνία επίσης πρέπει να υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 7. Έχουμε και τη Ρουμανία, έχουμε τη Μάλτα που δεν τις έχουμε προσέξει ε, ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να εστιάσουμε στη Βαλέτα και τον Βουκουρέστι. Δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μπορούμε να προβάλλουμε την ένωσή μας, να τη στηρίξουμε όταν τα μέτρα είναι τα ίδια για όλους. Δεν πρέπει να παίζει ρόλο ε, η φιλία με το δικαστήριο στην περίπτωση της Μάλτας και της Ρουμανίας θα πρέπει άπαξ και διαπαντός να υπάρξει παρέμβαση της Κομισιόν. Ο κύριος Νίκα, 1,5, 2,5 ε, ε, λεπτά. Ξαναγίνεται μια συζήτηση προεκλογική. Είναι μια συζήτηση για την οποία πρέπει να πούμε πως ε, τελικά δεν μιλάμε για την Ρουμανία. Πολύ συχνά λέμε πράγματα χωρίς να είμαστε σαφής. Ποια είναι η κατάσταση του κράτους δικαίου. Χωρίς ελευθερίες για τους πολίτες δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το 2009 στη Ρουμανία υπογράφηκε ένα μυστικό πρωτόκολλο με την ε, μυστική υπηρεσία πληροφοριών. Αυτό το μυστικό πρωτόκολλο βγήκε στο φως, διέρευσε και αυτό αποκάλυψε σημαντικές παρανομίες και καταχρήσεις. Η Ρουμανία λοιπόν έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά στη δικαιοσύνη της. Σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα δικαιώματα των πολιτών. Τα ρουμανικά φαρμακευτικά προϊόντα, για παράδειγμα, δεν, έχουν τις, ε, δεν τυχαίνουν τις ίδιες μετακόμι, με, μεταχείρισης με άλλα προϊόντα της νέας εσωτερικής αγοράς. Το ίδιο και στα αεροδρόμια, ε, στους λιμένες από τη μια μεριά πηγαίνουν Ρουμάνοι, από αλλού πηγαίνουν οι υπόλοιποι. Ε, το 90% των Ρουμάν πολιτών θεωρεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν ε, θεωρούν ε, τις παραβάσεις και τις καταχρήσεις που έχουν γίνει στη δικαιοσύνη. Στη Ρουμανία ο πληθυσμό, η κοινή γνώμη είναι πολύ ευαίσθητη σε θέματα δικαιωμάτων λόγω του κομμουνιστικού παρελθόντος. Δεν θέλουμε να εκβιαζόμαστε. Δεν θέλουμε να ε, κινηματογραφείται η προσωπική ζωή των εισαγγελέων στην Ρουμανία προκειμένου να εκβιαστούν μετά. Θέλουμε να μας μεταχειρίζονται με, τους ίδιους, ε, με τον ίδιο τρόπο ε, που μεταχειρίζονται τους πολίτες σε όλες οι υπόλοιπες χώρες. Αυτοί που έχουν αυτιά ας ακούσουν και αυτοί που έχουν μάτια α δουν. Η Ρουμανία ε, αξίζει περισσότερο. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ρουμανία είχε ενταχθεί στο μηχανισμό αξιολόγηση και ε, του, του κράτους δικαίου ε, της Κομισιόν και έχει επικριθεί για πρακτικές ε, σχετικά με την απόδοση δικαιοσύνης. Πριν από μερικές εβδομάδες, ε, αρχηγοί ε, των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν από τα δικαστήρια της Ρουμανίας να σταματήσουν έρευνα που γίνεται εναντίον ε, γίνονται σχετικά με Ρουμάνο πολίτη ε, που είχε υποστεί παραβίαση των δικαιωμάτων του. Το Ανώτατο ε, Δικαστικό Συμβούλιο της ε, Ρουμανίας είπε ότι ο Ταγιάννη, ο Φερχόφστατ και ο Βέμπερ μέσω των δηλώσεών τους θέτουν πίεση στους εθνικούς δικαστές που έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση και υποσκάπτουν την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη στη Ρουμανία. Οπότε, συνάδελφοι, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αρχίστε να συμπεριφέρεστε όπως ζητάτε από τους άλλου πολιτικούς να συμπεριφέρονται. Ευχαριστώ. Ο κ. Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεν εκπροσωπείται εδώ η ρουμανική κυβέρνηση, παρόλο ότι το θέμα μας είναι ακριβώς η Ρουμανία. Κανείς δεν εκπροσωπεί εδώ λοιπόν την Προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό δείχνει την περιφρόνηση που δείχνει το Συμβούλιο προς το όργανο μας. Είναι πραγματικά κρίμα σε αυτή την πρώτη Ρουμανική Προεδρία να βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση. Κάποιος θα έπρεπε να είναι εδώ. Όμως το καθεστώς του Βουκουρεστίου ε, δεν συνδέεται πλέον με το κράτος δικαίου. Η πλειοψηφία που κυβερνά τη χώρα από το 2016 κάνει αυτό που είπε ο κ. Νίκα. <laughs> Ε, πιέζει τους εισαγγελείς και τους δικαστές και δημιουργεί ε, θεσμούς που θα οδηγήσουν, θα επιτρέψουν στην αναθεώρηση τελεσίδικων αποφάσεων ε, αποφάσεις που είχαν ληφθεί προκειμένου ε, να καταπολεμηθεί η ε, διαφθορά. Ο πρόεδρος τους έχει καταδικαστεί δύο φορές για διαφθορά, αυτός ο αστείος τύπος. Δείξτε μου μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, κυβερνάται από τέτοιο άνθρωπο. Άνθρωπος ο οποίος παρέμεινε στο αξίωμά του έχοντας καταδικαστεί δις. Καταδικάστηκε για απάτη. Πώς είναι δυνατόν να δεχόμαστε συμμαχίες τέτοιων ε, ανθρώπων που θα καταστρέψουν τη χώρα μας. Ευχαριστώ. Κυρία Γκραπίνη. Και κυρία Γκραπίνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ ε, αγαπητοί συνάδελφοι, να κάνω μια παρατήρηση. Αυτή η συζήτηση είναι μια αποτυχία, κύριε Επιτροπή. Το βλέπετε και από τον κόσμο που είναι εδώ. Δύο άνθρωποι είναι εδώ. Οι σημαντικότεροι ηγέτε δεν είναι εδώ, είναι δειλοί. Ε, θα έρθετε στη Ρουμανία, στη χώρα μου κύριε Βέμπερ και θα πείτε ε, να σταματήσει μια υπόθεση ενώπιον των δικαστηρίων. Κύριε Επίτροπε, ξέρετε ότι στον τομέα της δικαιοσύνης δεν μπορείτε να πάτε σε μια κυβέρνηση και να τους πείτε τι θα κάνουν. Ακόμη και αν είστε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και οι παρεμβάσει ε, των Ευρωπαίων αξιωματούχων έχουν επηρεάσει αρνητικά τη δικαιοσύνη στη Ρουμανία. Οι πολίτε στη Ρουμανία δεν καταλαβαίνουν γιατί ορισμένοι αξιωματούχοι και ευρωβουλευτέ ε, θέλουν να παρέμβουν σε υποθέσει ενώπιον ρουμανικών δικαστηρίων. Ναι, ε, είμαστε σε προεκλογική φάση. Ναι, το καταλαβαίνω, ναι. Ο κύριο Πρέντα το είπε ότι και εσεί έχετε προεκλογική εκστρατεία αυτή τη στιγμή. Οπότε το ΕΛΚ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κερδίσει κάτι από αυτή την εκστρατεία. Ε, Επίτροπε, θέλω να πείτε στου Ρουμάνου ότι δεν δώσατε ούτε ένα παράδειγμα παραβίαση του κράτου δικαίου. Ούτε ένα. Η ρουμανική κυβέρνηση έχει μια επιτυχή προεδρία. Λυπάστε που είχαν τόση επιτυχία, που ολοκλήρωσαν τόσα θέματα και τόσα αρχεία. Γιατί το κάνετε αυτό. Πέρυσι είχαμε ένα ψήφισμα, ήταν άδικο και το ξέρετε. Ξέρετε ότι υπάρχει κάτι σε αυτό το ψήφισμα το οποίο δεν θα λέγατε και καμιά άλλη χώρα. Ε, κατηγορείται τη Ρουμανία που άλλαξε τον επικέφαλή ε, ενός φορέα, ε, ο οποίο κατέστρεψε το φορέα αυτό, τη δικαιοσύνη. Μιλάμε για τι ζωέ χιλιάδων ανθρώπων, χιλιάδε δίκε που ακόμη και εσείς είχατε πει ότι έπρεπε να ξαναγίνουν. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, να υποφέρουν από την αδικία. Ποιον προστατεύεται η Ρουμανία. Δεν είναι ε, ένας άνθρωπος, ε, είναι 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο κύριος Πρέντα παρακαλώ. Θα δώσω τον κύριο, λόγο στον κύριο Χεκμάρκ. Κυρία Πρόεδρε, το να υπονομεύουμε την ανεξαρτησία του δικαστικού, η Τη ανεξαρτησία των εισαγγελέων, η παρεμπόδιση της δημιουργία νέων κομμάτων, απόπειρα νομιμοποίηση της διαφθορά, καταπολέμηση όχι της διαφθορά, αλλά αυτών που καταπολεμούν τη διαφθορά, το να σε ενοχλητικού ηγέτε ανεξαρτήτων φορέων, απαγόρευση εξόδου τους από τη χώρα, Φυσικά και μιλάμε εδώ για μια κατάρρευση του κράτους δικαίου. Και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η άρνηση. Αλλά πρέπει να πω όμως, ε, ε, κύριε Βιντεχόζερ, ότι η σιωπή των σοσιαλιστών είναι εκοφαντική. Η συμβολή σας εδώ, απόψε, δεν ήταν εντυπωσιακή, αλλά και θα σας πω γιατί. Η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας δεν ακολουθεί κομματικές γραμμές. Η κατάχρηση της εξουσίας στην Ουγγαρία και στην Πολωνία δεν αιτιολογεί την κατάχρηση εξουσίας στη Ρουμανία και άκουσα πολλούς από εσάς να το λέτε ε, πολύ ηχηρά για την Ουγγαρία όπως και εγώ και για την Πολωνία αλλά η σιωπή σας είναι εκοφαντική. Καταχράστε τις υποχρέωσή σα να υπερασπίζεστε τη δημοκρατία. Εσείς ως ηγέτες εδώ απόψε της ε, ομάδας των σοσιαλιστών. Είστε λάθος. Το λόγο έχει ο κύριος Αρβαμά για ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα πού είναι ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς δεν βλέπω. Η Ρουμανική Προεδρία πού είναι. Ούτε εκείνους τους βλέπω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε για να προωθήσει την ειρήνη, στις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου. Όπως και οι άλλοι συνάδελφοι του ΕΛΚ, ανησυχώ πολύ για τη Ρουμανία και το κράτος δικαίου εκεί, δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων. Η Ρουμανία επιχειρεί να προχωρήσει σε αλλαγή του ποινικού κώδικα, ναι, αποποινικοποιώντας όμως τα τη διαφθορά. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τις συνεχείς παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη ε, τα ειδικά τμήματα για τις ε, έρευνες ε, που ασκούν πιέσεις στους δικαστές και στους εισαγγελείς. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει η ρουμανική κυβέρνηση να σταματήσει να υποσκάπτει τις βασικές αξίες της Ένωσης. Αυτό πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα όλων μας. Επίσης, κυρία Ίνφελ, θα σας συμβούλευα να δείτε καλύτερα την απόφαση του ΕΛΚ στις 20 Μαρτίου από 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται οι παρατηρήσεις σας στην αλήθεια αυτής της δήλωσης. Κύριε Μποστινάρο, περιμένετε. Μου ζητήσατε διαδικαστικό. Θα είναι μόνο αυτό, όχι άλλο σχόλιο. Ε? Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποια πράγματα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΕΛΚ ίσως δεν ήσασταν παρόντες αλλά η απόφαση του Συμβουλίου να μην εκπροσωπείται εδώ είναι απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων. Ζητήστε από τους αρχηγούς των ομάδων σας ε, πώς λήφθηκε αυτή η απόφαση. Θα έπρεπε να αναφέρετε ένα άρθρο. Ε. Δεν ε, κάνετε αναφορά στον κανονισμό. Ο Μωρίς, Μωρίσα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η Ρουμανία είναι φιλοευρωπαϊκή χώρα. Ο ρουμανικός λαός έχει ασπαστεί τις ευρωπαϊκές αξίες, την ειρήνη, την ελευθερία, το κράτος δικαίου, την προηγούμενη διετία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών. Οι πολιτικοί έχουν υποχρέωση να ακούσουν τη φωνή του λαού. Οι πολιτικοί δεν επιτρέπεται να αλλάζουν τον νόμο προς ίδιων συμφέρον. Το ξαναλέω, εκατομμύρια ε, ε, Ρουμάνοι δεν θέλουν αμνηστία, δεν θέλουν συγχώρεση όλων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν η, η ρουμανική κυβέρνηση να προχωρήσει στις αποφάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ρουμανική κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τι λέει ο λαός. Ο πρόεδρος Ιωάννης στις 22 Μαΐου αποφάσισε δημοψήφισμα που θα δώσει την ευκαιρία στους Ρουμάνους να εκφράσουν την επιθυμία τους σε σχέση με το δικαστικό σύστημα. Μπορεί να πούνε όχι στην άφεση, στην αμνηστία, Μπορεί να πούνε όχι ε, στις ε, ε, αρνητικές τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα, ο οποίος πρέπει να αλλάξει λαμβάνοντας υπόψη την άποψη των δικαστών, των ειρηνοδικών και των εταίρων. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον ρουμανικό λαό στη μάχη που δίνει για τη δικαιοσύνη και τις ευρωπαϊκές αξίες. Πλέκαρτα από την κυρία Γκραπίν, τη δέχεστε. Μάλιστα. Αγαπητέ συνάδελφε, έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Είπατε ότι άλλαξαν εν μια νυχτή νόμοι. Ποιοι νόμοι? Εκτός από αυτόν που ανέφερε και ο Τσόλος. Ξέρετε κάποιο άλλο νόμο που να άλλαξε? Ευχαριστώ κυρία Γκραπίνη. Υπάρχει μια μακρά σειρά διαταγμάτων τα οποία έχουν εκδοθεί τον τελευταίο καιρό από αρχή, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2017, το 2013, την επόμενη μέρα εκατοντάδες χιλιάδες άτομα βγήκαν στους δρόμους ε, για να διαμαρτυρηθούν. Τελειώσατε? Ωραία. Περνάμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Κύριε Γιάροκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θέλω να μιλήσω εναντίον των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Ε, οι ίδιες κατηγορίες έχουν απευθεί και εναντίον της Ουγγαρίας. Παρ' όλα αυτά, η Ρουμανία έχει κάνει σημαντικότατη πρόοδο σε ό,τι αφορά την ένταξη των πιο φτωχών τμήματων του πληθυσμού. Ε, αντιθέτως, τα ε, ευρωπαϊκά κονδύλια φτάνουν πολύ καθυστερημένα και γι' αυτό το λόγο ε, θα πρέπει να συνεννοηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των Επιτρόπων και κυρία Κρέτσου, έτσι ώστε να φτάνουν χρήματα από τα διαχρονικά ταμεία έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι πολίτε τη Ευρωπαϊκής Ένωση που δεν λαμβάνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια αυτή τη στιγμή διότι υπάρχουν ε, γραφειοκρατικά προβλήματα. Και αυτό το λόγο ε, ε διώκονται από τις αιστείες τους η Επίτροπος κύριε Επίτροπε ε, είναι το δικό μας σχέδιο είναι ένα ευρωπαϊκό όραμα ο λαϊκισμός και η μικρές τοποθετήσεις ε, που αμφισβητούν το ευρωπαϊκό όραμα ε, έχουν ε, τις ρίες τους στην πραγματικότητα του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακριά από τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάμπει δια της απουσίας της. όταν βλέπουμε το τι έχει γίνει. Ε, απ' την άλλη μεριά, σε άλλα θέματα, ε, παρεμβαίνει στα εσω, εσωτερικές υποθέσεις ε, της χώρας. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει στις δικαστικές και συνταγματικές υποθέσεις χωρών. Ε, μας χρησιμοποιείτε ως ε, πιόνι για να κερδίσετε κάποιους ε, πόντους στις ευρωεκλογέ. Το ΚΑΤΣΔΙΑ είναι ε, ομιλίες ενός λεπτού. Παρακαλώ πολύ να το σεβαστείτε. Ο λόγο στον κύριο Γιούρεκ. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι, κυρία Επίτροπε. Υπόθηκε ότι αν η κατάσταση στη Ρουμανία δεν αλλάξει, τότε η Κομισιόν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Ευτυχώ η Επιτροπή αυτή δεν πρόκειται να λάβει πλέον κανένα μέτρο. Αρκετά μέτρα είδαμε από την Ευρωπαϊκή αυτή Επιτροπή μόνο εκλογικές κινήσεις μπορεί να κάνει τώρα. Ε, ρωτήσαμε γιατί δεν ήταν εδώ ο κύριος Τίμερμαντς. Πιστεύω ότι έχει συνηθίσει με εκλογικές κινήσεις τέτοιου είδους. Όσον αφορά τη Ρουμανία, η κατάσταση στη Ρουμανία είναι δύσκολη και περίπλοκη. Ε, το ίδιο όπως και στο Ηνωμένο Δεν καταλαβαίνω τι ανοχή έχει η κυβέρνηση και στη μικρή διαφθορά, γιατί η διαφθορά είναι ένα γενικευμένο κακό αλλά αυτό που δεν μου αρέσει επίσης είναι η εποπτεία των πολιτικών και των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα. Είναι πρόβλημα, αλλά οι Ρουμάνοι πρέπει να το λύσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Νικολάη, η σειρά σας. Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή για το κράτος δικαίου, βασικό θεσμό της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν προκαλείται μια τέτοια συζήτηση και δεν ε, παρίσταστε εδώ, είτε είναι ότι περιφρονείτε τη συζήτηση ή περιφρονείτε τους πολιτικούς που συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Δεν είναι σωστή αυτή η συζήτηση και φιλότιμη ε, μας ε, προσβάλλει εδώ σε αυτό το ημικύκλιο, μας προσβάλλει από αυτούς που δεν συμμετέχουν έχει κανείς την εντύπωση ότι παίζει σε μια ταινία με κάποιον που καταδικάζεται για αυτά που σκέφτεται. Αυτό που θα κάνατε, αν είχατε ε, ένα ελάχιστο αξιοπρέπεια, ε, θα πηγαίνετε να δείτε τι έχει γίνει στη Ρουμανία. Δεν έχουμε υιοθετήσει καμία νομοθεσία και όμως μας επικρίνουν γι' αυτό. Αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι να μαζέψετε ψήφου ε, όσοι θέλουν να μείνουν στην εξουσία, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αυτού του είδου συμπεριφορά απομακρύνει του πολίτε από την Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παρατήσετε το λαϊκισμό που βλέπουμε σήμερα. Ολοκληρώθηκαν εδώ. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το Κατζιάι. Όλοι θα μιλήσετε, κυρία Βαΐ. Ευχαριστώ πολύ. Για να απαντήσω στην Επίτροπο Γιούροβα, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε του Ιστφαν Μπέκε και έναν άλλον Ρουμάνο ε, που αντιμετωπίζει ποινική δίωξη. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα. Η πολιτική ασκεί πιέσεις στην ποινική δικαιοσύνη και ξαναζούμε ε, τις ε, πιο δύσκολες εποχές του, του όπου τους αντιπάλους οι πολιτικοί τους αντιμετώπιζαν με φυλάκιση και με ποινικέ διώξεις για να επιτύχουν τους πολιτικούς τους στόχους. Έχουμε δύο πολίτες εδώ που αντιμετωπίζουν ποινικέ διώξεις ενώ το μόνο που έκαναν ήταν να δώσουν μάχη για τα ε, δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στη Ρουμανία. Τα γνωρίζετε αυτά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ο κύριος Πόπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Και πάλι δεν πρόκειται για συζήτηση, πρόκειται για μια φιέστα προεκλογική. Όπως άλλωστε ήταν και ο σκοπός αυτών που άρχισαν τη συζήτηση. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο, δεν υπάρχει ουσία. Δεν θέλουμε να μπούμε σε ε, ουσιαστικές λεπτομέρειες. Κανείς δεν θέλει να γίνει συγκεκριμένος. Μιλάμε γενικά για φόβους, ανησυχίες, κινδύνους. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να ανησυχούμε. Πρέπει να μιλάμε για κινδύνους. Όταν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το Στρασβούργο υπαγορεύουν στους ε, Ρουμάνους δικαστές τι πρέπει να κάνουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το κράτος δικαίου σημαίνει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν επιτρέπεται να υπαγορεύεται όποιοι κι αν είστε ε, τι θα, στη δικαιοσύνη τι θα κάνει. Κυρία Ταπεντέν. Κυρία, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Θα αρχίσω με μία ερώτηση. Μιλάμε για το κράτος δικαίου. Εννοούμε βέβαια και σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε στη Ρουμανία. Θέλουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης που θα είναι δίκαιο, που θα σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών, όπου δεν θα υπάρχουν καταχρήσεις από τους εισαγγελείς, ε, η ζωή και η σταδιοδρομία των ανθρώπων δεν θα καταστρέφονται. Το μήνυμα μου προς όλους τους ε, βουλευτές ε, που χρησιμοποιούν σλόγγαν τη Ρουμανία στην προεκλογική τους εκστρατεία είναι «Έχετε εκλεγεί γιατί είστε αξιόπιστοι στα μάτια των ψηφοφόρων». Δεν επιτρέπεται τώρα να γίνει μια συζήτηση ακόμη η οποία ε, επιτίθεται σε ένα κράτος μέλος. Αυτό ε, εισάγει διπλά μέτρα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εδώ θέλετε να αποκομίσετε ωφέλη, αλλά αυτό υποσκάπτει το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος ε, Τζάκον. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να καταλάβω πώς μπορούμε να μιλάμε για ένα θέμα, το κράτος δικαίου, όταν αυτό δεν ορίζεται συγκεκριμένα. Στο βαθμό που η ποινική δικαιοσύνη αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών, δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε ε, μια απόφαση. Γι' αυτό απλώς θορυβούμε θορυβούμε εδώ μέσα και τίποτε περισσότερο. Πρόκειται για μια εθνική αρμοδιότητα της Ρουμανίας και βεβαίως το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ρουμανική Δικαιοσύνη θα λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές αξίες και τους κανόνες, αλλά ε, πέραν αυτού πρέπει να πω ότι δυστυχώς δεν έχουμε κράτος δικαίου, ε, χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσουμε εκεί. Περιμένω όμως από το επόμενο κοινοβούλιο να ορίσει το κράτος δικαίου και να το θέσει σε εφαρμογή. Κυρία Πρόεδρε, συναδελφοί, κυρία Επίτροπε, η ε, Ρουμανία είναι η χώρα μου και ποτέ δεν θα επιτρέψω να κυκλοφορούν ψεύδι ε, σε βάρος της. Υπάρχει κράτος δικαίου στη Ρουμανία. Το λέω και το τονίζω. Κάποια ρουμανικά πολιτικά κόμματα προσπαθούν να παρουσιάσουν στον ε, δημόσιο χώρο μια τελείως διαφορετική εικόνα. Για αυτό ωφελεί την αντιπολίτευση, κάποια ευρωπαϊκά κόμματα και γι' αυτό ε, ε, διαστρεβλώνεται τελείως η εικόνα της ε, δικαιοσύνης στη Ρουμανία. Εκείνοι που κατηγορούν είναι οι ίδιοι που ασκούν πιέσεις στη δικαιοσύνη στην χώρα μου προσπαθώντας να επιβάλλουν καταδίκες, ποινές, ακόμα και λήψη αποδεικτικών στοιχείων και ασκούν πιέσεις στους δικαστές για να αθωώσουν κάποιους δικούς τους. Όταν τα μέλη της Ρουμανικής Αντιπολίτευσης εντοπίσει κάποια αμφιλεγόμενα θέματα από νομικής άποψης ε, σταματούν ε, να ασκούν πιέσεις. Αυτό που βλέπετε σήμερα διακοπή. Εγώ ήμουν υπέρ της ε, ένταξης της Ρουμανίας ε, δεν ήθελα να μείνει στην άκρη η Ρουμανία και να υπάρχει δικαιοστάσιο. Ήμουν ε, μεταξύ εκείνων που ε, καταπολέμησα τη διαφθορά, την εκμετάλλευση των παιδιών. Μετά από 15 χρόνια βλέπω ότι η Ρουμανία ασκεί την Προεδρία, δεν μπήκε στον κόπο να έρθει εδώ και έχει δημιουργήσει ε, ε, ε, εγκληματική οργάνωση η οποία αποσπά ενωσιακά κονδύλια. Θα πρέπει να μην διστάσουμε να καταγγείλουμε αυτά που γίνονται στη Ρουμανία. Όπως είπε και η Επίτροπος Γιούροβα, πρόκειται για το κράτος δικαίου στην Ένωση, όχι μόνο στην Ρουμανία εδώ. Θέλουμε να στηρίξουμε τους ε, ε, ε, αθώους Ρουμάνους πολίτες που αψήφισαν κινδύνους κρύο για να διαδηλώσουν υπέρ του κράτους δικαίου. Ο κ. Λόπεθ κύριε Επιτροπέ, ως σοσιαλιστής παρεμβαίνω. δεν μιλώ ούτε στα ουγγρικά ούτε στα ρουμανικά ε, σε, σεβόμενος την παρουσία αυτών των χωρών. ο, η συζήτηση για το κράτος δικαίου πολύ συχνά καταλήγει να γίνεται ε, διαξυφισμός κατηγοριών. Ε, στο άρθρο, από το άρθρο, στο άρθρο 7 εντάχθηκαν διάφορες χώρες όπως γνωρίζετε και δεν θέλω αυτές οι χώρες ε, να ανταλλάσσουν κατηγορίες με τις υπόλοιπες. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το βασικό είναι ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μπροστά μα. Ε, χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο μηχανισμό επαλήθευση ε, του κατά πόσον πληρούνται οι αρχέ του άρθρου 12 της Συνθήκη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτο δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, ποιότητα τη δημοκρατία και καταπολέμηση τη διαφθορά. Αυτό ο μηχανισμό κυρία Γιουρόβα, είναι κάτι το οποίο απαιτούμε εδώ και καιρό από την Κομισιόν, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν θα πρέπει στην επόμενη θητεία να υποβάλει προτάσεις για ένα τέτοιο μηχανισμό. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Γιουροβά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να εκφράσω την πεποίθηση ότι εκπροσωπώ όλη την Κομισιόν, το σύνολο του οργάνου. Αυτό για όσους επικρίνουν την απουσία του κ. Τίμερμανς, του πρώτου αντιπρόεδρου. Ο κ. Τίμερμανς ε, προσπαθεί εντατικά να διατηρήσει ανοιχτό τον πολιτικό διάλογο με τη ρουμανική κυβέρνηση και είναι ο τελευταίος ο οποίος θα πρέπει να επικριθεί για οτιδήποτε έχει κάνει για οποιαδήποτε παράληψή του. Δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι το εξή. Η Κομισιόν δεν παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις. Αυτό το αναφέρω στην κυρία Γκραπίνη. Αυτή είναι η αρχή μας. Δεν παρεμβαίνουμε. Εξετάζουμε μόνο συστημικά προβλήματα που προκύπτουν από την ομοθεσία της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αναφερθεί στις πρόσφατες ε, ε, μεταρρυθμίσεις που έγιναν στο δικαστικό σύστημα στη Ρουμανία. Γιατί το συνολικό αθρηστικό αποτέλεσμα όλων αυτών των αργών μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση του κράτους δικαίου στη Ρουμανία. Τελευταίο μου σχόλιο. Κυρία Μοργκάη, όχι, δεν γνωρίζω αυτές τις δύο περιπτώσεις, Μπέκε και Σουίτς. Θυμάμαι μου στη δική μου περίπτωση, τη δική μου υπόθεση από το 2006. Εγώ κατηγορήθηκα για διαφθορά το 2006. Στο πλαίσιο μιας πολύ βρώμικης υπόθεσης ε, που έγινε με μοναδικό γνώμονα πολιτικά συμφέροντα και αμαυρώθηκε η εικόνα μου στα μέσα ενημέρωσης και θυμάμαι τον εαυτό μου. Ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν πίστευα ότι, δεν πίστεψα ότι κάποιος δικαστής θα με έστελνε στη φυλακή πίστευα στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη στη χώρα μου. Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι η υπόθεση δεν έφτασε καν στα δικαστήρια ποτέ. Ήτανε απλώς λάσπη. Το θυμάμαι πολύ καλά όμως. Και είναι παράδοξο το ότι η Ρουμανία μου προσέφερε δουλειά μετά από αυτό. Γιατί όλα είχαν καταστραφεί όλη μου η καριέρα μέχρι η οικογένειά μου είχε καταστραφεί. Δούλεψα στη Ρουμανία. Η Ρουμανία μου έδωσε μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τη γνώση μου, να την προσφέρω και γι' αυτό είμαι ο, ο τελευταίος άνθρωπος που θα πρέπει να κατηγορηθεί ότι φέρεται κατά της Ρουμανίας. Στην Ρουμανία μπορεί να φτάσουμε στην κατάθεση στάση μη αναστρέψιμων αλλαγών του δικαστικού συστήματος με συστημικές παραβάσεις του κράτους δικαίου της ε, ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του δικαστικού συστήματος. Αυτοί, αυτές κινδυνεύουν. Πολύ στενά παρακολουθώ το τι κάνει η Ρουμανία μέσω του μηχανισμού CVM. Ε, και ανησυχώ για τις αλλαγές που ξεκίνησαν ξαφνικά προς λάθος κατεύθυνση ενώ όλα πήγαιναν προς τη σωστή κατεύθυνση πριν. Η, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι σημαντικός πυλώνας του δημοκρατικού καθεστώτος του δημοκρατικού συστήματος και έχει αναπτυχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι μια αργή προοδευτική διαδικασία που οδηγεί σε ένα ισορροπημένο συνταγματικό σύστημα. Ο δικαστικός πυλώνας είναι βασικό κομμάτι αυτού. Μπορεί όμως να καταστραφεί. Εν μία νυχτή, πραγματικά εν μία νυχτή. Και αυτό θέλει να αποφύγει η Κομισιόν στη Ρουμανία. Οπότε ο διάλογος συνεχίζεται. Θα συμφωνήσω με αυτούς και αυτές που είπαν ότι οι Ρουμάνοι και οι Ρουμάνες αξίζουν περισσότερα, θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Οι συζητήσει γίνονται σε τεχνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Θα ζητήσω να επιστρέψει σε πολιτικό επίπεδο ο διάλογος και να είναι θετικός, επικοδομητικός, να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές και στην επάνωδο των μεταρρυθμίσεων στη σωστή άκουσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παβέλ. Δεν σας δίνω το λόγο. Ήρθατε τελευταία στιγμή. Δεν ζητήσατε μπλε κάρτα. Δεν μπορείτε να θέσετε μπλε κάρτα για την κυρία Γιούροβα. Εάν λοιπόν δεν έχετε κάτι διαδικαστικό με κάποιον αριθμό και μην μιλάτε και σε, χωρίς μικρόφωνο, δεν έχει νόημα. Ζητώ συγγνώμη. Έπρεπε να είχατε έρθει λίγο νωρίτερα για να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση η οποία έχει ολοκληρωθεί. Αλλάζουμε θέμα στην ημερήσια διάταξη αλλά προβλέπετε να αλλάξουμε επίτροπο και θα μιλήσουμε ε, για ε, τα για τα συλλογικά επενδυτικά ε, κεφάλαια, την εκθέση του κυρίου Κλίντσα. Ε, το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Κλίντς δεν είναι εδώ. Οπότε θα στραφώ στον κύριο Ντομπρόφσκης, ο οποίος δεν με ακούει αυτή τη στιγμή και θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Ντομπρόφσκης, ευχαριστώ. Madam Chair, uh, honorable members. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέρη, τα επενδυτικά ταμεία προσφέρουν ευκαιρίε ε, στου Ευρωπαίου πολίτε να κάνουν οικονομίε για το μέλλον του. Είναι σημαντικό εργαλείο για την διοχέτευση των αποταμιεύσεων στην οικονομία και για την αύξηση τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών εταιριών. Σήμερα όμω οι αγορέ επενδυτικών κεφαλαίων είναι εθνικέ. Για παράδειγμα, 70% των επενδυτικών τίτλων πολλούνται σε εγχώριε αγορέ ε, το μερίδιο τίτλων που πολλούνται σε τρίτες χώρες ε, είναι 35% πολύ μικρό και για εναλλακτικά, μία, για εναλλακτικά κονδύλια είναι ακόμα μικρότερο, περίπου 7%. Αυτό οφείλεται κυρίως στα ρυθμιστικά εμπόδια, στα διασυνεροϊκά ε, εμπόδια. Ω μέρο τη Ένωση κεφαλαίου προτείνει η Κομισιόν μέτρα άρση των εμποδίων για να βελτιωθεί η λειτουργία τη ενιαία αγορά για τα επενδυτικά κεφάλαια. Στόχο μα είναι οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να πουλήσει επενδυτικά προϊόντα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, να ε, υπονομεύεται η προστασία των επενδυτών. Το προτείνουμε να γίνει με τη μείωση των εμποδίων και προτείνοντας λύσεις ε, στους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή και όλους τους συνεισηγητές για τις προσπάθειες που έκαναν να προωθηθεί γρήγορα το θέμα και θα ήθελα επίσης να συγχαρώ και εσάς κύριε Τομπρόφσκης να σας διακόψω ένα λεπτό. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, διερμηνίας, κυρία είναι αν έχετε πρόβλημα διερμηνίας σε ποια γλώσσα. Όχι. Το κανάλι στα αγγλικά δεν ακούγεται στα αγγλικά, ακούγεται σε κάποια άλλη γλώσσα. Και δεν καταλαβαίνω. Α, πρόβλημα είναι αυτό, λέει ο Πρόεδρος. Πράγματι, ε, προσπαθήσουμε να ξαναβάλουμε στα σωστά κανάλια τις σωστές γλώσσες. Μπορείτε να πείτε αν τώρα λειτουργεί, μπορείτε να ακούσετε, να μας πείτε αν ακούτε αγγλικά από τα αγγλικά. Κύριε Ντομπρόσκης, μπορείτε να συνεχίσετε. Λοιπόν, για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας συγχαρώ επειδή γρήγορα επιτύχατε μια πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο στις ε, τριμερείς διαπραγματεύσεις η Κομισιόν υποστηρίζει τη συμφωνία η οποία βρίσκει ισορροπία μεταξύ της διευκόλυνσης της διασυνοριακής ε, κατανομής των ε, συλλογικών επενδύσεων και τη διασφάλιση ε, της προστασίας των επενδύσεων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να δώσουν τη δυνατότητα σε διαχειριστές να, μπορούν να προωθήσουν σε πιθανούς επενδυτές τα κονδυλιά τους χωρίς να συμμορφώνται με όλους τους κανόνες. Ταυτόχρονα οι συνομοθέτες έχουν εισάγει εχέγγυα ώστε να προστατεύονται ε, κάποιες από αυτές τις πρακτικές και να αποφεύγεται η παρακάμψη των ευρωπαϊκών κανόνων. Οπότε αύριο πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτός αυτή η σημαντική συνιστόσα της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Λαμασούρ εκ μέρους του ΕΛΚΙ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ήθελα να ευχαριστήσω τη διαπραγματευτική ομάδα υπό την αιγίδα του εισηγητή μας του κύριου Κλίντσα, ο οποίος θα έρθει σε λίγο, για το αποτέλεσμα που είχαμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Αύριο θα ψηφίσουμε ένα κείμενο σημαντικό για την ολοκλήρωση της ε, Ένωσης Κεφαλαίου Αγοράς. Όπως υπενθύμησε ο κύριος Πρόφσκης, η απερχόμενη Κομισιόν ε, την οποία συγχαίρω για τις προσπάθειές της, ε, έδωσε μια απάντηση στοχευμένη και ακριβή για τα ε, διασυνοριακά εμπόδια που υπήρχουν εντός της Ένωσης. Η συμφωνία που επιτεύχθη με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των δια... διοργανικών διαπραγματεύσεων φαίνεται ικανοποιητική και ισόρροπη. Λαμβάνει υπόψη τα περισσότερα ζητήματα που έθεσε το Κοινοβούλιο και προτείνει κυρίως η διαδικασία αποτιτλοποίησης των ε, κονδυλίων να γίνει πιο λογική ε, καταργώντας τα κατόφλια τα οποία ήταν ε, αυθαίρετα. Ο μηχανισμός διευρύνθηκε στα προϋπάρχοντα επενδυτικά μέσα και εξορθολογίστηκε η όλη διαδικασία. Έτσι το εργαλείο θα είναι πιο προσαρμοσμένο στους στόχους που επιδιώκουμε στο σύνολο καταφέραμε να διατηρήσουμε τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε να αποφύγουμε αυτές τις νέες ευκαιρίες να οδηγήσουν σε πιθανές παραβιάσεις και παρακάμψεις κυρίως από φορείς τρίτων χωρών. Τέλος, με την ιδέα της ευρωπαϊκής εποπτείας σε, υπό τη μορφή μιας ευρωπαϊκής αρχής παρότι να με αυτή η ιδέα χαίρομαι που ο συμβιβασμός που ανταποκρίνεται στις απαιτήσει του Κοινοβουλίου παρέχει με καλύτερο ρόλο στην ε, Ευρωπαϊκή Αρχή ε, εποπτείας κεφαλαιόρων. Αυτό θα είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της δικής μας Ένωσης Κεφαλαιογορών. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Ντελβό εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την ομάδα αλλά κυρίως τον εισηγητή τον κύριο Κλίντς που ήταν πολύ αποτελεσματικό στον τριμερή διάλογο, κάτι που μας επέτρεψε να κλείσουμε το θέμα πριν το τέλος της θητείας μας. Η νομοθεσία αυτή έχει ως στόχο να επιτρέψει την πιο εύκολη και διασυνοριακή διανομή ε, συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων. Αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία της διάθεσης γίνεται σε, ε, σε αγορέ αγορές μόνο και πολλοί διστάζουν να μπουν σε μια καινούρια διαφορετική αγορά, ε, κάτι που επηρεάζει τα συμφέροντα των ε, επενδυτών. Χρειαζόμαστε αυτή τη διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσουμε τις οικονομίες μας. Θέλουμε λοιπόν να άρουμε τα εμπόδια και να μπορέσουμε να ε, διευκολύνουμε για παράδειγμα τις δραστηριότητες πρώτης διάθεσης στην αγορά και άλλες ε, ρυθμίσεις. Ε, θα πρέπει ε, να ενημερώνεται οι εποπτικές αρχές έτσι ώστε να μπορούν να τελούν τα καθήκοντά τους. Ε, και να υπάρχει μια πραγματική ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα ε, στους, ε, στις, στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και στην αρχή αυτή, όπως επίσης, στις αρχές αυτές, όπως επίσης και στην, με την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Κινητών Αξιών. Ένας διαχειριστής θα πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις ενημέρωση επίσης και σε ό,τι αφορά τους επενδυτές, ακόμα και όταν αυτοί έχουν φύγει από τη χώρα. Τέλος, ε, θα ήθελα να μιλήσω για την PRIPS. Ε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δώσουμε ε, μία παράταση δύο ε, ετών για τους ΟΣΕΚΑ. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα επιταχύνει τις εργασίες της έτσι ώστε αυτή η παράταση να μην χρειαστεί να διαρκέσει δύο έτη αλλά λιγότερο, όσο δυνατό λιγότερο. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Μαριά. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κεφαλαίου αγοράς πραγματικά είναι αναγκαιότητα, ιδίως σε μια φάση όπου το ίδιο το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ε, ρευστότητα η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό η... τα συλλογικά επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και μάλιστα συγκεντρώνουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ ταυτόχρονα όμως πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά τα κεφάλαια δεν κατευθύνονται στην πραγματική οικονομία. επί του πρακτέου αποτελούν μέρος και λειτουργία αυτού που ονομάζουμε οικονομία καζίνο. γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει ένας επιπλέον έλεγχος τόσο φυσικά διευκόλυνση σε επίπεδο διασυνοριακή αλλά ταυτόχρονα οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να βλέπουν ότι αυτά τα κεφάλαια πραγματικά επενδύονται στην πραγματική οικονομία και προστατεύονται οι ίδιοι επενδυτές. ευχαριστώ. Euh, η ρύθμιση αυτή για την απλοποίηση της διασυνοριακής διανομής των επενδυτικών συλλογικών κεφαλαίων είναι σημαντικό βήμα για την απάλληψη εμποδίων στην εσωτερική αγορά, προωθούν την επικοινωνία, τη διαφάνεια, οδηγούν σε πιο ολοκληρωμένη αγορά. Η αύξηση του ανταγωνισμού επιτρέπει στους παρέχοντες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να αυξήσουν και να διευρύνουν την προσφορά. Οι επενδυτές έχουν περισσότερες δυνατότητες και δημιουργούνται έτσι περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ κυρίως. Ε, εγώ το λέω όχι μόνο από άποψη ε, οικονομίας αλλά και από την άποψη της ανάπτυξης. Ε, πιστεύω ότι ε, το μέτρο αυτό είναι υποχρεωτικό διότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευημερία. καλό είναι να υποστηρίξουμε το μέτρο αυτό που στοχεύει σε μεγαλύτερη συνεργασία και ε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί και για την αύξηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ε, ε, αγορές κεφαλαίων. Και εκεί υπάρχει δυνατότητα απλούστευσης η οποία βλέπουμε να διευκολύνεται εδώ. Και έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον ρόλο των ενδιάμεσων. Ευχαριστώ. Κυρία Νίνα Γκίλ. Ε, ένα λεπτό. Καταρχήν, ε, εκφράζω τη θλίψη μου για την πυρκαγιά στην, στον καθεδρικό της Νότρου Γιατί είναι, πολύ θλιβερό αυτό. Ε, η έκθεση αυτή αποσκοπεί στην κατάργηση εμποδίων. Ε, από τα τρισεκατομμύρια επενδύσεων, 70% όλων των περιουσιακών στοιχείων ε, διακρατούνται ε, από ε, μία ε, τα οποία λειτουργούν στις εσωτερικές αγορές. Μόνο 37% διατίθενται από, σε τρία κράτη-μέλη από διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. αυτό λοιπόν το πρόγραμμα επιτέλους θα μειώσει κάποια εμπόδια, θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα ε, αντικαταστήσει κάποιους ε, ε, πολύ δυσκίνητους εθνικούς κανόνες. Πιστεύω ότι αυτό είναι κρίσιμο βήμα. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε πάρα πολλές χώρες, από Πορτογαλία μέχρι Λετωνία. Ερωτώ λοιπόν τον Αντιπροδιακόπη, υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί η διαφάνεια και να υπάρχει τυποποίηση σε ό,τι αφορά τη θέση ανωτά των ορίων στα τέλη, χρέος, που χρεώνονται. Ε, κυρία είναι Ε, χρειάζονται ε, κεφάλαια κινδύνου και ε, κεφάλαια επενδυτικά στην Ευρώπη. Όπως είπε η συνάδελφος Νίνα ε, Τζιλ, ε, τώρα σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή τις ασιατικές χώρες η θέση της Ευρώπης ε, υπολείπεται γιατί τα κράτη-μέλη θέτουν διαφορετικούς κανόνες, ε, είναι διαφορετική η δομή του κόστους, η ρύθμιση της αγοράς δεν είναι σαφής και αυτό είναι αποθαρρυντικό για τους επενδυτές. Χαιρετίζω λοιπόν αυτό το νομοθέτημα, το οποίο ελπίζομαι ότι ε, θα θέσει σαφέστερους κανόνες για το, το marketing, ε, τις διαδικασίες πριν από την εμπορική προώθηση, το marketing κλπ. Το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι ε, μια εποπτεία ε, πλήρως ευρωπαϊκή και μεγαλύτερη διαφάνεια εις ό,τι αφορά τις δομές ε, του κόστους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κομπέρν είχε εγγραφεί για τέσσερα λεπτά, αλλά δεν είναι εδώ και δεν είχε εγγραφεί κανείς για το ΚΑΤΣΔΙΑΙ, οπότε επιστρέφουμε σε εσά κύριε Ντομπρόφσκης για να κλείσουμε τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κλίντς και τους χειώδεις εισηγητέ για τη δέσμευση που ανέλαβαν. Ε, αναμένω ε, με ενδιαφέρον την αυριανή ψηφοφορία. Περίπου 440 εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομηθούν για τους διαχειριστές ε, ε, κεφαλαίων ε, χάρη στα μέτρα μας. Ε, θα βελτιωθεί ο ανταγωνισμός και θα υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικέ επιλογές σε χαμηλότερο κόστος για τους επενδυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Περνάμε στο επόμενο σημείο, ή μάλλον ήμουν έτοιμη να περάσουμε στο επόμενο σημείο, αλλά δεν έχω τον κατάλογο των ε, αγορητών, οι οποίοι βρίσκονται καθοδόν. Θα ζητήσω λοιπόν για λίγα λεπτά την υπομονή σας μέχρι να έρθουν στην αίθουσα. Κυρία Πιετικάνε, ναι, είχα δει τον κύριο Εκμάρκα. Ναι. Αλλά περίμενα να έρθουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, περνάμε στην κοινή συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα. Η συζήτηση είναι ο κύριος Πέτερ Σίμων για την τροποποίηση που αφορά τις απαιτήσει για τα ίδια κεφάλαια, τις κεφαλαίκες απαιτήσει, ε, την έκθεση του κ. Χαϊκμάρ και ικανότητα απορροφή ζημιών και ανακεφαλαιοποίηση των πιστοτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων και μετά η οδηγία που σχετίζεται με αυτή ε, το θέμα πάλι του κ. Χαϊκμάρκ για την ικανότητα απορρόφηση των ζημιών και ανακεφαλαιοποίηση των πιστοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τροποποίηση τη οδηγία. Ξεκινάμε λοιπόν με ε, το να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ζήμων. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική συνεργασία που διήρκεσε δυόμιση χρόνια και χαρακτηρίστηκε από εξισορρόπηση συμφερόντων ε, και συγκερασμό διαφορετικών απόψεων σχετικά με το πώς θα κάνουμε ασφαλέστερη την Ευρώπη. Μετά την τραπεζική κρίση του 2008 που στήχησε 200 δις τους Ευρωπαίους ε, φορολογουμένους, πώς μπορούμε να ε, σώσουμε τους, ε, τους πολίτες μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές, ε, Κάρας Κόξε και τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Αντιπροέδρου Ντομπρόφσκης. Ευτυχώς η Κομισιόν σε δύσκολες διαπραγματεύσεις, σε δύσκολες εποχές ε, ανταποκρίθηκε, ήταν στη διάθεσή μας ε, επί 24 ώρου βάσεως, ούτω ώστε να έχουμε υποστήριξη στις συμβιβαστικέ λύσεις. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Ε, στην τραπεζική εποπτεία έχουμε ακολουθήσει την Επιτροπή της Βασιλείας. Ε, ε, έχουμε εισαγάγει έναν δίκτυ μόχλευσης, περιορισμό του χρέου των τραπεζών ε, και κατοχύρωση κατώτατου ορίου ιδίων πόρων. Επίσης, θέσαμε όρια για τις τράπεζες που είναι συστημικά πολύ σημαντικές παγκοσμίως. Εισαγάγαμε ένα ε, ε, ποσοστό ε, ρευστότητας. Στις μεγάλες τράπεζες θα πρέπει να προβλέπεται διαδικασία ανάκαμψης. Αυτό που με απασχόλησε πάρα πολύ είναι ότι παρεκκλίναμε για πρώτη φορά στου κανόνες που εισαγάγαμε ως πρώτη αντίδραση μετά την κρίση. Τώρα πήραμε ε, μια απόσταση και μπορέσαμε να δούμε καλύτερα το μέλλον με προσανατολισμό πιο μακροπρόθεσμο. δημιουργούμε ε, ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες στην Ευρώπη. Όχι όμως με ίδιους κανόνες για όλους, αλλά με διαφοροποιημένη προσέγγιση. Αυτό δεν το κάναμε στο παρελθόν δεν λάβαμε υπόψη μας ότι οι μικρές τράπεζες χαμηλού κινδύνου πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ότι οι μεγάλες διεθνώς συστημικά σημαντικές τράπεζες. Πρέπει να, διαπιστ... να, να, να ε, τις ελευθερώσουμε από την γραφειοκρατία και να μην τους επιβάλλουμε κι άλλους γραφειοκρατικούς όρους. Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους διότι για πρώτη φορά καταφέραμε να ε, προστατεύσουμε τις μικρότερες τράπεζες κάτω από 5 δις που αποδεδειγμένα δεν ε, ενέχουν μεγάλους κινδύνους. Άρα δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται γραφειοκρατικά. Ε, σήμερα μπορούμε να αποφύγουμε την υπερβολική γραφειοκρατία και ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, μελλοντικές συγχωνεύσεις μικρών τραπεζών με πιο ευέλικτο τρόπο. Επίσης, ε, δημιουργήσαμε ένα ενιαίο σύστημα κοινοποιήσεων, το οποίο είναι αξιόπιστο και δίνει στοιχεία σχετικά με τράπεζες και τις κινήσεις τους. Ε, στο παρελθόν, η δια η, ε, παρακολούθηση ε, όλων αυτών των στοιχείων ε, επιβάρυνε πάρα πολύ τις υπόλοιπες τραπεζικές εργασίες και ε, δεν ακολουθούσε η διαδικασία αυτή μία ομαλή ροή. Αυτό τώρα εξασφαλίζεται. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε μακρές συνεδριάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν στο Κοινοβούλιο και επίσης και τους συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χακμάρκ. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους συναδέλφους τους και όσοι ηγητές στην Κομισιόν και το Συμβούλιο για την ε, εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Η... Εξαιτία τραπεζικής κρίσης ε, δημιουργήθηκαν τρία νομικά κείμενα. Η ιεραρχία στην οποία αποφασίσαμε ένα χρόνο πριν ήταν, ε, έφερνε αυτά τα δύο κείμενα στην, στη βάση της, τα κείμενα που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ε, έχει σχέση το θέμα αυτό με τον μηχανισμό εξυγείας των τραπεζών που υιοθετήθηκε. Βασικός στόχος ήταν να αλλάξουμε την λογική του τραπεζικού τομέα, να διευκρινίσουμε ότι όσοι έχουν τράπεζες στο χαρτοφυλάκιό τους ή επενδύουν σε τράπεζες έχουν και την ευθύνη να καλύψουν τις ενδεχόμενες ζημιές μαζί με, το θέμα, μαζί με τα εργαλεία που είχαμε με τις ε, ε, ε τραπεζών και λοιπά ε, δημιουργούμε ένα σύστημα έτσι ώστε αυτοί που επενδύουν σε τράπεζες να ξέρουν ότι μπορεί να χάσουν τα λεφτά τους. Αυτό χρειάζεται προκειμένου να πετύχουμε δύο στόχους. Πρώτον, να διευκρινίσουμε σε όλους ότι οι επενδύσεις σε τράπεζες εγκυμονούν κάποιους κινδύνους. Δεύτερον, ε, η συμφωνία του Βερολίνου θα πρέπει να εφαρμοστεί με ένα προβλέψιμο τρόπο. Και το δικό μου, ε, κατά τη δική μου άποψη ήταν σημαντικό να εξασφαλίσουμε ακριβώς ότι η εισαγωγή του τίλακ δεν είναι ένας τρόπος για να παρακάμψουμε την την ε, ε, ανάγκη οι επενδυτές σε τράπεζες να καλύπτουν και τις ζημίες. Το γνωστό bail-in. Οπότε έχουμε καλύτερους κανόνες για την εφαρμογή του TILAC με αυτό το νομικό κείμενο. Έχει τεθεί ένα ε, ανώτατο όριο ε, που σημαίνει ότι δεν καθορίζουμε υπερβολικά ψηλά ίδια κεφάλαια για τις ε, τράπεζες, αλλά από την άλλη μεριά επαρκεί. Αυτό το πετύχαμε. Ποτέ δεν είχαμε καλύτερη ευκαιρία να εξηγιάνουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις ε, τράπεζες σε δύσκολες στιγμές. Η εξηγένση θα γίνει πιο εύκολη και ταυτόχρονα οι αγορές θα είναι πιο έτοιμες να αποφύγουν να μπουν οι τράπεζες σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Διότι οι επενδυτές που επενδύουν σε τράπεζες ξέρουν πια ότι κάτι διακινδυνεύουν. Και θα έχουμε πάρα πολλές εγγυήσεις έτσι ώστε ε, να υφίστανται τα κατάλληλα κεφάλαια και τα κατάλληλα MREL, οι ελάχιστε απαιτήσει δύο κεφαλαίων. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές και την Κομισιόν. Έχουμε ένα πολύ καλό θεμέλιο για την Τραπεζική Ένωση, αλλά και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Ευχαριστώ. Το τραπεζικό πακέτο υιοθετήθηκε από την Κομισιόν πριν από δυόμιση περίπου χρόνια, το Νοέμβριο του 2016 συγκεκριμένα. Ε, βασιζόμαστε σε υπάρχοντες ε, τραπεζικούς κανόνες προκειμένου να ρυθμίσουμε την υγιεινή κατάσταση που προέκυψε μετά την κρίση με μείωση των κινδύνων αλλά και προκειμένου να συμμορφωθούμε τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Εφαρμογή διεθνών προτύπων, ενώ ταυτόχρονα οι τράπεζες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την πραγματική οικονομία. Το Συμβούλιο το Μάιο του 2018 κατέληξε σε κοινή θέση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιόνιο του ίδιου χρόνου ε, εξέφρασε τη δική του γνώμη. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις για την προσήλωσή τους και για την αποφασιστικότητά τους τον κύριο Ζήμων ιδιαίτερος και τον κύριο Χόκμαρκ. Οι προσπάθειές σας ήταν ε, πολύ αξιόλογες. Τα κείμενα αυτά, ε, μάλλον το Κοινοβούλιο βελτιώνει τις αρχικές προτάσεις της ε, Κομισιόν. Ε, ιδιαίτερα σε θέματα τη της παράνομων εσόδων κλπ. Ε, περιλαμβάνονται μέτρα τα οποία θα αυξήσουν την ε, σταθερότητα των τραπεζών, για παράδειγμα το ποσοστό μόχλευσης, το δίκτυο μόχλευσης και μέτρα έτσι ώστε οι τράπεζες να μην εξαρτώνται από ε, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και καταθέσεις. Ενισχύουμε την εποπτεία από τις εποπτικές αρχές και την κάνουμε πιο ευέλικτη. Επίσης έχουμε περισσότερα εργαλεία για την εξηγένση των τραπεζών, ιδιαίτερα μεταγράφουμε το διεθνές πρότυπο για την απορρόφηση των ζημιών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα ελάχιστο ποσοστό ελάχιστο ε, δίκτυο MREL, ελάχιστον απαιτήσεων ιδιών κεφαλαίων και θα διασφαλίσουμε έτσι ότι οι τράπεζες έχουν επαρκές μαξιλαράκι έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την εξογίανσή τους χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση ε, με κρατικά ε, κονδύλια. Ταυτόχρονα το πακέτο δίνει σημασία σε διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την, οικονομία, με την ε, χρηματοδότηση πραγματικής οικονομίας. Ε, για παράδειγμα, την ικανότητα ε, δανειοδότηση των τραπεζών, με την βελτίωση δυνατότητας χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σχεδίων υποδομών, διαρθρωτικών σχεδίων. Επίσης, το πακέτο αυξάνει την αναλογικότητα μειώνει το διοικητικό άχθος για τις ε, μικρές και μη σύνθετες τράπεζες και εκεί που δεν χρειάζονται ενιαία ε, πρότυπα προβλέπουμε συνεργασία. Οι μεγάλες τράπεζες από την άλλη μεριά υποχρεούνται να ενημερώνουν για τους κινδύνους σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τους κοινωνικούς κινδύνους που ε, ε, ε, υπάρχουν στην δραστηριότητε τους. Επίσης, βελτιώνουμε την συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κλπ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Το πακέτο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να συμπληρωθεί το νομοθετικό πανόραμα μετά την τραπεζική κρίση, έτσι ώστε οι τράπεζες να είναι πιο σταθερές, να βρίσκονται σε πιο σταθερά θεμέλια. Πρέπει να εφαρμόσουμε την συμφωνία για το Ταμείο Εξυγίανσης και να προχωρήσουμε στις συζητήσεις για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές των ομάδων, το ΕΛΚ, ο κύριος Κάρας για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, καταρχήν ένα θερμό ευχαριστώ στους ε, συναδέλφους Σίμων και Χέκμαρκ ε, στην ε, Κομισιόν και στους δικούς μας συνεργάτες βέβαια. Από κοινού με το νέο κανονισμό για τις τράπεζες κάναμε ένα μεγάλο βήμα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μείωση ρίσκου και κόστους στον κανονισμό και στη ρύθμιση για τις τράπεζες. Ε, αυτό το κάναμε με βάση κάποιους ακρογωνιαίους λίθους που θέσαμε. Καταρχήν λάβαμε υπόψη μας τις διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες του τραπεζικού ε, του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα. Ε, δεύτερον, για πρώτη φορά έχουμε ορισμό της αναλογικότητας των μικρών μη σύνθετων ιδρυμάτων και βέβαια έχουμε και ποιοτικά κριτήρια που προσετέθησαν. Τρίτον, δημιουργήσαμε μεγάλη διοικητική ελάφρυνση κατά 20% λιγότερο ρυθμιστικό κόστος για τις μικρότερες τράπεζες. Τέταρτον, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη προώθηση της πραγματικής οικονομίας μέσω του ε, ε, ε, ορίου αυτού των τον 1,5 με 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, έχουμε λάβει υπόψη μας την ψηφιοποίηση και τις επενδύσεις σε λογισμικό. Τέλος, πρόκειται να τεθεί τέλος στην υποχρεωτική ε, διπλή κοινοποίηση στα Μητρώα. Ε, από τη μία πλευρά ε, συμβάλαμε στη σταθεροποίηση της χρηματοοικονομικής αγοράς και από την άλλη πλευρά βοηθήσαμε και προστατεύσαμε τις μικρότερες τράπεζες. Έτσι ενισχύσαμε την οικονομική διάσταση της πολιτικής μας. Ευχαριστώ θερμά για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω σε λίγο το λόγο στην κυρία Μπερέ. Ευχαριστώ που μου επισημάνατε την τρομακτική πυρκαγιά που πλήττει ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία παγκοσμίω. Μιλάμε για την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Πανεγία των Παρισιών. Κυρία Μπερέ, έχετε το λόγο εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ. Μερικές φορές ε, βλέπουμε παράδοξα πράγματα. Εδώ βρισκόμαστε υπό το θόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ αυτός ε, της ε, Παναγίας των Παρισίων μόλις έχει καταρρεύσει. Είτε πιστεύει κανείς είτε όχι. Πιστεύω είναι ένα σύμβολο πολιτισμού. Εγώ δεν είμαι θρήσκος, αλλά είμαι συγκλονισμένη. l'adoption du paquet bancaire. Η υιοθέτηση τη δέσμη μέτρων για τι τράπεζε για να επιτραπεί η υλοποίηση των μέτρων που ελήφθησαν σε διεθνές επίπεδο μετά από την ε, οικονομική κρίση είναι ένα σημαντικό στάδιο που θέλησαν η Επιτροπή Βασιλείας και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Είναι σημαντικό αυτό το στάδιο για τη μείωση των κινδύνων που μπορεί να αναπτυχθούν εντός του τραπεζικού συστήματος. Η δέσμη αυτή μέτρων θα ενισχύσει το πλαίσιο για την εξηγένση των τραπεζών. Θα απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, παγκόσμια συστημικής σπουδαιότητας ε, να έχουν δυνατότητες δανεισμού ανακεφαλαιοποίησης. Ζήτω συγγνώμη. Μπορείτε να ξαναπάρτε το λόγο αργότερα, αγαπητή κυρία. Δίνω το λόγο στον κύριο Πακέτ για δύο λεπτά εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Κύριε Πακέτ. Κύριε Πακέτ, συγγνώμη δεν σας είχα δει. Ε, είναι όλοι συγκλονισμένοι. Έχετε το λόγο εκ μέρους του ECR για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς ε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τραπεζικό μας τομέα να βρίσκονται υπό έλεγχο οι κίνδυνοι και να υπάρχουν μαξιλαράκια για να μπορεί να αντιμετωπίσει ε, καταιγίδε όπω αυτέ που είδαμε από 10 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, την κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα που οδήγησε σε μια βαθιά ύφεση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη μεταρρύθμιση, παρότι θεωρούμε ότι οι διεθνεί νομοθεσίε έπρεπε να είναι πιο αυστηρέ. Αυτό που είναι σημαντικότερο δεν είναι οι νέοι κανονισμοί και η εποπτεία, αλλά αυτό που παρατηρούμε ότι Υπάρχουν ζητήματα άγνωστα σε κάποια κράτη-μέλη, κρυφά, τα οποία δεν μας έχουν απασχολήσει και αυτά τα τεράστια, τα διωγγωμένα χρέη ορισμένων κρατών μελών που ε, παραμονεύουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, δεν είναι εδώ ο κύριος Μακτεγάλ, οπότε δεν μπορώ να δώσω το χρόνο. Ζητώ συγγνώμη για την προφορά, κύριο αν Έχετε μισή λεπτό εκ μέρους της Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η χρηματοπιστωτική κρίση οφείλεται στις τράπεζες. Έπρεπε βέβαια να διασωθούν. Ε, όμως δεν θέλαμε να δώσουμε χρήματα των φορολογουμένων ε, και στο μέλλον ε, στις τράπεζες. Μετά την ε, εξυγίανση των τραπεζών, βέβαια, ε, δόθηκαν και άλλα κονδύλια. Ε, είχαμε ε, αναγκαστεί να προχωρήσουμε σε ένα σωρό εξαιρέσεις ούτως ώστε να σώσουμε τις τράπεζες. Έπρεπε επίσης να προσπαθήσουμε να διαχωρίσουμε τα, ε, ε, τις δραστηριότητες ε, των, ε, λοιπές δραστηριότητες των τραπεζών από τα δάνεια ε, και αυτό σίγουρα ε, θα οδηγούσε σε μια ε, ε, μεγάλη εξοικονόμηση. Σίγουρα θα μπορούσαμε να προβλέψουμε διαδικασίες πιο αποτελεσματικές και εις ό,τι αφορά τη συγχώνευση των τραπεζών. Ε, πώς θα έπρεπε να γίνει μετά από μια κρίση η διαμόρφωση της πολιτικής των τραπεζών που δεν θα οδηγήσει σε μέγα τράπεζες ε, ούτε όμως και σε ε, τράπεζες υψηλού συστημικού κινδύνου. Κύριε Γκίγκολ, δέχτε το λόγο για ένα λεπτό εκ των Πρασίνων. <coughs> Κύριε Πρόεδρε, είναι σουρεαλιστική αυτή η συζήτηση, θεωρώ. Η Παναγία των Παρισίων καίγεται. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τράπεζες. Ο χριστιανικό πολιτισμός ε, βλέπει να αναλώνεται στις σε ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία του. Ε, ελπίζω ε, να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ε, είναι αυτό που συμβαίνει είναι μια τραγωδία για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και πραγματικά ε, νομίζω ότι είναι τρέλα σε μια τέτοια στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρία άλλα συγγνώμη για την προφορά ήρθατε. Θέλετε να πάρετε το λόγο για δύο λεπτά εκ μέρου των Δημοκρατών και Φιλελευθέρων για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η πιστοτική κρίση μας έχει μείνει εξέχαστη. Οι Ευρωπαίοι θυμούνται πως χρειάστηκε να σφίξουν το ζωνάρι. Υπήρξε τεράστια δυσπιστία προς τον τραπεζικό τομέα. Ουδέποτε υπήρξε τόσο άσχημη και τώρα εδώ ε, συμφωνήσαμε στο Κοινοβούλιο ότι δεν θέλουμε ποτέ ξανά να βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση. Είναι ευτυχέ γεγονό λοιπόν που έχουμε αυτή τη δεσμή μέτρων, πολλά μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν ώστε να αποφευχθούν τέτοιε καταστάσει στο μέλλον. Στο μέλλον οι τράπεζες θα υποχρεούνται να έχουν ε, μεγαλύτερα αποθέματα, ε, αποθεματικά τα οποία ε, θα είναι κάτι θετικό. Αλλά δεν ολοκληρώνεται το καθήκον μας εδώ. Πολλές τράπεζες έχουν ε, κακά δάνεια ε, στους ισολογισμούς τους ε, και ξέρετε οι ψηφοφόροι μας θεωρούν ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό με στην επόμενη πενταετία. Χρειαζόμαστε αυστηρότερους κανόνες για τα δάνεια για παράδειγμα. Εγώ θεωρώ ότι οι τράπεζες πρέπει να προσέχουν και περισσότερο όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα. Δεν θέλουμε να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις ε, για τους καταθέτες. Χρειαζόμαστε ένα υγιές οικονομικό κλίμα να μπορούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε καινοτόμε νέες ιδέες. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να ξεφορτωθούμε όλα τα μήλα του συστήματος. Ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθόμαστε και μιλάμε τώρα για μια δέσμη μέτρων που ονομάζεται μείωση των κινδύνων εντός του τραπεζικού συστήματο τη Ευρώπη. Και αυτό που διαρωτώ με εγώ είναι πραγματικά έχουμε πιστεί ότι μειώσαμε του κινδύνου εντός του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματο, του σημαντικότερου κινδύνου. Εδώ και μια πενταετία επαναλαμβάνω σε αυτό το κοινοβούλιο ο Κίνδυνο είναι οι ρευστοί τίτλοι που κρατούν οι συστημικέ ευρωπαϊκέ τράπεζε. Μιλάμε για τα παράγωγα. Μιλάμε για τίτλου ε, που είναι δύσκολο να τιμολογηθούν και σε περίπτωση κρίσης μπορούν να υποτιμηθούν πολύ γρήγορα. Αυτοί οι τίτλοι λοιπόν της επαγρύπνησης και αυτών των κανόνων αυτή τη στιγμή καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία και αυτό είναι ένα τεράστιο σφάλμα το οποίο πιθανότατα θα πληρώσουμε ακριβά. Το μεγαλύτερο σφάλμα της μείωσης των κινδύνων είναι η συγκέντρωση της μείωσης των κινδύνων μόνο για την πίστοση. Η πίστοση είναι αυτή που δίνει ζωή στην ευρωπαϊκή οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οικογένειε που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι, μηχανήματα, οτιδήποτε. Το να περιορίζουμε μια τράπεζα να παρέχει πιστώσει ε, μόνο ε, ζητώντα ε, πολλές απαιτήσει, υπερβολικέ μερικέ φορέ, σκεφτείτε ότι παρά τις απαιτήσει που υπάρχουν ήδη με την αναθεώρηση της BRRD θα ζητάμε στις τράπεζες να πηγαίνουν να βάζουν και άλλους τίτλους στις αγορές για να παίρνουν και άλλα κεφάλαια σε περίπτωση Μπελίν και οι αρχέ εξηγήσει μπορούν να απαιτούν από τις τράπεζες να αυξάνουν και αυτές τις απαιτήσει. Και τώρα προσπαθώ να καταλάβω τώρα ποιος έχει, όποιο έχει τα χρήματα σε αυτέ τι τράπεζε θα είναι βέβαιος που τα έχει εκεί μέσα. Αν ε, μια αρχή ζητήσει από αυτή την τράπεζα να πάει στην αγορά, να ζητήσει κεφάλαια, αυτό που κάνουμε κατά την, μου, κατά την άποψή μου θα οδηγήσει σε καταστροφή. Πρέπει να ξαναδούμε ολόκληρο το οικοδόμημα τη τραπεζική Ένωση, διότι δημιουργεί σοβαρέ ανισορροπίε και ισχυρότατα προβλήματα ε, δυσπιστίας των πολιτών προ την ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπέρε. Θέλατε να ξαναπάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Να συνεχίσετε από προηγουμένω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αναχρηματοδότηση των τραπεζών είναι αναγκαία Ευτυχώς μετά από την ε, ε, οικονομική κρίση η Επιτροπή ε, Σταθεροποίησης και η Επιτροπή Βασιλείας βοήθησαν στη βελτίωση του μηχανισμού. Σήμερα έχουμε αυτό το μηχανισμό για να μειώσουμε τους κινδύνους όπου υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν στο τραπεζικό μας σύστημα. Ενισχύουμε το πλαίσιο εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών. Ενισχύουμε τους ελέγχους για τα συστημικά ε, ιδρύματα όσον αφορά την δυνατότητα απορρόφησης μειών από αυτά και την ανάγκη, ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των απαιτήσεων σε επίπεδο ποιότητας των ιδιών πόρων ε, και επιλέξιμων υποχρεώσεων. Είναι το φημισμένο MRL. Επίση, ε, ενισχύουμε όλε τι διατάξει για τι αρχέ εξυγίανση. Το πακέτο αυτό θα καταστήσει πιο στήρου του ε, κανόνες ε, ε, προβλέποντας κάποιο, κάποιο δίκτυ μόχλευσης και κάποιον δίκτυ καθαρής σταθερής χρηματοδότησης. Θα βελτιώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων υποδομών από τις τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά κριτήρια και την ανάγκη ενίσχυσης των ε, της διαχείρισης. Ωστόσο δεν επιλύει τα πάντα αυτό το πακέτο, είναι ένα βήμα μόνο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο κάτω. Για μια τραπεζική ένωση ε, θέλουμε να αποκομίσουμε όλα τα ωφέλη. Θα πρέπει να αποκομίσουμε όλα τα ωφέλη που μπορούμε να έχουμε από τις ε, απαλλαγές που μπορούν να δοθούν σε περίπτωση διασυνοριακών συναλλαγών. Επίσης αυτή η αρχή της αναλογικότητας δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι που λαμβάνονται βάσει του μεγέθου και των μοντέλων κάθε αγορά. Τέλο, μετά από χρόνια υπέρ τη ανακεφαλαίωση των τραπεζών, έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη αλληλεγγύη και επιτέλους να υιοθετήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων που έχουμε υποσχεθεί στους Ευρωπαίους ε, ε, αποταμιευτέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Φέρμπερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά τη χρηματοοικονομική κρίση η σταθερότητα είναι στο επίκεντρο του νομοθέτη. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επανελειφθεί μια κρίση όπως αυτή πριν από 10 χρόνια. Όμως ε, ε, δεν ε, είναι όλες οι τράπεζες Lehman Brothers, ούτε τόσο μεγάλες. Κάθε τράπεζα έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο έχει επίσης κινδύνους. Ε, παρόμοιος πολλές φορές με την Lehman Brothers. Ε, επίσης ε, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα των τραπεζών, τα παράγωγα κλπ. Δεν μπορεί να υπόκεινται όλοι στους ίδιους κανόνες. Θα πρέπει επίσης να μην είναι το κόστος πάντοτε το ίδιο. Πρώτη φορά με το πακέτο για τις τράπεζες έχουμε ορίσει ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ε, για το τι είναι ένα ίδρυμα ε, απλό, μη σύνθετο και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Έτσι θα πρέπει να έχουμε στην ρύθμιση για τις τράπεζες ε, αναλογικότητα. Ε, κατά την επόμενη θητεία θα πρέπει να ασχοληθούμε με το τελικό στάδιο της Βασιλείας 3 γιατί και εκεί θα πρέπει να παρέμβομαι με ανάλογο τρόπο ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε διαφοροποιημένα τα διαφορετικά ιδρύματα. Κύριε Σίλβα Περέιρα, για ένα λεπτό. Χωρίς, χωρίς μικρόφωνο. Ωραία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το καινούριο πακέτο είναι πολύ σημαντικό Στόχος είναι να ενισχυθεί η σταθερότητα του τραπεζικού στήματος στην Ευρώπη έτσι ώστε να μπορεί να αντισταθεί σε σοκ και να εξασφαλίσει την ε, εμπιστοσύνη των ε, φορολογουμένων ε, και των επενδυτών. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την εξυγίανση των τραπεζών μεταγράφουν τους πιο αυστηρούς διεθνούς κανόνες. Και οι τράπεζες οι μεγάλες τράπεζες θα πρέπει να ενισχύσουν την ε, κεφαλαϊκή τους επάρκεια. Οι κανόνες αυτοί θα μπουν σε εφαρμογή μετά από μια μεταβατική περίοδο που θα επιτρέψει στις ε, τράπεζες να προσαρμοστούν στις καινούργιες απαιτήσει χωρίς να υποσκαφθεί η δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές ε, Ζήμων και Χόκμαρκ για την εξαιρετική δουλειά τους και την εξαιρετική μας συνεργασία σε αυτά τα μέτρα μείωση του κινδύνου στο τραπεζικό τομέα. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής ε, Ένωσης με την κατανομή των κινδύνων. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Μαριά. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η μεταρρύθμιση στον τραπεζικό τομέα ήταν απαραίτητη βεβαίως μετά την τεράστια κρίση η οποία έπληξε τις κοινωνίες την τελευταία δεκαετία. βέβαια το συμπέρασμα είναι ότι οι φορολογούμενοι διέσωσαν τις τράπεζες και εν συνεχεία πλέον οι τράπεζες ιδίως στην ελλάδα επιπίπτουν επί των φορολογουμένων επί του ελληνικού λαού προκειμένου να ρυθμίσουν δήθεν τα κόκκινα δάνεια και έτσι τα κοράκια αρπάζουν τα σπίτια του ελληνικού λαού. είναι σίγουρο ότι χρειάζεται αυξημένη εποπτεία διαφοροποιημένη εποπτεία βεβαίως για τις μικρότερες τράπεζες αλλά και εκεί πρέπει να υπάρξει έλεγχος και εποπτεία. και θα ήθελα να υπάρχει έλεγχος για να δούμε τη σχέση που έχουν οι τράπεζες με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτούς οι οποίοι έχουν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις ιδίως στην ελλάδα επίσης με τις δημοσκοπικές εταιρείες διότι βλέπουμε πλέον εν ώψη ευρωεκλογών όσοι αρθρώνουν λόγο κριτικής απέναντι στις τράπεζες αποκλείονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ελλάδα όπως υπάρχει η περίπτωση η δική μας του κινήματός μας ελλάδα ο άλλος δρόμος. να ελέγξετε ποιοι έχουν πάρει δάνεια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ελλάδα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ Καλωσορίζω πολλές από τις σημαντικές εξελίξεις ε, στο πακέτο κεφαλαίων απαιτήσεων, όπως οι νέες ε, διατάξεις για την καταπολέμηση του ξεπλήματο μαύρου χρήματος και οι απαιτήσει ε, ίδιων κεφαλαίων. Το TILAC θεωρείται από πολλού αποτελεσματική λύση για να επιληθεί το πρόβλημα των τραπεζών που είναι πολύ μεγάλε για να αποτύχουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό είναι δυνατόν χωρί μια μεγάλη μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα και μεγαλύτερο δίκτυ μόχλευση. Ε, η εξηγήνση των τραπεζών έχει αποδειχθεί ήδη ότι τελικά ε, πληρώνεται από τους φορολογουμένους. Ε, στη αρχή των διαπραγματεύσεων εμείς είχαμε εκφράσει ανησυχίες για το 3% δίκτυ μοχλευσής. Θα, να θυμηθούμε ότι ο ΣΑ και η ΕΠΑ συνιστούν δίκτυ μόχλευσης τουλάχιστον 5% για ιδρύματα συστημικής σημασίας. Ε, ε, αφήνουμε δηλαδή να γίνουν ανταγωνιστικέ οι τραπεζέ μα προ Αμερικέ ε, θέτοντα σε κίνδυνο τη σταθεροποίηση. Το πρόβλημα του too big to fail δεν θα το λύσουμε με μια μεταρρύθμιση μόνο. Για να μειώσουμε τον κίνδυνο πρέπει να διαχωρίσουμε τι υπηρεσίε λιανική από τι επενδυτικέ υπηρεσίε. Το θέμα ότι μια δεκαετία μετά από την οικονομική κρίση οι νομοθέτε δεν καταφέρουν να το επιτύχουν είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου. Απόλυτη αποτυχία κάλυψη ικανοποίηση των προσδοκιών των Ευρωπαίων πολιτών προς εμάς. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ουρτασούν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι πρώτε μου σκέψει στρέφονται προ του Γάλλου, του Παρισινού άνδρε και γυναίκε για αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε στην Πανεγία των Παρισίων. Είναι φρικτή η είδηση, είναι μια μαύρη ημέρα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και θα ήθελα να εκφράσω την ελληνική μου προ του πυροσβέστε τη υπηρεσία που καταβάλουν προσπάθειες για να κατασβέσουν την πυρκαγιά αυτή και θα ήθελα να αφαιρώσω τα λίγα δευτερόλεπτα που μου μένουν για να ευχαριστήσω τον κύριο Χόκμαρ. Κάναμε πολύ καλή δουλειά μαζί ε, ε, σημαντικά επίπεδα MRL και TILAC ώστε να μην ξαναχρησιμοποιήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων στην επόμενη κρίση. Κάναμε πρόοδο. Θέλω να τον ευχαριστήσω επειδή δέχτηκε και τις προτάσεις μας ε, περί προστασίας και να αποφύγουμε να παγιδευτούν οι μικροί αποταμιευτέ σε καταστάσεις ε, bail-in όπως έγινε στο παρελθόν. Το επιτύχαμε πιστεύω αυτό στο κείμενο και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. κυρία Πιέτικανεν για ένα μισή λεπτό. Uh, Τα θερμά μου συλληπιτήρια για την ε, καταστροφή που υπέστη η πολιτιστική αυτή ε, αυτό το μνημείο, το πολιτιστικό μνημείο που ανήκει όχι μόνο στη Γαλλία αλλά σε όλους τους Ευρωπαίους. Εδώ ολοκληρώνεται η μεγάλη δέσμη μέτρων που θεσπίσαμε μετά από την οικονομική κρίση για να σταθεροποιήσουμε τον τραπεζικό τομέα σε σχέση με κινδύνου ε, και να δημιουργήσουμε μηχανισμού εξυγίανση και να επιβάλλουμε τι απαραίτητε κεφαλαίκε απαιτήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ του συζητητέ για την καταπληκτική δουλειά που έκαναν. Θα ήθελα όμω να υπενθυμίσω στην Κομισιόν και στο επερχόμενο Κοινοβούλιο ότι απομένουν δύο προκλήσει μπροστά μα. Η πρώτη είναι οι δέσμοι μέτρων ε, που αφορά το διαχωρισμό μεταξύ των επενδυτικών τραπεζικών συναλλαγών και των λιανικών. Και απ' την άλλη είναι ότι οι τράπεζες και οι δανειοδότηση θα έπρεπε να ανήκουν στα βιώσιμα κεφάλαια, διότι εκεί θα πρέπει να αποφύγουμε οικονομικές κρίσεις, ε, χρηματοπιστωτικές κρίσεις που ενέχουν κάποιες επενδύσεις. στα ορυκτά καύσιμα, για παράδειγμα. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Τάν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι λυπηρό το, λυπηρές ειδήσεις από το Παρίσι. Το τέλος θητείας αναρωτιόμαστε αν έχουμε μάθει τα διδάγματα της ε, χρηματοοικονομικής κρίσης. Δεν έχουμε κανόνες που να ξεχωρίσουν ε, την επενδυτική τραπεζική από την λιανική τραπεζική και ταυτόχρονα δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση. Οι τράπεζες ακόμα είναι υποκεφαλοποιημένες και ευαίσθητες, ευάλωτες. Οπότε αυτοί οι κανόνες είναι θετικοί. Οι συστημική σημασία τράπεζες θα πρέπει να έχουν πολύ περισσότερα ίδια, ε, ε, ίδια κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Ε, Επίσης, δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το ρόλο ε, της αξιολόγησης, του αξιολογητή. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μαθαίνει από την κρίση και κοιτάει στο μέλλον. Ε, είναι ένα θετικό βήμα, αλλά ένα μόνο βήμα στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταρμπάτη, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ο πρώην ε, πρόεδρος ε, ο Χόρστ Κέλλερ είχε ε, δει την αντιμετώπιση της κρίσης μέσα από την διαφοροποίηση του κόστους τη τα, τα, ε, επιτόκια ε, έπαιξαν επίσης ένα πολύ μεγάλο ε, ρόλο και δημιουργήθηκε έτσι ένας φαύλος κύκλος που χαρακτηρίζει και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα πρέπει ε, να, τα, τα, ε, ομόλογα να στηρίζονται από τους ίδιους πόρους. Αυτό όμως απορρίπτεται. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα underpricing of risk και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται με τις υπερχρεωμένες χώρες και την ε, ε υπονόμευση της νομισματικής ένωσης. Ε, θα ήθελα να έκανε λάθος η Ομοσπονδιακή Τράπεζα σε εκτιμήσεις της, αλλά ε, δυστυχώς έχει δίκιο. Ο κ. Βιέγας, πάνω από μια δεκαετία πέρασε από την κρίση του 2008. Τέσσερα τρισεκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν ε, για την αναχρηματοδότηση τραπεζών. 16 δισεκατομμύρια ε, στην Πορτογαλία μόνο. Μετά από τόσα χρόνια κρίση, μετά από δεκάδες οδηγίες, κανονισμούς, το ερώτημα είναι ποια είναι η πρόοδος. Γιατί στην Πορτογαλία βλέπουμε ότι η βρύση είναι ανοιχτή. 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην Novo Μπάνκο ε, το 2018-2019 για παράδειγμα. Και, στο, και Άλλα 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπονται για την περίοδο 2020-2021. Ας είμαστε σαφείς, αυτές οι οδηγίες, αυτοί οι κανονισμοί δεν είναι τίποτα άλλο από καλοπιστικά κείμενα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο δημόσιος έλεγχος στο τραπεζικό σύστημα έτσι ώστε οι τράπεζες να εξυπηρετούν την οικονομία και όχι η πραγματική οικονομία της τράπεζα, όπως, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστούμε. Άνοιξε το Catch the Eye με τον κύριο Καπούτο, ο οποίος θα το κλείσει κιόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να ολοκληρώσουμε ε, την Τραπεζική Ένωση, έχουμε πολύ δρόμο. Χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις ώστε να προλάβουμε τις μελλοντικέ τραπεζικές κρίσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει, για παράδειγμα, να διασφαλίσουν επαρκή απορρόφηση των ζημιών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να μειωθεί η επίδραση στην χρηματοπιστική σταθερότητα και τους φορολογουμένους. Είναι σημαντικό να υπάρχουν αρχές ικανές να παρεμβαίνουν άμεσα ώστε να απορροφούνται ε, οι δυσκολίε ε, του τραπεζικού τομέα και να διασφαλίζονται οι διασυνοριακέ αγορέ όπου όλοι οι καταναλωτέ θα μπορούν να υποφελούνται από τα θετικά αποτελέσματα ενό ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματο. Μέγιστη προσοχή χρειάζεται τέλο στην αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον κοινωνικό τομέα, ευνοώντα μέτρα που θα μα ε, επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε αυτού του κινδύνου επαρκώ. Θα πρέπει να κινηθούμε προ αυτή την προσπάθεια ώστε να μειώσουμε του κινδύνου του χρηματοπιστωτικού συστήματο, διασφαλίζοντα ταυτόχρονα τον πιο ενεργό ρόλο των τραπεζών για την αύξηση, την ανάπτυξη και τι επενδύσει. Αφού ολοκληρώθηκε το Catch the Eye, ο κ. Ντομπρόφσκη θα μα βοηθήσει να κλείσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα και εγώ να ε, εκφράσω ότι είναι, λείπουμε και βρίσκομαι σε σοκ σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην Νότρνταμ, στο Παρίσι. Η Νότρνταμ ε, είναι ένα σύμβολο όλου του ευρωπαϊκού πολιτισμού και όλη τη ανθρωπότητα, όχι μόνο της Γαλλίας. Τώρα επιστρέφοντας στο τραπεζικό πακέτο. Το πακέτο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση των κινδύνων του χρηματοοικονομικού χρηματοπιστωτικού τομέα. Οπότε χαίρομαι που το Κοινοβούλιο έχει στηρίξει την ομοθέτηση αυτού του πακέτου και μετά την ψηφοφορία αύριο θα ενισχυθεί όχι μόνο ε, η αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος αλλά θα τεθούν και τα θεμέλια για να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Οπότε χαίρομαι που θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για αυτό το θέμα. Ο χρηματοπιστωτικό μας τομέας θα γίνει πιο σταθερός, πιο ανθεκτικός και θα ανοίξουμε το δρόμο για την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Ελπίζω ότι η πολιτική συμφωνία θα υπερψηφιστεί αύριο. Σε ευχαριστώ όλους. Euh, Ο λόγος του κύριου Χόκμαρ καταρχήν. Καταρχήν στην κυρία Μπερέση και στους Γάλλους συναδέλφους θα ήθελα να πω ότι τα είδη είναι πολύ δυσάρεστες από τη Γαλλία, από το Παρίσι και δυσάρεστες για όλους μας. Γιατί η Νότρο Ντάμ είναι η δική μας κυρία, Νότρο Ντάμ. Και στην ιστορία αλλά και ως ε, εμβληματικό σημείο της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Σε ό,τι αφορά το τραπεζικό πακέτο Ήδη ελέγχθησαν πολλά σήμερα. Όμως είναι σωστό να πούμε ότι το πανόραμα πια έχει αλλάξει. Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας είναι αυτή τη στιγμή πολύ πιο αθεκτικός και πολύ πιο προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη κρίση του στο μέλλον. Αν τέτοιου είδου κρίση παρουσιαστεί. Και προφανώ κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί. Το θέμα είναι πώ θα την αντιμετωπίσουμε. Εμεί είμαι πεπισμένο ότι ε, με όσα έχουμε αποφασίσει μέχρι τώρα και με αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή, με την ε, με την ιεραρχία, με τη δυνατότητα των διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών, όλα αυτά ε, έχουμε βελτιώσει την κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα έχουν λυθεί. Έχουμε δημιουργήσει όμως τους μηχανισμούς έτσι ώστε αυτοί που είναι υπεύθυνοι στην α ή τη β περίπτωση να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Και χαίρομαι που το πετυχαίνουμε αυτό. Είναι η τελευταία έκθεση που παρουσιάζω στην Ολομέλεια σε αυτή τη θητεία, κυρία Πρόεδρε. Και είμαι περήφανος που τα καταφέραμε μαζί. Θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου στους συναδέλφους από όλα τα από όλες τις πολιτικές ομάδες ανεξαρτήτως χρώματος και προέλευσης, χρώματος ενώ πολιτικού χρώματος και προέλευσης και ε, από το καναπέ μου θα παρακολουθήσω τη συνέχεια τα επόμενα χρόνια. Obwohl jeder der Kollegen, der hier sprechen konnte, eine sehr Οι συνάδελφοι είχαν περιορισμένο χρόνο, αλλά όλοι ε, μίλησαν για την τρομερή αυτή πυρκαγιά που μας οδηγεί σε αλληλεγγύη με την Γαλλία και τους Γάλλους συναδέλφους. Ε, επί δυόμιση χρόνια με αυτό το πνεύμα εργαστήκαμε και πάντα αυτό το σώμα εργάζεται ε, με αυτό το πνεύμα. Ε, όταν δούμε την άκρα αριστερά και άκρα δεξιά ε, βλέπουμε ε, μία απουσία όσοι όμως εργάστηκαν επί δυόμιση χρόνια για την έκθεση αυτή ή βρίσκονται εδώ και έπρεπε να λάβουν θέση όλο αυτό το διάστημα. Ε, ας ακολουθήσουμε το δρόμο προς μεγαλύτερη ασφάλεια, μικρότερο κίνδυνο, με παράλληλη ε, διευκόλυνση εκείνων που δεν ε, συνέβαλαν στην ε, πρόσφατη κρίση και που αντιμετωπίζουν κινδύνους οι ίδιοι. Ε, νομίζω ότι τα προηγούμενα δυόμιση χρόνια μπορέσαμε να δούμε τις ανάγκες των άλλων, τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Ε, αν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό με πνεύμα αλληλεγγύης, και αν μπορέσαμε να σταθεροποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο τις τράπεζες, όχι όμως ε, σε βάρος ε, άλλων, τότε συμβάλαμε στην εξισορρόπηση των συμφερόντων στην Ευρώπη και αυτό ε, αποτελεί μια καλή βάση για περαιτέρω συνεργασία στην Ευρώπη και για καλύτερη ακόμα εξυγίανση των οικονομικών της. Ευχαριστώ ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Κλείνει εδώ η συζήτηση. Περνάμε στην έκθεση Φερνάντες. Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα. Κύριε Φερνάντε, έχετε το λόγο αμέσω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Τόμπροφσκη. Ε, είναι πράγματι δύσκολη στιγμή να συζητάμε εμείς εδώ ακούγοντας τις ειδήσει από το Παρίσι αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που καταστρέφει ε, ένα από τα σημεία, πολιστικά σημεία αναφοράς της Υπήρου μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η τελευταία συζήτηση για αυτό τον κανονισμό προκειμένου ε, πριν από την αυριανή ψηφοφορία να συζητήσουμε μια πρόταση την οποία η Κομισιόν είχε επιβάλει εδώ και αρκετό καιρό και ήταν αρκετά περίπλοκη. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την στήριξη και την αλληλεγγύη, το πνεύμα συνεργασία όλων των εισηγητών των διαφορετικών πολιτικών ομάδων, διότι πραγματικά δεν θα ήταν εύκολο να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία η οποία επικυρώθηκε πριν μερικέ εβδομάδε στην Επιτροπή και ελπίζω αύριο από την Ολομέλεια. Συζητάμε για το τραπεζικό πακέτο που θα ψηφίσουμε αύριο και την ανάγκη ε, το τραπεζικό σύστημα να είναι πιο ανθεκτικό εναντί κρίσεων στο μέλλον. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή και θα ψηφίσουμε αύριο είναι πώς θα αποφύγουμε ε, μεσονομικές κρίσεις όπως αυτή του 2010-2012 διότι ε, τα, οι εξηγιάνσεις δημιούργησαν κρατικά ελλείμματα ε, που έθεσαν σε πολύ δύσκολη θέση το κράτο, ε, ε, την δημοσιονομική κατάσταση των ορισμένων κρατών μελών, μάλιστα που ζήτησαν και την και, ε, συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα επιτρέπουν να καταπολεμήσουμε αυτές τις κρίσεις ε, ε ρευστότητας ε, σε ό,τι αφορά το δημόσιο κρέος. Η πρόταση της Κομισιόν ήταν ε, στη σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι καταφέρουμε να τη βελτιώσουμε έτσι περισσότερο. Να βελτιώσουμε την δυνατότητα των ευρωπαϊκών αρχών να εποπτεύουν ε, τους τίτλους που είναι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα. Η ΕΜΣΑ έχει πλέον μεγαλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας και ε, βελτιώνουμε επίσης ε, την κατάσταση της ε, την χρήση αυτού του μέσου που θα επιτρέψει, του εργαλείου που θα επιτρέψει ε, την διαφοροποίηση των εργαλείων που διαθέτουν τα κράτη και οι τράπεζες. Οι προτάσεις μας εξασφάλισαν μια ευρεία συμφωνία. Ε, χρειάζεται να μεταρρυθμιστεί η ζώνη του ευρώ έτσι ώστε να διαθέτουμε μέσα εργαλεία που θα μας ε, βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε κρίσεις παρόμοιες με αυτήν του 2010-2012. Θέλουμε ένα τραπεζικό σύστημα ασφαλές, αλλά και εργαλεία που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν μελλοντικές κρίσεις χωρίς να χρειάζεται ε, να ε, καταλήγουν σε μνημόνια ε, που χειροτερεύουν την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης. Είναι ένα βήμα, ένα αποφασιστικό βήμα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας προκειμένου η, η ζώνη του ευρώ να έχει μέλλον, να είναι αθεκτική και σταθερή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντομπρόφσκης. Έχετε το λόγο. So, <clears throat> uh, uh, Madam Chair, uh, Mr. Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι αγαπητά μέλη, είναι σημαντική αυτή η συζήτηση σήμερα για τους τίτλους που είναι εξασφαλιζόμενοι με κρατικά ομόλογα. Αυτά τα SBBS είναι ένα σημαντικό εργαλείο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε μια πιο ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση και πιο αποτελεσματική ένωση κεφαλαίου Θα βοηθήσουν τον καταμερισμό των κινδύνων και διασυνεργειακά στον τραπεζικό τομέα και αποτελεί για τις τράπεζες ένα επιπλέον εργαλείο διαφοροποίησης ε, των ε, ανοιγμάτων του σε κρατικά ομόλογα. θα βοηθήσει να αποφύγουμε παλιότερα ευάλωτα σημεία που οδήγησαν στην κρίση. Όπως ξέρετε, το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει ε, και κάποια εμπόδια για τι ε, SBBS όπου θα βρισκόταν σε ρυθμιστική ε, μειονεκτική θέση σε σχετικά με κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης. Με την πρότασή μα ουσιαστικά θα υφίστανται την ίδια ρυθμιστική μεταχείριση όπως και τα κρατικά ομόλογα χωρίς να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβαιότητα αφού θα είναι ιδιωτικά ε, μέσα για ιδιωτική χρήση. Επίσης θέλω να τονίσω ότι η πρότασή μας ε, δεν αλλοιώνει τη ρυθμιστική μεταχείριση των ε, κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης. Απλά δίνει σε αυτά τα, στους τίτλους την ίδια μεταχείριση στον κύριο Φερνάνδε, εισηγητή και σε όλα τα μέλη τη Επιτροπή ε, ΕΚΟΝ. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου για αυτό το αρχείο, για ε, αυτό το θέμα που ψηφίστηκε επιτυχώ ε, στι 21 Μαρτίου και που ελπίζουμε να υπερψηφιστεί εδώ. Αυτό θα στείλει ένα χειρό μήνυμα στο Συμβούλιο για το πόσο σημαντικό είναι για την Κομισιόν και για το Κοινοβούλιο το θέμα αυτό. Γεγονός που θα πρέπει να ε, οδηγεί το Συμβούλιο να δώσει νέα προτεραιότητα σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα τις ομάδες. Το ΕΛΚ ο κύριο Γκέρολ για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η παρούσα πρόταση για την ε, απάλληψη ρυθμιστικών εμποδίων ε, για τους τίτλους είναι σημαντική συνεισφορά σταθερότητα του, του χρηματοοικονομικού συστήματος. Οι διατάξεις δημιουργούν μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη ολοκλήρωση και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε σε σχέση με άλλες εναλλακτικέ και δημιουργεί λιγότερους κινδύνους για τα δημόσια, τους δημόσιους προϋπολογισμούς. Οι κίνδυνοι ε, σημαίνουν ότι οι επενδυτές ε, διαφοροποιούν πανευρωπαϊκά τα, ε, την προσφορά τους. αυτό είναι θετικό γιατί οδηγεί και σε δικτύωση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών. Πιστεύουμε ότι μπορούμε έτσι να δημιουργήσουμε βάσεις για να οικοδομήσουμε περαιτέρω την ε, πολιτική μας μετά την ε, χρηματοπιστωτική κρίση. Θα πρέπει με φιλοδοξία και στοχοπροσύλωση να συνεχίσουμε λαμβάνοντας περισσότερα μέτρα ε, προς τη σταθερότητα και να μην υπονομεύσουμε μακροπρόθεσμα το σύστημά μας. Είναι σημαντικό ότι ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ε, ως το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για την επίτευξη όλων αυτών. Ο κ. Πάκετ. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να συζητάμε την ώρα που καίγεται, γίνεται στάχτη η Νότρονταμ. Είναι μια πολιτιστική καταστροφή τεραστίων διαστάσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, οδηγία, την ε, πρόταση για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού μας συστήματος, προφανώς ε, τα ε, κρατικά ομόλογα αποτελούν πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα με εργαλεία τα οποία δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Τέτοιου είδου εργαλεία τα χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε για παράδειγμα αξιόγραφα τα οποία εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια και τέτοια. Ε, η αδιαφάνεια ήταν πολύ μεγάλη και ε, οι αγορές αυτές ήταν αγορές πολύ ψηλού κινδύνου. Πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί ο κίνδυνος και στα κράτη-μέλη με αυτόν τον τρόπο. Χρειαζόμαστε καλύτερα μέτρα για να βελτιώσουμε το τραπεζικό μας σύστημα. Ο κ. Καλβέ Σομπό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάλφε Χωνάς Φερνάντεθ και από τη συναλφή ασφαλώς και δεν μπορώ να αρχίσω με άλλο τρόπο παρά ε, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μου για την κατάρρευση ενός τμήματος της ε, ψυχής της Ευρώπης. Ε, τα συλληπιτήριά μου λοιπόν όχι μόνο στους Γάλλους ε, φίλους αλλά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε όμως ε, κατασκευάσει και πολλά άλλα πράγματα με πολλή προσπάθεια. Η, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ για παράδειγμα. Και είναι εξαιρετικά ευάλωτοι. Ευάλωτα αυτά τα πράγματα και πέρασε μια ολόκληρη σχεδόν θητεία χωρίς να έχουμε στηρίξει επαρκώς το ευρώ. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια της Κομισιόν, εξαιρετική η δουλειά του Χώνας ε, και, και των συναδέλφων, έτσι ώστε να έχουμε ένα στοιχείο ενεργητικού ευρωπαϊκής φύσης που θα συνδέεται και θα στηρίζει το ενιαίο νόμισμα που είναι το ευρώ. Γίνεται λόγος για αμοιβαία κάλυψη κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανενός είδους αμοιβαία κάλυψη. Δεν υπάρχει. Είναι λόγια του αέρα αυτά. Λέγεται ότι δεν θα το θέλουν οι αγορές κλπ. Ε, ας το αφήσουμε να λειτουργήσει και θα δούμε αν θα το θέλουν οι αγορές ή όχι. Ας δούμε τι θα πούν οι αγορές. Το προϊόν αυτό είναι ευρωπαϊκό προϊόν που στηρίζει το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, επιτρέπει την διαφοροποίηση των ε, αξιογράφων και επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στις ε, χώρες που έχουν υψηλό κρατικό δανεισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν οι ε, κοινωνικές πολιτικές, για παράδειγμα. Και παρά τα εμπόδια είναι μια προσπάθεια ε, να αυξηθεί η αλληλεγγύη στη ζώνη του ευρώ. Δεν περιθωροποιείται κανένα κράτος ε, της ε, ζώνης του ευρώ. Κανένα. Σε αντίθετη περίπτωση ασφαλώς θα είχαμε αποτύχει. Τώρα, δεν αρέσει στον γαλλογερμανικό άξονα, ας προτείνουν κάτι άλλο. Αν, αν δεν το κάνουν, ε, ας είμαστε περήφανοι διότι καταφέραμε κάτι το οποίο πραγματικά υποστηρίζει το ευρώ. Ευχαριστώ. Εκ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, ε, είναι δύσκολο να συζητήσουμε ε, με περιορισμένο ε, χρόνο για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης ε, που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η καταπολέμηση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί σίγουρα ε, έχει αυξηθεί η σταθερότητα και εδώ ε, έχει ε, παίξει ρόλο και η πολιτική μας για τα μέτρα αυτά κεφαλαϊκές απαιτήσει, μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα τα SBBS ε, σίγουρα δεν αποτελούν εκβάθρο διορθωτικό μέτρο αλλά ε, θα μπορούσαν ενδεχομένως να αυξήσουν κατά τη τη σταθερότητα. Εμείς θέλουμε σταθερή ευρωζώνη γι' αυτό όμως χρειάζεται πρωτίστως μια κεντρική τράπεζα η οποία ε, θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και δεν θα προβάλλει η Γερμανία μόνο ε, ε, με την υπέρμετρη προάσπιση των συμφερόντων τους. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και ε, ευρωπαϊκά ομόλογα. Ευχαριστώ κύριο Σερτουσόν. Ούρτασουν για ένα λεπτό. Θέλω να ευχαριστήσω, <clears throat> να συγχαρώ τον κύριο Φερνάντεθ. Ε, δεν ήταν εύκολο το έργο του, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πολύ καλή δουλειά του. Η δική μου πολιτική ομάδα θεωρεί ότι αυτό δεν αποτελεί λύση των διαστατικών προβλημάτων που έχει το ευρώ. Ε, προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε τα ευρωπαϊκά ομόλογα με ένα άλλο όνομα. Δεν πρόκειται όμως να μας ε, βγάλει αυτό το εργαλείο από τα διαστατικά προβλήματα που έχει ο σχεδιασμός του ευρώ. Ε, χαίρομαι παρόλα αυτά που ο κ. Φερνάντε δέχτηκε μερικέ από τι προτάσει μα ε, για του τίτλου εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε πολύ καθαρά ε, την ε, ρευστότητα των τραπεζών έτσι ώστε η δημιουργία αυτού του εργαλείου να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις. Επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ε, θα έχει ε, μια ένα μακροεποπτικό ρόλο πολύ σημαντικό. Συγχαρητήρια λοιπόν μια φορά στον κύριο Φερνάντε. Ο για ένα λεπτό για μια ακόμη φορά η ευρωπαϊκή ένωση μηχανεύεται τρόπους να στηρίξει το χρηματοπιστωτικό τομέα μειώνοντας τον κίνδυνο για τις τράπεζες με την ανάπτυξη τίτλων στην αγορά εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα. δυστυχώς κύριοι το έργο το έχουμε ξαναδεί. στην ελλάδα οι ομολογιούχοι που είχαν επενδύσει αγοράζοντας κρατικά ομόλογα είδαν σε μια νύχτα τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται πολλοί έλληνες επενδυτές είδαν τις περιουσίες τους να χάνουν το 53,5% τρία πέντε της αξίας τους ενώ η ζημιά σήμερα υπερβαίνει το. 75%. πέντε στις 12 μαρτίου του 2012 με το περίφημο psi για το κούρεμα του ελληνικού χρέους το οποίο στην ουσία έγινε για τη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών εκτός από τους μικροεπενδυτές έχασαν και τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία γύρω στα δώδεκα δισεκατομμύρια ευρώ. αυτή ήταν η αρχή με την οποία καθ' υπόδειξη των δανειστών και τη συνεργασία των πρόθυμων ελληνικών κυβερνήσεων μειώθηκαν συντάξεις κύριες και επικουρικές τα επιδόματα προνοίας μετοχικών ταμείων και ταμείων αλληλεγγύη. για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε πως τι λάθο πολιτικές τη ενώσεω τι πληρώνουν οι πολίτες των ευρωπαϊκών κρατών. ευχαριστώ. η χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. ιδίως στην ελλάδα είχαμε το περίφημο psi το κούρεμα των κρατικών ομολόγων αυτό που οδήγησε στη φτώχεια χιλιάδες μικροομολογιούχους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν χρήματα ούτε καν να πάνε να έχουν μια ιατρική περίθαλψη. ταυτόχρονα κουρεύτηκαν και τα κρατικά ομόλογα τα οποία είχαν τα ασφαλιστικά ταμεία. η ζημιά ξεπέρασε τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. ποιος όμως εξαιρέθηκε; εξαιρέθηκαν τα ομόλογα που είχε η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο κέρδισε η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα διαλύθηκε η ελληνική οικονομία. τα προβλήματα της ευρωζώνης δεν αντιμετωπίζονται με ασπιρίνες όπως είναι η συγκεκριμένη πρόταση ούτε με κρατικές εγγυήσεις διαφόρων ομολόγων που θα εκδώσουν οι τράπεζες. χρειάζεται αλλαγή στη δομή της ευρωζώνης. πρέπει να είναι μια ευρωζώνη που θα υπηρετεί όλους τους λαούς και δεν θα υπηρετεί τη γερμανική ευρώπη. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε ομιλητές κατσιά, οπότε δίνω μαζί στο λόγο στον Επίτροπο των Πρόσκης. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις προσπάθειες για το προτινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους τίτλους που είναι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα. Όπως είπα πρωτήτερα, ελπίζω να φέρει καλά αποτελέσματα και στο Συμβούλιο το θέμα αυτό. Σημειώνει η Κομισιόν τα αιτιολογήσεις του Κοινοβουλίου, τις μελετά προσεκτικά με σκοπό να ξεκινήσει επικοδομητική συζήτηση και με το Συμβούλιο στο άμεσο μέλλον. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο εισηγητή, τον κύριο Φερνάντες σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Φερνάνδες. Θέλω να επωφεληθώ αυτών των δύο λεπτών για να ευχαριστήσω ειλικρινά και εκ βάθους καρδίας όλων των εισηγητών, όλους τους εισηγητές, ε, Θυμάστε ότι είχαμε ξεκινήσει με πολλέ απορρίψει και μια κατάσταση πολύ περίπλοκη, αλλά του τελευταίους μήνε όλε οι πολιτικέ ομάδε έδειξαν μια βούληση να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Όμπε που ήταν εισηγητή σε ένα μεγάλο τμήμα του προηγούμενου έτους. Χωρίς τη δική του δουλειά ε, δεν θα τα είχα καταφέρει όταν μου ανατέθηκε το έργο. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλείνει μια θητεία με ένα σημαντικό επιτεύγμα. Η σημερινή συζήτηση και η αυριανή ψηφοφορία όλων αυτών των κανονισμών και οδηγιών δείχνουν ότι το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να προωθήσει τη ζώνη του ευρώ. Η ψηφοφορία αυτή ιδιαίτερα είναι ένα ακόμα βήμα στην δημιουργία της Νομισματικής Ένωσης, μια σταθερής ζώνης του ευρώ. Προφανώς ε, θα θέλαμε να είχαμε προχωρήσει περισσότερο. Το Κοινοβούλιο όμως ε, δίνει μάθημα ε, φιλοευρωπαϊσμού και ελπίζουμε ότι στην επόμενη καδιάρκεια της επόμενης θητείας το Συμβούλιο θα κλείσει το, ε, την διαδικασία αυτή. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και θα πρέπει να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συναδέλφοι, κλείνει η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Υποπτείας. Εκθέσεις των κυρίων Κάρας και της κυρίας Μπερές, Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και Χρηματοοικονομικές Αγορές. Και πάλι μια εκθέση των ιδίων καρά και Μπερέ, μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματο Ευρωπαϊκή Ένωση και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Και η τρίτη έκθεση και πάλι των ιδίων Καρά και Μπερέ, αγορέ χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλιση και αντασφάλιση. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Δίνουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Κάρας, για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά παράδοξο. Πριν από δέκα χρόνια ε, συμμετείχα σε μια μεγάλη έκθεση για τις επιπτώσεις ε, της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και συνεργάστηκα με μια Γαλλίδα, την συνάδελφο Μπερές. Πρόσφατα ανέλαβα έκθεση ε, ε, για την ε, Τρόικα και τη δράση της στις χώρες που λειτουργήσαν με μνημόνια. αργότερα με την Περβάνς Περές προχωρήσαμε στην τελευταία έκθεση. Παράλληλα και ε, τώρα ε, κατέρευσε η Νότρο ε, όλοι ε, εκφράζουμε τη θλίψη μας, όλοι νιώθουμε θλίψη γιατί δεν είναι μόνο πυρκαγιά, είναι κατάρρευση και ένα δικό μας κομμάτι νιώθουμε ότι κατέρευσε. Είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάντα προσπαθούσαμε να ξεπερνούμε τα ιδεολογικά μας όρια και να προβάλλουμε τα κοινά σημεία. Ε, πάντοτε ε, προσπαθήσαμε να ε, κάνουμε ένα συγκερασμό των ιδεών. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Περβάνς, ε, για το έργο σου σήμερα, τη μέρα αυτή της θλίψης κάποια ε, σημαντικά στοιχεία βλέπουμε ε, να καταραίουν άλλα όμως ε, στοιχεία βλέπουμε μέσα από τη συνεργασία μας να προχωρούν και ποτέ δεν πρέπει να παραιτηθούμε από αυτή την προσπάθεια. Οι τρεις εκθέσεις που καταρτήσαμε από κοινού αποτελούν ένα ορόσημο και σε ευχαριστώ και εσένα και όλους τους σκιώδεις για τη συνεισφορά σας. Δημιουργούμε νέες αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών ε, με ε, ε, συνδυασμό εποπτείας και ελέγχου. Μια άμεση εποπτεία ευρωπαϊκή σε κάποιες διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη ε, λήψη υπόψη ε, ιδιαιτεροτήτων, σύνθετων στοιχείων, διαφορετικών προφίλ, ε, καλύτερα, ε, καλύτεροι μηχανισμοί, καλύτερα μέσα, καλύτερο συντονισμός, περισσότερη προστασία των καταναλωτών και αντιμετώπιση κινδύνων συνεχών. Ε, μεγαλύτερη, ε, καλύτερη ρύθμιση ε, διασυνοριακών συναλλαγών και καλύτερη λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενισχύουμε τη διακυβέρνηση με καλύτερη αποτελεσματικότητα, ταχύτερες αποφάσεις, αποφυγή, σύγκρουση συμφερόντων περισσότερες ε, ε, αρμοδιότητες των οργάνων, ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς ε, λέμε ότι θα πρέπει να διατίθενται στις αρχές αυτές ε, επαρκής οικονομική πόρη αλλά και προσωπικό. Και δημιουργούμε ε, συνθήκες βελτίωσης στο μέλλον για την αντιμετώπιση των συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων υπάρχει πρόοδος γιατί συνεργαστήκαμε όλοι. Και αυτή η συνεργασία ελπίζω να συνεχιστεί ε, και κατά την προεκλογική εκστρατεία και να καθορίσει και την πολιτική του επομένου Κοινοβουλίου. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπερέζ για τέσσερα λεπτά. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητέ Οτμαρ Κάρας, είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε πράγματι και πράγματι πιστεύω συνεργαστήκαμε τόσο καλό σου και την πρώτη φορά. Η Επιτροπή πρότεινε κάτι πολύ καλό, με συνοχή. Αν τα κράτη-μέλη θέλουν μια ένωση κεφαλαίου αγορών, πρέπει να ενισχυθούν οι ε, εποπτικές αρχές. Ε, δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επόμενη κρίση για να αντιληφθούμε ότι όταν αναπτύσσουμε μια αγορά καλύτερα είναι να υπάρχει κάποιο χωροφύλακα να τον επιτηρεί, ανεξάρτητα από την ποιότητα των συμμετεχόντων. Και πράγματι, κύριε Οτμαρκάρα, όταν αναλάβατε την ευθύνη μαζί μου για αυτή την έκθεση, ε, το παιδί αυτό δεν πήγαινε πολύ καλά. Μερικοί θεωρούσαν ότι είχε πεθάνει και μάλιστα κάποια κρατημέλη χαίρονταν. Και εμείς το σώσαμε φροντίσαμε τα κράτη-μέλη να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόσχημα ότι πολιτικά θα τους ήταν ωφέλιμο να κάνουν πρόοδους μόνο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, αλλά να θεωρούν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πρόοδους πραγματικές χωρίς να αντιμετωπίσουμε το πραγματικό πρόβλημα, την άσκηση της εξουσίας των εποπτικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως είναι κάτι λιγότερο δύσκολο, αλλά είναι ένα στάδιο που απαιτείται το εξή το να σημειωθεί πρόοδος για τα θέματα βιωσιμότητας, οι αρχές εποπτείας στον τραπεζικό τομέα, στον ασφαλιστικό τομέα, στο τομέα των ακινήτων θα πρέπει να βλέπουν πόσο βιώσιμα είναι τα μοντέλα που υλοποιούν οι θεσμοί. Παρομοίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, έχουμε πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα βάσει των εξουσιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την εποπτική αρχή των κινητών αξιών στον τομέα των τραπεζών και των ασφαλίσεων. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει ένα καλό βήμα. Τέλος, με πρωτοβουλία κάποιων συναδέλφων μας έχουμε ξεκινήσει συντονισμό των μυστηριωδών ερευνών ε, των ερευνών για μυστηριώδεις περιπτώσεις. Καλός τρόπος για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές και τελικά για κάθε μία από τις αρχές έχουμε βελτιώσει το μηχανισμό εδώ για την τραπεζική αρχή για να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση του ξεβλήματο μαύρου χρήματο. Ήταν φυσιολογικό και σωστό να έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή για καλύτερο συντονισμό. Στον τομέα των ασφαλίσεων, λάβαμε υπόψη την πραγματικότητα ότι πολύ συχνά υπάρχουν ε, κάποιες ε, ασφαλίσεις ε, που δρούν μέσω επιχειρήσεων που είναι βιτρίνες και δεν σέβονται τα δικαιώματα καταναλωτών σε άλλα κράτη-μέλη. Ε, χαίρομαι που το καταπολεμούμε και αυτό. Και τέλος, η ε, ΕΣΜΑ, η Αρχή Κινητών Αξιών, θα μπορεί να παρέμβει σε προμηθευτές που παρέχουν συγκεκριμένα προϊόντα όσον αφορά τους δείκτες αναφοράς και τα λοιπά και τα άλλα μέσα. Αλλά φυσικά το βασικότερο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν το θέμα της διακυβέρνησης. Εκεί βελτιώσαμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να γίνεται βάση περισσότερων γνώσεων, κυρίω σε περίπτωση συγκρού συμφερόντων. Οι πρόεδροι τη ΕΣΑ θα μπορούν να αποφασίζουν σε περίπτωση δυσκολιών ε, επίτευξη πλειοψηφία θα μπορούν να ακολουθήσουν μια σιωπηρή διαδικασία για τη σύγκληση τη εποπτείας, την ε, ξεκίνημα αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και των προβλήματων αρμοδιότητα μεταξύ ε, εθνικών αρχών σε διασυνοριακέ υποθέσει. Με τον ίδιο τρόπο, οι αρχέ θα υποχρεούνται να θεσπίζουν ομάδε συντονισμού όταν ε, το ζητήσουν πέντε εθνικές αρμόδιες αρχές. Αλλά είμαστε ειλικρινείς και πιστεύω κύριε Αντιπρόεδρε ότι θα αναγκαστείτε να συμφωνήσετε με το δικό μου διαγνωστικό. Διακρίνουμε κάποια υποκρισία εκ μέρους του Συμβουλίου διαρκώς ε, μας λέει πως θέλει να υλοποιήσει αυτή την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών που θα χρηματοδοτήσει τόσο ωραία την πραγματική οικονομία αλλά οπότε θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη διακυβέρνηση γυρνάνε και μας λένε ότι πρέπει οι εποπτικέ αρχές να είναι ελεγχόμενες από τα κράτη-μέλη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ε, σπάσουμε αυτή την προκατάληψη να ξέρουμε ότι πετύχαμε πολλά μέχρι σήμερα, αλλά δεν είναι παρά ένα βήμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Δομπρόφσκης. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η επανεξέταση ε, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας είναι πολύ σημαντικό εγχείρημα ε, είναι σημαντικό να εξευρεθεί συμφωνία ε, σε, αυτό, σε αυτή τη σημαντική δέσμη ε, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της θητείας, πριν από τις διακοπές, μπορεί να προχωρήσει η εργασία και έτσι να υπάρξουν πρόοδοι στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Ε, είναι υψηλή η φιλοδοξία που ε, συνδέουμε με την ε, προσπάθεια αυτή. Το αποτέλεσμα βέβαια δεν θα μπορούσε να καταστεί εφικτό αν δεν υπήρχε η επικοδομητική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο έδειξε κατά τις διαπραγματεύσεις ότι έχει πλήρη επίγνωση του ρόλου του ε, στην επίτευξη της ε, ολοκλήρωση της αγοράς. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους συνεισηγητές και την κυρία Μπερές και τον κύριο Κάρας για το επίτευγμα αυτό, για την εργασία τους και ε, περιμένω να ψηφιστεί. Είναι σημαντικό διότι έτσι υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση ε, των πρακτικών στην Ένωση και αποτελεί και σημαντικό βήμα μπροστά για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος ε, και αυτό ε, ανταποκρίνεται στη φιλόδοξη πρόταση της Κομισιόν του Σεπτεμβρίου του 2018. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα μπορεί έτσι να παίξει καλύτερα το ρόλο της στην καταπολέμηση του ξεπλήματος. Είναι σημαντικό και η σύγκληση των εποπτικών αποτελεσμάτων ε, και αυτό είναι σημαντικό και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για τους επενδυτές. Ε, έτσι θα υπάρξει μια πλήρης κεφαλαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που θα μπορέσει να ωφελήσει την οικονομία, τους καταναλωτές και βέβαια θα προεφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες μέλη. Χαιρετίζω την συμφωνία που επετεύχθη για την προώθηση της σύγκλησης ε, στον τομέα της εποπτείας θα είναι πιο αποτελεσματική η λειτουργία της εποπτείας μετά από αυτήν την ε, ε, επαναξέταση και την αναθεώρηση θα υπάρχει καλύτερη συνεργασία ούτω ώστε να υπάρχουν και ίσοι όροι ανταγωνισμού. Επίσης υπάρχουν περισσότερες ε, αρμοδιότητες ε, στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορών. Ε, χαιρετίζω επίσης τις τρεις αρχές για την προστασία καταναλωτών, την εταιρική διακυβέρνηση και τη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Ε, θα ε, υπάρξει καλύτερη συνεργασία ε, στις αρμόδιες αρχές και οι νομοθέτες θα διατηρήσουν τις, τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται Χαιρετίζω επίσης την συμφωνία της 21ης Μαρτίου ε, για την σύσταση ε, ενός ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου που θα διασφαλίσει την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία θα έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου ε, οι περισσότερες ε, ε, τροπολογίες του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου λαμβάνονται υπόψη στον τριμερή διάλογο και οι διαβουλεύσεις θα γίνουν με πιο ε, σωστό τρόπο. Ε, η ορατότητα του Συμβουλίου θα αναδειχθεί ε, λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου Προέδρου Αντιπροέδρου. Και όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, ο νέος κανονισμός ενισχύει και την προστασία των μαρτυρών δημοσίου συμφέροντος. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο και στη συνάδελφο την Επίτροπο κυρία Γιούροβα. Θεωρούμε <clears throat> απόλυτη προτεραιότητα ε, να ολοκληρωθεί η ε, αγορά, ε, η Ένωση των Αγορών Κεφαλών και η Τραπεζική Ένωση. Αυτό το κείμενο έχει σχέση με τα προβλήματα της καταπολέμησης του ξεπλήματος χρημάτων και άλλα προβλήματα <clears throat> υπό το φως των σοβαρών προβλημάτων που είχαμε αντιμετωπίσει τον τελευταίο καιρό σε σχέση με τράπεζες στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε τον αγώνα κατά του ξεπλήματος και να ε, ενισχύσουμε το ρόλο των υποπτικών αρχών. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που, λύθη, που η πολιτική συμφωνία. Οι καινούργιοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι η πρόληψη και η μείωση του κινδύνου ξεπλήματος χρήματος στον τραπεζικό τομέα θα ε, γίνει, θα επικεντρωθεί, θα συγκεντρωθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιογράφων και Αγορών. Όλες οι αρμόδιες αρχές ε, θα εποπτεύουν αποτελεσματικά και συνεχώς τον κίνδυνο ξεπλήματος χρήματος και θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Όταν γίνεται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, ξεκαθαρίζονται πλέον το θα, το ποιο θα, ξεκαθαρίζεται πλέον το ποιο θα πρέπει να δράσει, προκειμένου η δράση να αναμάνεται αμέσω όταν παραβιάζονται σε εθνικό επίπεδο κανόνε για το ξέπλυμα του χρήματο. Χρειάστηκε πολλή δουλειά για να εξασφαλίσουμε συμφωνία σε αυτό το θέμα και θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ρουμανική Προεδρία για τις προσπάθειές τους. Καταλήξαμε στη συμφωνία πολύ σύντομα Με καθησυχάζει που βλέπω τα τρία θεσμικά όργανα να δρούν ενωμένα για να επιτύχουν ε, αλλαγές σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ. Η κυρία Χίμπνερ, εκ μέρους της ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συναδελφοί, το Ευρωπαϊκό Σύστημα χρηματοπιστωτική Εποπτεία βασίζεται σε μια συγκεκριμένη δομή με πολλά μέλη, εθνικέ τράπεζε, επόπτες και θεσμικά όργανα. Κατά την απόψή μου έχει αποδειχθεί αποτελεσματική πλατφόρμα συντονισμού και κόμβο πληροφόρηση για την παρακολούθηση των κινδύνων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν ανάγκη αναθεώρηση όμω του κανονισμού για να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο που εξελίσσεται και οι πρόσφατες θεσμικές αλλαγές, ειδικότερα όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση και την δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Συμφωνώ με τον Επίτροπο Ντομπρόφσκι. Μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερες αλλαγές, αλλά πιστεύω πραγματικά σημειώσαμε πρόοδο. Ενισχύσαμε τα εργαλεία ελέγχου, τη δημοκρατική λογοδοσία, τη βελτίωση της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας. Όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε τελική ανάλυση αυξάνουν την, τα αποτελέσματα των δράσεων της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ευχαριστώ η κυρία Πιέτη για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές το ενδεχόμενο της κοινή εποπτείας ε, για, τις, ε, για, την ε, Ένωση Κεφαλαίου και τις εποπτικές αρχές. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων. Αν αυτό είναι σημαντικό για μας και αν θέλουμε να μειώσουμε τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, χρειαζόμαστε και κατάλληλη ευρωπαϊκή εποπτεία των διαφόρων ιδρυμάτων. Θέλω να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές που προχώρησαν και έκαναν πολύ σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της Ένωσης αυτής. Όμως θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σωστό σημείο και είναι πολύ ε, δυσάρεστο να βλέπουμε ότι εξακολουθούν κάποια κράτη-μέλη να αντιστέκονται στο ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής ε, ε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις ακόμα σχετικά με την εποπτεία. Η ευρωπαϊκή Τα εθνικά συμφέροντα δεν είναι μόνο εμπόδιο για την Ευρώπη, αλλά είναι ε, και ε, πολύ σημαντική βάση για την ανάπτυξη των εθνών μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήταν σε χειμερία ανάρκη το εγχείρημα αυτό για πολύ καιρό και δεν είχαμε συχνά ευκαιρία να το συζητήσουμε. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους ε, Μπερές και Κάρας. Ε, πρόκειται για σημαντικό βήμα μπροστά ε, προς την κατεύθυνση κοινών κανόνων για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Αυτό συμβάλλει στην καλή λειτουργία των κεφαλαίων αγορών. Αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε ε, πριν δώσουμε περισσότερες ε, αρμοδιότητες στις ρυθμιστικές αρχές είναι τα τοξικά προϊόντα που πρέπει να προλαμβάνονται και θα πρέπει να υπάρχει και ε, συμπερίληψη κανόνων περιβαλλοντικών και κοινωνικών. Αυτό το εγχείρημα μπορεί να ε, μην έχει νόημα αν δεν καταπιαστούμε με το ξέπλυμα του χρήματος με μεγαλύτερη στεναρότητα. Γι' αυτό χαιρετίζω τη δέσμευση της Επιτρόπου Γιούροβα. 20 δις ε, ευρώ χάθηκαν τα, τους τελευταίους μήνες λόγω του ξεπλήματος χρήματος. Οι ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών πρέπει να θέσουν φιλόδοξους στόχους για να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο αυτό φαινόμενο. Ακόμη δεν έχουμε βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ του ευρωπαϊκού και του εθνικού επίπεδου. Βέβαια είναι πολύ λεπτή η γραμμή, αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προχωρήσουν πέρα από το status quo. Ε, το οποίο ήταν συνταγή καταστροφής και αυτό άλλωστε οδήγησε και στην τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση. Πρέπει οι επόπτες να αλλάξουν σημαντικά την οτροπία τους. Ε, αν η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαίων πρόκειται να γίνει πραγματικότητα που θα εξυπηρετήσει τους πάντες. Ευχαριστώ. Ο Μαριάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε ο κύριος κάρας προηγουμένως αναφέρθηκε στην έκθεση την οποία είχε φτιάξει πριν από δύο τρία χρόνια ίσως και πιο πριν για το ρόλο της τρόικας στην ελλάδα και νομίζω ότι αυτή ήταν μια σημαντική έκθεση αλλά τα συμπεράσματα που βγήκαν δεν είχαν κάποιο απτό αποτέλεσμα γιατί η τρόικα συνέχισε την ίδια δουλειά στην ελλάδα και ταυτόχρονα δεν υπήρξε καμία αποζημίωση του ελληνικού λαού για τη ζημιά την οποία υπέστη ζημιά την οποία συνομολόγησε ακόμη και ο κύριος Ντάισεμπλουμ σε ερώτηση που του έκανα που είπε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν στην ελλάδα στην ουσία έσωσαν το ευρώ και τις ξένες τράπεζες και όχι βέβαια τον ελληνικό λαό. είναι σίγουρο ότι χρειάζεται η εποπτεία είναι σίγουρο ότι χρειάζονται μέτρα όπως υπόθηκε από την κομισιόν για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. εκεί βρίσκεται το κλειδί πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις πρακτικές αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατία στην ευρωπαϊκή ένωση αν θέλουμε να λειτουργεί σοβαρά το υποπτικό σύστημα αν θέλουμε πραγματικά να παταχθεί η μάστιγα που είναι το βρώμικο χρήμα. ευχαριστώ. Όπω θα ξέρουν οι Επιτροποί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότεροι τίθενται κατά του εγχειρήματο των κεφαλαγορών. Και αυτό το πράττουν διότι υπάρχουν προβλήματα μέσα στον τραπεζικό τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Επεκτείνεται ο σκιώδης αυτό τομέα ε, και πέρα από τα σύνορα. Αυτό λοιπόν εισάγει ε, απαράδεκτους νέου κινδύνου ε, για τη χρηματοδότηση τη οικονομική σταθερότητα. Αυτή η αναθεώρηση όσον αφορά τουλάχιστον τη δική μας ομάδα οδηγεί στο ότι θα πρέπει να επεκταθούν οι αρχές ε, της εποπτικής αρχής τραπεζών. Είναι απολύτω απαραίτητο. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις αναγνωρίζουμε ότι η αντίδραση ορισμένων κρατών να επεκτείνουν τις ερμοδιότητες του ε, Ευρωπαϊκού ε, Μηχανισμού Διάσωσης είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια οφείλεται στο ότι υπάρχει αντίδραση που οφείλεται στο ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη του να υπάρχει μια γενική επισκόπηση την εποπτεία. Αυτή λοιπόν η μυστικοπάθεια και η έλλειψη της εποπτείας είναι εκείνη η οποία επιτρέπει το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Ως εκ τούτου, εγώ είναι κάτι ε, το οποίο χαιρετίζω, το νέο εγχείρημα. Βέβαια δεν είναι, είναι μακριά από το ιδανικό και θα έπρεπε το σχέδιό μας να είναι πολύ πιο φιλόδοξο. Δεν χρειάζεται απλά να επιτείνουμε την εποπτεία, πρέπει να αυξήσουμε τις, ε, την, ε, τον έλεγχο των περίπλοκων ε, χρηματοπιστωτικών εργαλείων που γίνονται στο σκοτάδι και που θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο της οικονομίας. Ο κύριος Γκίγκολτ, για ένα λεπτό. Αυτή η έκθεση για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής καταδεικνύει τη σημασία που έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μια ισχυρή πρόταση και θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινή υποπτία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την πλειοψηφία των ξεδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών, των φιλελευθέρων και των πρασίνων κατέθεσε και αυτό ισχυρέ προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, κυρίως όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματο και τι βιώσιμε χρηματοπιστωτικέ αγορέ. Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο, αλλά δυστυχώ είναι μια θλιβερή πραγματικότητα το ότι τα κράτη-μέλη όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, ναι μεν ε, βγάζουν πανηγυρικού, ε, αλλά παρόλα αυτά δεν πράττουν τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο οι εσωτερικέ ε, δομέ λήψη αποφάσεων εξακολουθούν να μην είναι επαρκώ ευρωπαϊκέ και για για το λόγο αυτό εξακολουθούμε να έχουμε μακρύ δρόμο να διανύσουμε μέχρι την κεφαλαγορά. Και είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονό ότι η γερμανική κυβέρνηση σε αυτό το εγχείρημα είναι στη λάθο πλευρά. Ο κύριος Τάν για δύο λεπτά. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές είχαν πολλά προβλήματα. Πολύ λίγο προσωπικό, λίγοι πόροι, ε, εθνικός διαχωρισμός ανεπαρκής. Τα κράτη-μέλη θέλουν να διονύσουν αυτή την προβληματική κατάσταση. Γι' αυτό συγχαίρω τον εισηγητή, τους εισηγητές που προσπάθησαν να προασπίσουν το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Μια κοινή Ευρωπαϊκή Υποπτική Αρχή είναι εκ των Ουκάνευ για τι ευρωπαϊκέ κεφαλαίε αγορέ, επιτρέπει να επιμεριστεί ο κίνδυνο και να γίνουν πιο ανθεκτικέ οικονομίες οικονομίε μα. Όπω και για το τραπεζικό πακέτο που συζητήσαμε σήμερα, το πακέτο για τι υποπτικέ αρχέ θα προλάβει τις μελλοντικέ ε, εξελίξεις. Μία από αυτές είναι το Brexit. Σε, ποια, σε ποιο βαθμό το Brexit θα προκαλέσει κούρσα προς τα κάτω. Επίσης, ε, είναι σημαντικό ε, το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να σταθούμε ενωμένοι. Ένα ενιαίο εποπτικό πλαίσιο στην Ευρώπη χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του Brexit, αλλά και τη νέα νομοθεσία για τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά, την καταποτολέμηση του ξεπλήματος του χρήματος, την, ε, χρηματοδότηση της τα κτλ. Για τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά. Γιατί οι εποπτικές αρχές πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο. Υπάρχουν, ε, υπάρχει ο κίνδυνος με τις κλιματικές πολιτικές. Δεν έχουμε κοστολογήσει, τιμολογήσει το κόστος τους. Ούτε οι εταιρείε αξιολόγηση του πιστοτικού κινδύνου το έχουν κοστολογήσει. Θα πρέπει λοιπόν οι εποπτικέ αρχέ να παίξουν καθοριστικό ρόλο και να πιέσουν ούτω ώστε να κοστολογήσουμε το κόστος καταπολέμησης τη κλιματική αλλαγή, ούτω ώστε ο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έτοιμο. Συγχαίρω τους συζητητές ε, που πέτυχαν συμφωνία που αντιμετωπίζει αυτές τις μελλοντικέ προκλήσεις μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες ε, συγκυρίες. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τους ομιλητές εδώ. Ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης έχει το λόγο. Αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση και τις θέσεις που πήρατε. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο φιλόδοξο, όπως είπα, όσο θα θέλατε ορισμένοι από εσάς. Είμαι πεπισμένο ότι αυτή η πολιτική συμφωνία όμω θα μα επιτρέψει να επιτρέψουμε μεγαλύτερη υποπτική σύγκληση στο μέλλον. Είναι βασικό σταθμό σε μια πραγματική ε, ένωση κεφαλαίων Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Μπερέ και τον κύριο Καρά, του δύο εισηγητέ. Και θα ήθελα να στηρίξετε το αποτέλεσμα με την αυριανή σας ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κάρας έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους Ευρωπαίους πολίτες που ενδεχομένως να μας παρακολουθούν ότι αυτή η τελευταία εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τι σημαίνει. Σημαίνει σήμερα μόνο είχαμε 13 διαφορετικές εκθέσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και αυτές οι εκθέσεις θα ψηφιστούν αύριο. Ξεκινήσαμε λοιπόν πριν από 8 χρόνια τότε που υπήρξε για πρώτη φορά η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Αρχίσαμε τότε να αντιδρούμε και αύριο λοιπόν θα αποφασίσουμε με τις ε, τρεις αυτές εκθέσεις να δρομολογήσουμε μια ευρεία αναθεώρηση έτσι ώστε αυτό το σύστημα να γίνει πιο ελπιδοφόρο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης ε, της Ένωσης Κεφαλαίου και προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής είναι λοιπόν ε, ευχάριστη είδηση για του Ευρωπαίους ε, πολίτες το ότι η πραγματική οικονομία, οι θέσει απασχόληση, η ανάπτυξη στην Ευρώπη μπορούν να προχωρήσουν και όλα αυτά καταδεικνύουν ότι είμαστε και σε θέση να αντιδράσουμε, ότι αναζητάμε λύσεις και αυτό το πράττουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή θέλω να πω ότι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προύκατ Βάλτς, τον προκάτοχό μου, από τον οποίο ανέλαβα αυτήν την έκθεση και την ε, ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ όλους σας και για την ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία. Η κυρία Πέρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων για το χρόνο και το ύφος που υιοθέτησαν στη συζήτηση. Όλοι οι συνάδελφοι, ανεξάρτητα το από τη θέση τους, από το που κάθονται σε αυτό το ημικύκλιο, σε αυτή την ολομέλεια, ε, συμφωνούν με, την, με τους εισηγητές. Εμείς θέλαμε να πάμε πιο μακριά. Ε, αλλά τελικά ε, προσκούσαμε στον τοίχο του Συμβουλίου. Στο Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ακούω περίεργα επιχειρηματά, απίστευτα. Όταν έχουμε μια διασυνοριακή ας δραστηριότητα, αν εκδίδεται ας πούμε δελτία ή αν ε, η ασφαλιστική σας εταιρεία είναι μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, τότε η αρμόδια εθνική αρχή, λόγω της γειτονία και της επικουρικότητας, αυτή αξιολογεί τους κινδύνους. Είναι λάθος αυτό εκ μέρους του Συμβουλίου. Ε, καταφέραμε μαζί με τον Νότμαρ Κάρας ε, να πετύχουμε τελευταία στιγμή αυτή την συμφωνία σε ό,τι αφορά το δελτίο ε, σε ό,τι αφορά το εσωτερικό μοντέλο που δεν θα πρέπει να είναι μόνο υπό την αιγίδα μίας ε, εσωτερικής αρχής. Σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες ε, ασχολούμαστε και με τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης ή με, τους, με τα καταθετήρια χωρίς πολλούς τίτλους πρώτων πυλών είναι οι ευρωεκλογέ. Και οι πολίτες μας καταλαβαίνουν όταν, όταν ψάχνουν το ευρωπαϊκό πνεύμα, όταν ψάχνουν αυτή τη δυνατότητα να βρίσκουμε μαζί ευρωπαϊκές κοινέ λύσεις, γιατί αντιμετωπίζουμε και όλοι μας την ίδια αγορά, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, κάνουμε μια δουλειά πραγματικά πάρα πολύ έντονη υπό την αιγίδα της Κομισιόν ε, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προς το συμφέρον των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ, Βρες, Ψηφίζουμε βεβαίως αύριο και περνούμε στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης και είναι η συζήτηση για την πολιτική εποπτεία επενδυτικών εταιριών. Ο κ. Φέρμπερ ως εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε θέσει ως στόχο μια ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών ε, που προσανατολίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου. Δηλαδή η ε, ρύθμιση θα πρέπει να είναι στοχευμένη. Παρόλα αυτά όμως ε, έχουμε τις επενδυτικές εταιρείε, τις οποίες τις ρυθμίζουμε εδώ και καιρό ως να ήταν τράπεζες. Όμως οι επενδυτικές εταιρείε έχουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο διαφέρει κατά πολύ από αυτό των τραπεζών και επίσης οι επενδυτικές εταιρείε ε, χειρίζονται και θέματα που είναι συνδεμένα με κινδύνους. Ως εκ τούτου οι επενδυτικές εταιρείε θεωρούμε ότι δεν ήταν σωστά ρυθμισμένες. Τώρα το νέο εποπτικό πλαίσιο έχει ως στόχο να ρυθμίσει αυτό το γεγονός. Εγώ ως εισηγητής θεώρησα ότι είναι σημαντικό γι' αυτό το καθήκον να θεσπίσουμε ένα αρκετά σοβαρό, σταθερό πλαίσιο και αυτό σημαίνει σε αντίθεση με τους συναδέλφου και από κάποια κρατημέλη εμείς δεν θέλουμε μόνο να υιοθετήσουμε με τους νέους κανόνες από τη δέσμη μέτρων για τις τράπεζες, αλλά να έχουμε ένα πιο λογικό πλαίσιο για τις επενδυτικές στηρίες. Αυτό ήταν ο στόχος και τον επιτύχαμε. Υπάρχουν λοιπόν τρεις ε, κατηγορίες επενδυτικών εταιριών στο μέλλον. Ε, το καθεστώς ε, θα ρυθμίζεται με βάση το μέγεθος. Υπάρχουν λοιπόν τρεις κατηγορίες μεγάλες επενδυτικές εταιρείε, οι οποίες εξακολουθούν να ελέγχονται από την Τραπεζική Υποπτική Αρχή. Οι μεσαίες εταιρείε, οι οποίες ε, υπάγονται στις ρυθμίσεις ε, για την κέφαλα αγορά και υπάγονται και σε κάποιους κανόνες οι οποίοι είναι καθοριστικοί για τέτοιου είδους εταιρείε και αξιολογούν τους κινδύνους. Και τέλος έχουμε τις μικρές επενδυτικές εταιρείε, οι οποίες έχουν ένα μικρό προφίλ κινδύνου και ως εκ τούτου αυτές δεν υπάγονται στο ίδιο αυστηρό καθεστώς. Αυτή λοιπόν η βαθμινόμηση, η ταξινόμηση μάλλον σε τρεις, ε, σε κατηγορίες είναι και η ουσία αυτής της νέας ρύθμισης. Λαμβάνει υπόψη της αυτή η νέα ρύθμιση και όλα εκείνα τα οποία εξετάσαμε όταν θελήσαμε να ρυθμίσουμε τις τράπεζες. Αυτό το νέο πλαίσιο για τις επενδυτικές εταιρείε είναι όχι μόνο πιο αναλογικό, είναι και πιο σταθερό. Κυρίως έχοντας κατά νου ε, το καθεστώς που επικρατεί σε τρίτες χώρες. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά κατά νου, ε, ξέρετε ότι ε, υπάρχει το ενδεχόμενο της αποχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίω αυτό έχει αναβληθεί για δύο φορές. Παίζει όμως ρόλο η αποχώρηση της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί σε τελική ανάλυση οι περισσότερες επενδυτικές εταιρείε είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, άρα δηλαδή σε ένα μελλοντικό τρίτο κράτος. Με αυτή τη νέα ρύθμιση διασφαλίζουμε οι βρετανικές επενδυτικές εταιρείε μετά το Brexit να υπάγονται σε ένα πολύ αυστηρό καθεστώς εφόσον επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διευρύνει τον κατάλογο των κριτηρίων αναλογικότητας. Οι ε, λογοδοσία έναντι των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών έχει ενισχυθεί, το ίδιο και έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν πρόκειται πάλι για ε, ρυθμίσεις αναλογικότητας. Με τον τρόπο αυτό έχουμε καθορίσει ένα αυστηρό πλαίσιο, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε τις επενδυτικές εταιρείε. Παράλληλα, η υποχρέωση λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι του Κοινοβουλίου έχει ενισχυθεί, άρα δηλαδή θα ενημερωνόμεθα για αυτά που πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως εκ τούτου, αυτό το νέο σχέδιο είναι ένα σημαντικό βήμα για να αντιμετωπίσουμε και το ενδεχόμενο αποχώρηση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή και αυστηρή ρύθμιση. Σε γενικέ γραμμέ πιστεύω ότι καταλήξαμε σε έναν καλό συμβιβασμό και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την καλή και αγαστή συνεργασία με όλου του σκιώδει ηγητέ από τι διάφορε πολιτικέ ομάδε. Να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου και βεβαίω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επικοδομητική τη στάση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον Αντιπρόεδρο τον κύριο Ντομπρόφσκης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα πρώτον να ευχαριστήσω τον κύριο Φέρμπερ για το έργο του, για την αναθεώρηση δηλαδή τον κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσει προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων. Σημαντικό μέτρο για την αγορά μα. Είχαμε κανόνε για επιχειρήσει οι κατά μείζωνα λόγο είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν στην Ένωση και να προαγάγουμε τις ε, αγορές κεφαλαίων. Ο κανονισμός επίση διασφαλίζει ότι οι συστημικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν μαζί με τις τράπεζες. Οι μεγαλύτερε από αυτές ε, υπάγονται πλέον στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας στο πλαίσιο της ενιαίας τραπεζικής αγοράς για να υπάρχουν ίσοι ίδιοι κανόνες για τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Εισάγουμε και μερικές αλλαγές σχετικά με τις επιχειρήσεις τρίτων χωρών και το πώς παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική οδηγία και τον κανονισμό. Οι αγορές μας παραμένουν ανοιχτές επιχειρήσεις τρίτων χωρών, διασφαλίζοντας διαφάνεια και διασφαλίσεις για τις επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές υπηρεσίες, όπως είπα, στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μεγάλη βεβαίω κλίμακα. Η ΕΣΜΑ ε, επίσης έχει περισσότερες δυνατότητες εποπτείας επί επιχειρήσεων τρίτων χωρών. Μέσα με τον κύριο Φέρμπερ καταλήξαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Η υποστήριξη του Κοινοβουλίου που την συνένεση ε, Ευχαριστώ επίσης και τους κοιόδης εισηγητές. Νομίζω πετύχαμε τους στόχους μας, τους φιλόδοξους στόχους μας σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στην λογική προσέγγιση που υιοθέτησε το Κοινοβουλίο. Κομισιόν από εδώ και πέρα θα κάνω την πορεία για την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Θα προχωρήσει ταχύτατα για να διασφαλίσει ότι τα ωφέλη των αλλαγών των, στις ευρωπαϊκές κεφαλαιογορές θα έχουν εφαρμογή για όλους. Πρώτα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντελβό, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ κατά πρώτον τον κύριο Φέρμπερτ, τον εισηγητή για την οργάνωση των εργασιών για το πώς υπεραμείνθηκε των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο. Καταλήξαμε λοιπόν σε έναν καλό κανονισμό. Αυτό θέλαμε, αυτό περιμέναμε. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δραστηριότητες και τους κινδύνους διαφόρων επιχειρήσεων επενδύσεων. Το νομοθέτημα επίσης ασχολείται με κάποιες εθνικές εξαιρέσεις για επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καμία επιτήρηση για κανέναν κανόνα. Η πρόκληση ήταν να συγκεράσουμε τους 11 διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων σε τρει ή κατηγορίε. Κατηγορία 1 που περιλαμβάνει τι μεγαλύτερε επιχειρήσει που έχουν, θα έλεγα, συστημική διάσταση και που υπόκεινται στη νομοθεσία περί τραπεζών. Στην κατηγορία 2, εδώ έχουμε 6.000 επιχειρήσεις, μεγαλύτερη κατηγορία. Εδώ κίνδυνο υπολογίζεται με βάση του γνωστού παράγοντε Κ. Και τρίτον, κατηγορία 3, έχουμε τι μη συνδεδεμένε επιχειρήσει, μικρέ επιχειρήσει μικρού κινδύνου που υπόκεινται σε μειωμένες απαιτήσεις υποπτίας. Καταλήξαμε λοιπόν σε ένα συμβασμό, συγκεράσαμε τις απαιτήσει και των τριών κατηγοριών για τα ίδια κεφάλαια που πρέπει να εγγυώνουν την σταθερότητα. Λέβαμε υπόψη μας επίσης τους κανόνες διακυβέρνησης που αφορούν πάρα πολλέ επιχειρήσει που πρέπει να έχουν επιτροπή διαχείριση κινδύνου και επιτροπή αμοιβών, πολύ σημαντικέ επιτροπέ. Οι επιτροπέ αυτέ πρέπει να αποτελούνται από άντρες και γυναίκες σε ίσα ποσοστά. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εκεί γίνεται και λόγος για τι αμοιβέ που πρέπει να είναι ίσε για άντρες και γυναίκες. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τον κανόνα σύμφωνα με τον οποίο δεν πρέπει να περισχύει η αρχή του βραχυπρόθεσμου κέρδους. Και επίσης χαιρετίζω και τα κριτήρια τα οποία ορίσαμε για τις ισοτιμίες και τον αυξημένο ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην ρύθμιση των επιχειρήσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. δεν είναι εδώ, άρα περνάμε στο Κατσουδιά και δίνω τον λόγο αμέσως στον κύριο Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στο γαλλικό λαό για το πλήγμα το οποίο υπέστη και η Γαλλία και βέβαια όλη η ανθρωπότητα με την καταστροφή η οποία έχει διαμορφωθεί από την πυρκαγιά στην ε, Παναγία των Παρισίων. Ένα μνημείο το οποίο είναι μνημείο ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Η συζήτηση που κάνουμε σήμερα για την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων είναι σημαντική διότι μπαίνει μια τάξη στο θέμα αυτό λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε να υπάρχει εποπτεία εποπτεία στις ιδιαίτερα μεγάλες ε, επιχειρήσεις επενδύσεων οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν και συστημικό κίνδυνο και ορθώς εφαρμόζονται εκεί κανόνες που έχουν σχέση και μοιάζουν θα έλεγε κανείς το μεγαλύτερο μέρος τους με τους κανόνες που αφορούν τον τραπεζικό έλεγχο. στις μεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει μια ιδιαίτερη ρύθμιση και φυσικά στις μικρότερες όπου νομίζω ότι εκεί ορθώς λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα. αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το brexit διότι οι περισσότερες επιχειρήσεις τέτοιου τύπου είναι εγκατεστημένες στο λονδίνο. εδώ χρειάζεται ρύθμιση και προσοχή στο θέμα αυτό. ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και για τις διαφορετικές σκοπιές που αναδείξατε. Η συζήτηση δείχνει ότι η μεταρρύθμιση είναι πρόσδεκτη. Μεγαλύτερη αναλογικότητα θα βοηθήσει τις επενδυτικές εταιρείε να δραστηριοποιηθούν ε, προς το συμφέρον το δικό τους, ε, των οικοκυριών και της δραστηριότητάς τους. Το να κρατήσουμε κάποιες μαζί με τις τράπεζες έχει νόημα. Ε, λόγω του επιχειρηματικού μοντέλου και του κινδύνου που ενέχουν. Επίσης, ε, εξασφαλίζουμε και ισοτιμία για τις επενδυτικές ε, εταιρείε της Ένωσης. Γιατί δεν θα θέλει η Ένωση για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών να βασίζεται σε ξένες επιχειρήσεις, ειδικά εν ώψη του Brexit. Ε, κατέγραψα διάφορες παρατηρήσεις σας για τις αλλαγές που εξετάζουμε. Το νέο καθεστώς προβλέπει ε, σωστή εφαρμογή και μια βαθμία εφαρμογή και αναθεώρηση σε κάποια χρόνια. Βασίζομαι στην υποστήριξή σας, ούτως ώστε ε, η διάταξη αυτή, οι διατάξη αυτές μάλλον, να εξυπηρετούν το στόχο. Ο εισηγητής, ο κ. Φέρμπερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ένα πολύ θερμό ευχαριστώ σε αυτούς που ήταν θαραλέοι και συμμετείχαν στη συζήτηση. Ε, Βεβαίω, αγαπητοί Μέντι, θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν είχαμε παρόντες ε, περισσότερους και οτσιγητές και αν είχαμε εδώ και άλλους συναδέλφους, αν είχαν βρει το χρόνο να έρθουν. Με πάση περιπτώσει, ευχαριστώ θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να σας πω το εξή. Ε, σήμερα η ΕΚΟΝ έχει καταθέσει πάρα πολλές εκθέσεις. Αυτές οι εκθέσεις θα ψηφιστούν αύριο και με τον τρόπο αυτό δημιουργούν δημιουργούμε ένα πλαίσιο που είναι του επίπεδου μας, που πραγματικά είναι πολύ ικανοποιητικό. Λυπάμαι πάρα πολύ για το ότι εκτός από τους ε, λίγους ε, που ασχολήθηκαν ουσιαστικά με το θέμα, η κοινή γνώμη δεν ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για τα δικά μας θέματα, όμως εμείς μπορέσαμε να προλάβουμε κρίσεις, η Ευρώπη ε, σε περίπτωση κρίσης θα είναι πιο σταθερή, αλλά βλέπετε αυτά δεν προκαλούν το ενδιαφέρον. Συμβαίνει αυτό συχνά όταν τα θέματα είναι τεχνικά, όπου πρέπει κανείς να ασχοληθεί με λεπτομέρειες, όπου πρέπει να εμβαθύνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις ε, τα θέματά μας δεν εμφανίζονται στους επιχαίους ε, τίτλους των εφημερίδων. Όταν όμως τα πράγματα πάνε στραβά, τότε βεβαίως αυτά ε, εμφανίζονται πολύ περισσότερο. Ίσως ε, δεν ξέρω αν κάτι ξεχάσαμε, αν κάτι δεν ρυθμίσαμε, ενδεχομένως να δημιουργηθούν, ε, να προκληθούν διαμαρτυρίες και πρέπει να σας πω με χαρά θα το περιμένω αυτό. Με χαρά θα περιμένω τις επενδυτικές εταιρείε που θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Πάντως εγώ να σας πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι για όλα αυτά που επιτύχαμε σε αυτή τη θητεία στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Πετύχαμε πάρα πολλά, clearing houses, ε, τα παράγωγα, τις εποπτικές δομές, τις επενδυτικές εταιρείε σε όλους αυτούς τους τομείς επιτύχαμε πολλά έτσι ώστε να κάνουμε τις αγορές μας πιο σταθερές. Και ελπίζω τουλάχιστον κάποιοι να το κατανοούν αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φέρμπερ, η κοινή μας συζήτηση τελείωσε και θα ψηφίσουμε αύριο για το θέμα αυτό. Προχωρούμε στη συζήτηση του επόμενου σημείου, δήλωση της Κομισιόν για τη μη θέσπιση ενωσιακού φόρου ψηφιακών υπηρεσιών να ενημερώσω τους βουλευτέ ότι για αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει catch the eye, ούτε μπλε κάρτα γίνεται αποδεκτή. Απλώς έχουμε ένα γύρο ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες και τίποτα άλλο. Πρώτος ομιλητής από την ε, Επιτροπή, ο Αντιπρόεδρος κ. Ντεμπρόφσκης. Παρακαλώ ακόμα μια φορά έχει το λόγο. Ευχαριστώ ξανά, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Σας ευχαριστώ που οργανώσατε τη συζήτηση για να μιλήσουμε για την ε, φορολογία των ψηφιακών δραστηριοτήτων και των φόρων ψηφιακών υπηρεσιών, όπου δεν υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο. Για την ψηφιακή φορολόγηση. Ξέρω ότι θέλατε την πρότασή μα, ήσασταν υπέρμαχοι και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω να ξεκινήσω την παρέμβασή μου ε, υπενθυμίζοντας γιατί η Κομισιόν παρουσίασε μια πρωτοβουλία με αυτό το θέμα στις 21 Μαρτίου του 2018. Το κάναμε γιατί υπάρχουν διάφοροι λόγοι οι οποίοι υπάρχουν ακόμα και σήμερα και το πρόβλημα δεν έχει επιληθεί. Αυτό μην το ξεχνάμε όταν θα εγγύψουμε του θέμα του επόμενου μήνες, που είναι απλό. Οι διεθνεί ε, κανόνες για την ε, εταιρική φορολόγηση δεν προσαρμόζονται στην μοντέρνα οικονομία. Δεν ε, φορολογούν τα κέρδη μιας ψηφιακή εταιρεία όταν υπάρχει φυσική παρουσία στην χώρα. Με βάση τα του φορολογικού κανόνε δεν μπορούμε να φορολογήσουμε αυτέ τι δραστηριότητε. Ε, τα κέρδη από κάποιε δραστηριότητε ψηφιακέ δεν φορολογούνται ή βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μακάτε, ελάχιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μα ε, υποσκάπτεται, ε, ο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά και τα θεμέλια τη φορολογική δικαιοσύνη επίση τίθενται ένα αμφιβόλο. Γι' αυτό ακριβώ θέλουμε δίκαιη ε, φορολόγηση τη ψηφιακή οικονομία. Ε, Καταρχά, μια διαρθρωμένη πρόταση για να μεταρρυθμίσουμε του κανόνε για την ε, εταιρική φορολόγηση, ούτω ώστε να καταχωρούνται τα κέρδη και να φορολογούνται ε, όταν ε, διαπιτράει η εταιρεία με του ε, χρήστε μέσω των ψηφιακών καναλιών. Μια πλήρη λύση. Μια πιο στοχευμένη πρόταση επίση, κάτι που ζήτησαν κρατημέλη για προσωρινό φόρο για τι βασικέ ε, ψηφιακέ δραστηριότητε που σήμερα δεν φορολογούνται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Είναι μια ενδιάμεση έκθεση, ε, λύση ε, μέχρι να βρούμε την οριστική λύση. Όπω ξέρετε, οι συζητήσει στο Συμβούλιο εστιάσαν κυρίω σε αυτή την ενδιάμεση λύση και βεβαίω είμαστε απογοητευμένοι που τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε ομόφωνη συμφωνία για μια πρόταση για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών που ήταν υπέρ αυτή τη ιδέα. Ε, δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε ομόφωνη συμφωνία και αυτό εξηγείται από τον κανόνα τη ομοφωνία, σύμφωνα με τον οποίο το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα για προτάσει για θέματα φορολογικά. Όπω εξήγησα στην ανακοίνωση φέτο για την, ε, τον τρόπο φορολόγηση, ε, είναι ακόμα μία πρωτοβουλία για τα φορολογικά, όπου ε, ο κανόνας για την ομοφωνία παρεμποδίζει την πρόοδο ε, για να ενισχύσουμε την ενιαία αγορά και να αποφύγουμε τον καταγερματισμό της. Ε, μια πιο μοντέρνα Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να προχωρήσει εάν δεν φορολογήσουμε σωστά με βάση μοντέρνους κανόνες για την ψηφοφορία οι περίπλοκες εργασίες που μας οδήγησαν ε, στο συμβιβασμό για το φόρο ψηφιακών υπηρεσιών ε, ελπίζω να μην είναι ισμάτιν. Καταρχάς θέλουμε ένα πλαίσιο για τα κράτη-μέλη τα οποία θα αποφασίσουν να υιοθετήσουν την ενδιάμεση λύση σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, θα μπορέσουμε να επανεξετάσουμε την πρόταση ε, που είναι στο τραπέζι του Συμβουλίου μέχρι Εάν ε, ο κανόνας ε, που είναι στο τραπέζι του ΩΣΑ δεν ε, ευοδοθεί μέχρι το 2020 για το CCTB. Επίσης, θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς συνομιλίες στο G20 και στον ΩΣΑ για παγκόσμια λύση. Η ενδιάμεση έκθεση του ΩΣΑ για μια μακροπρόθεσμη λύση για τις φορολογικές προκλήσεις που απορρέει από την ψηφιοποίηση της οικονομίας Είναι το βασικό μας κείμενο. Πρέπει να φορολογήσουμε την, σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύουμε, την ψηφιακή οικονομία. Ε, οι Υπουργοί Οικονομικών ε, του G20 συζήτησαν και θα συνεχίσουν να συζητάνε αυτό το θέμα. Ε, είναι σημαντικό να συζητάμε με την εθνική κοινότητα και να συντονιζόμαστε στα πλαίσια του ΩΣΑ. Εάν μιλήσουμε με μία φωνή ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση προς το συμφέρον μας. Είναι σημαντικό οι προσπάθειές μας ε, για τον εξυγχρονισμό των φορολογικών ε, εταιρικών κανόνων ε, να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος και να μην δημιουργήσουν νέες, νέες τρώσεις περιπλοκότητας. Θέλουμε ένα απλό σύστημα κατάλληλο για το μέλλον. Δεν θα πρέπει να το αγγίξουμε το σύστημα, θα πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε εκ βάθρων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 Θα μιλήσω Ολλανδικά, κυρία Πρόεδρε. Πολλοί ζουν την κρίση. Βλέπουν τους μισθούς τους να μειώνονται. Πιέζουν από την φορολογία. Δεν είναι δείγμα κινησμού η Apple, η Google, η Amazon, η Facebook και λοιπά. είναι εταιρείε, οι επιχειρήσει οι πληρώνουν λιγότερα από όλου εν τέλει. στη Γερμανία, στην Ελβετία, στη Σουηδία και σε πολλές άλλες χώρες, ο κόσμος διερωτάται κάτι δεν πάει καλά. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν φορολογούνται παρκώς. Αυτή είναι μερική μόνο από τους λόγους τους οποίους ο κανόνας της ομοφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα φορολογικά πρέπει να αναθεωρηθεί. Οι σοσιαλιστές ε, δημοκράτες έχουν υποβάλει συνεφώς πρόταση. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια διαπραγμάτευση γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ αλλαγές στον χώρο της φορολογίας. Οι φόροι εφευρέθηκαν πολύ πριν την ε, ψηφιοποίηση, πριν την ψηφιακή οικονομία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι πλέον. Όχι μόνο να εισαγάγουμε έναν ελάχιστο φόρο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δρομολογήσουμε μια εκβάθρον αναθεώρηση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε την αποψή του και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, δύο τρίτων και κάτι περισσότερο. Έτσι, πλέον τα κράτη-μέλη είναι καιρός να αρχίσουν να εξετάζουν σοβαρά την θέσπιση ενό φόρου για τι ψηφιακέ υπηρεσίε. Γερμανία, Γαλλία και πολλέ άλλε χώρε. Καλό και τι άλλε χώρε να εξετάσουν σοβαρά την πρότασή μα και να στείλουν το σωστό μήνυμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Σήμερα οι διαπραγματεύσει πρέπει κάπω να καταλήξουν έτσι ώστε οι μεγάλες επιχειρήσεις, τεράστιε επιχειρήσει, να συνεισφέρουν και αυτέ. Στα σχολεία, στα νοσοκομεία, Όλοι λοιπόν να συνεισφέρουν και βεβαίω σίγουρα και οι μεγάλε πολυεθνικέ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εκ μέρου ε, τη ΓΟΥ, κύριο Σίντουαν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η φορολογική συμπεριφορά των εταιριών του διαδικτύου των γιγάντων είναι γνωστή. Η Apple το 2014 πληρώσε 50 ευρώ για κάθε εκατομμύριο κέρδου. Και η Netflix και η Amazon το έχουν τελείω ξεπεράσει. Δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα σέντ ε, φόρο στι ΗΠΑ και η Amazon όχι μόνο αυτό, αλλά στην Amazon και 109 εκατομμύρια. Είχε δηλαδή αρνητική φορολόγηση και εντωμεταξύ είχε προσποριστεί 11 δις. Ποιος θα τα καταλάβει όλα αυτά. Δυστυχώς όλα αυτά ε, ίσως είναι και ενδεικτικά για το ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει καμία συμφωνία για την ψηφιακή φορολόγηση. Προσπαθήσαμε κατά τον 21ο αιώνα να έχουμε ενιαία φορολόγηση, δεν τα καταφέραμε και στην προσπάθειά μας αυτή δεν πρόκειται πουδενού για δαιμονοποίηση του διαδικτύου όπως είχε ισχυριστεί ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών κ. Σόλτς. Όχι, πρόκειται για ε, δικαιοσύνη, ε, για άρση των αδικιών νομίζω ότι αυτό περιμένουν οι άνθρωποι από εμά, δηλαδή οι εταιρείε να φορολογούνται ανάλογα με τα κέρδη του. Ο κύριο ε, Γκίγκολτ έχει το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Εκ των Πρασίνων. Κυρία Πρόεδρε, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι το πολύ λυπηρό. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λειτουργήσαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόρθωσε να Άρη ή να θίξει το θέμα της αδικίας. Το ίδιο έπραξε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν στο Κοινοβούλιο διαμορφώθηκε μια ευρύτατη πλειοψηφία. Κατ' ουσίαν όλοι ήταν υπέρ μια σοβαρή φορολόγηση των ψηφιακών εταιριών. Όλα αυτά απέτυχαν στο Συμβούλιο. Και γιατί απέτυχαν, διότι ορισμένη φορολογική παράδοση και ορισμένε ευρωσκεπτικιστικέ χώρε, υποστηριζόμενε από τη Γερμανία, αυτέ όλε οι χώρε οδήγησαν τον Κύριε σε αποτυχία. Και αν ο κύριος Σόλτς πιστεύει ότι μπορεί να καθησυχάσει τον κύριο Τραμπ αρνούμενο σε ευρωπαϊκή λύση και παραπέμποντας τον θέμα στον ΩΣΑ, αυτό είναι λάθος. Αυτό το θέμα θα πρέπει να το δουν πολύ προσεκτικά όλοι οι πολίτες. Ο μεγάλος συνασπισμό στη Γερμανία φταίει φέρει ευθύνη για το ότι δεν επιβλήθηκε η ψηφιακή φορολόγηση και ελπίζω όταν οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν το τι θα ψηφίσουν να το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη τους. Πρόεδρος, το βλέπω, έχουμε προεκλογική εκστρατεία. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Ζόσκερνετς. Χαίρομαι που απέτυχε αυτή η κατάλληλα καλή ιδέα. Γιατί κάποιοι σπαταλούν τα λεφτά των φορολογουμένων. Κάθε τέτοια αποτυχία είναι νίκη για τους φορολογουμένους. Ένα δίκαιο σύστημα φορολόγηση είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να κρατούν τα χρήματά τους αντί να σπαταλώνται. Αφήστε λοιπόν τα χρήματα στα χέρια αυτών που τα κέρδισαν γιατί αυτοί ξέρουν κάτι ε, να κάνουν καλά. Και όταν λέτε ότι δεν έχουμε χρήματα για νοσοκομεία και σχολεία, σταματήστε τα Erasmus Plus για να βρείτε χρήματα που χρειάζεται για τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Σταματήστε να ξοδεύετε σε τρίτες χώρες ανά τον κόσμο. Σταματήστε να σπαταλάτε τα χρήματα και θα βρείτε τα χρήματα που σας λείπουν. Ο Επίτροπος παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για, την, ε, τον ενθουσιασμό που δείξατε στη συζήτηση αυτή. Λυπούμεθα που δεν επετεύχθη ομοφωνία βεβαίω για τον φόρο αυτόν στο Συμβούλιο. Βεβαίω ε, η δουλειά που έγινε δεν πάει χαμένη. Έχουμε ένα πλαίσιο στο πλαίσιο της οποίας θα κοιτάξουμε να, κάνουμε, να πρόοδο στο μέλλον. Εάν δεν καταλήξουμε σε παγκόσμια λύση στον ΩΣΑ θα παρέλθουμε στα της Ένωσης. Χαίρομαι ότι φτάσαμε κοντά σε ένα συμβασμό όσον αφορά και τον παγκόσμιο φόρο για τις ψηφιακές υπηρεσίε. Η συζήτηση για την αναθεώρηση του φόρου για τις επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Η συμμετοχή επίσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΩΣΑ και στο G20 θα πρέπει να είναι πιο συντονισμένη. Η πρόκληση από εδώ και πέρα είναι διτή. Πρώτον, πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μας και δεύτερον να εξασφαλίσουμε ισότιμη κατανομή των φορολογικών βαρών. Πετύχαμε πολλά μαζί πάνω στο θέμα αυτό, γνωρίζουμε όμως ότι δεν φτάσαμε στο τέλος. Πιστεύουμε επίσης ότι το φρένο που έθεσαν κάποια κράτη-μέλη πρέπει να αποτελέσει συναγερμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε δηλαδή σε ψηφορίε επί των φορολογικών θεμάτων με βάση τον κανόνα τη ειδική πλειοψηφία για να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια ρύθμιση τη φορολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε πίτροπε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι οι παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ δεν είναι παρούσα, ο κύριος Βίνκλερ είναι παρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την... ως επεισόδιο στην Ρουμανία. Ο δήμαρχος του Κορών ενμετώπισε πρόστιμο διότι έγραψε το όνομα ενός κτηρίου στα Ουγγρικά και όχι μόνο στα Ρουμανικά. Προκλήθηκε γενικότερη αναστάτωση και οργή. Θυμίζω τις Ευρωπαϊκές Αρχές είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει όχι μόνο στον νόμο, αλλά και εκθέτει τη Ρουμανία διεθνώς. Αφήστε που προκαλεί ένταση, η εμπιστοσύνη καταραίει, είναι πρόκληση για το κράτος δικαίου. Πρέπει να προστρέψουμε στη Ρουμανία τόσο τις μειονότητε όσο και όλου τους άλλου. Τα τιμωρητικά μέτρα δεν βοηθούν κανέναν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. επόμενο ομιλητή, ο κύριο Μπουζόη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωβαρόμετρο ε, λέει ότι θα έχει σημειωθεί πρόοδο σε, σε αυτή την θητεία. Ε, ε σχετικά με την τομοθεσία για, τα, για τις ιατρικές συσκευές και έχουμε προετοιμάσει την ε, μεγαλύτερη δυνατή έρευνα που μπορούσε να παίξει να υπάρξει. Ο καρκίνος ε, των παιδιών είναι ένα θέμα το οποίο θα ερευνήσουμε. Μας ε, ενδιαφέρει ε, να εξετάσουμε το θέμα της υγείας στο μέλλον. Επιθυμούμε να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι στο μέλλον. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τον καρκίνο, να άρουμε τις ανισότητες, να καλύψουμε τα κενά στα νοσοκομεία, να προάγουμε την καινοτομία, κυρίως όσον αφορά τα ιατρικά σκευάσματα και να προετοιμαστούμε για την ε, ψηφιακή επανάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Πόξορ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Ευρώπη και στην Ουκρανία όμως ε, θα γίνουν εκλογές και αυτό θα καθορίσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Ε, αυτό όμω που έχει σημασία και για την Ευρώπη είναι οι μειονότητες. Μετά την πεντηκοστή στην Ουκρανία θα έχουμε τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Ε, ξέρετε, έχουμε ελπίδες ε, στην Ουκρανία και ελπίζω αυτή τη φορά να εκλεγεί ο ΙΗ πρόεδρος με δημοκρατικό τρόπο και να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη. Ελπίζω η Ουκρανία να έχει έναν ή μία πρόεδρο ε, που δεν θα στηρίζουν ε, μια κοινωνία δύο κατηγοριών πολιτών, αλλά θα έχουν κατά νου τα κεκτημένα δικαιώματα. Οι εθνοτικές εντάσεις ε, θέλω να ελπίζω ότι θα εξαφανιστούν, δεν θα υποδαβλίζεται το μίσος και επίσης θα εξοβελιστούν οι ακραίες θέσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι θα προστατεύονται τα δικαιώματα των Ουκρανών στην Ουκρανία. τελευταία Ολομέλεια 2014-2019 ξανασυζητάμε το Brexit. Μία τελευταία παράταση τους δόθηκε, τελευταία στιγμή, λίγο πριν ε, εκπνεύσουν. Η Βουλή των Κοινοτήτων δεν μπόρεσε να φτάσει σε θέση. Εμείς ε, έπρεπε να στηρίξουμε την ε, ενότητά μας, μια ενότητα που δείξαμε, επιδείξαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ε, και ε, η θέση που θα πάρουμε, ε, ειδικά για, την, για κάποιες θέσεις, για κάποιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης Βρετανών. Πέντε εκατομμύρια Βρετανών επισκέπτονται τα Κανάρια. Ελπίζω η συζήτηση όμως να δείξει ότι όταν κάνουμε, έχουμε δικαίωμα, όταν τους δίνουμε ε, επεκτάσεις, να κάνουμε ερωτήσεις τουλάχιστον. Και οι ερωτήσεις μας αυτές θα πρέπει να παίρνουν και απαντήσεις. Τους δώσαμε παράταση, αλλά γιατί, για ποιο λόγο. Ο κ. Πολτσακ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κ. Πόπα, είναι αξιολύπητο το, γεγονόν, το γεγονός ότι σε αυτή την προεκλογική εξατία κόμματα και πολιτικοί στοχεύουν αντίον της Ρουμανίας και μας βάζουν στο σκαμνί. Είναι απαράδεκτο. Ακόμα μία φορά ε, μας επικρίνουν αδίκως εμάς τους Ρουμάνους. Οι Ρουμάνοι είναι θύματα τέτοιων επιθέσεων. Μιλάτε για τις δικές μας διαφθορές, αλλά δεν μιλάμε για, άλλες, για τις διαφθορές σε άλλες χώρες. Ε, αυτό που με ενοχλεί είναι ότι αυτές οι επικρίσεις δεν αναφέρονται με συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά με γενικολογίες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η, δεν θα πρέπει η προεκλογική εκστρατεία να επηρεάζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ε, με τέτοιου τύπου επιθέσεις και τέτοιου τύπου εκστρατείες. Ο κ. Σκρίπεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από λίγο μάθαμε ότι στην Ισπανία υπάρχει μια επιτροπή ε, στα σχολεία για την ισότητα των φύλων όπου ε, εξετάζει το κατά πόσον τα παραμύθια είναι σεξιστικά. Με εντυπωσιάζουν αυτές οι ιστορίες. Γιατί γενναίες επιγενεών ευρωπαϊκά παιδιά ανατράφηκαν ακούγοντας αυτά τα πανέμορφα παραμύθια με αξίες ε, για τη ζωή, για την αντιπαράθεση καλού και κακού. Μιλάμε για τις αξίες που σφυριλατούν τον άνθρωπο, για το τι είναι, του μαθαίνουν τι είναι καλό στη ζωή και τι είναι κακό στη ζωή. Επομένως, μου, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να αρνηθούμε αυτές τις τάσεις, να τις καταπολεμήσουμε. Δεν είναι σωστό ως κράτος να λέμε τι, τι παραμύθια θα πρέπει να ακούνε τα παιδιά. Τα, οι γονείς σας αποφασίσουν τι παραμύθια θα τους πούν. Ευχαριστώ κύριο Σελίμωβιτς. E Υπάρχει μεγάλη στήριξη για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 65% των Σουηδών πιστεύουν ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και σφιγμομετρήσεις που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χαίρεται τη εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν πιστεύουν οι πολίτε ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, η Ευρώπη τα προβλήματά του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ένα σχέδιο πάρα αυτά, ούτω ώστε να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργεί. Θα πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών τη. Γιατί αν δεν τα καταφέρει, τότε θα επηρεαστεί και αυτό το κοινοβούλιο με εξτρεμιστέ ε, και σε όλο το φάσμα αλλά και με επικύλα προβλήματα. Θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες λοιπόν ότι τους ακούμε, ακούμε αυτά που μας λένε και ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι για τα προβλήματα που έχουν στην καθημερινότητά τους για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Ο κύριος Τερικάμπρας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα προς τέλος της θητείας μας να μιλήσω Ολλανδικά. Είμαι καταλληνός, βεβαίως. Η Ισπανική κυβέρνηση δεν μου επιτρέπει να χρησιμοποιώ τη γλώσσα μου. Το Βέλγιο όμως είναι μια χώρα στην οποία κάποιος μπορεί να μιλήσει ελεύθερα γαλλικά, φλαμαδικά, γερμανικά. Προσπάθησα να μάθω τα Ολλανδικά όσο πιο καλά μπορούσα. Οπότε στη γλώσσα αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτερ, τον δασκαλό μου, ο οποίος μου επέτρεψε να σημειώσω πρόοδο στην γλώσσα αυτή. Αυτό θέλω να καταθέσω. Υπέρ της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Ελπίζοντας ότι σύντομα τα καταλανικά θα είναι επίσημη γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την Πρόεδρο. Ένα από τα θέματα αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας ε, που τελειώνει είναι η Καταλωνία. Πολλοί από εσάς ανακαλύψατε μια χώρα ε, η οποία θέλει να ανακαλύψει το μέλλον της με αυτοδιάθεση ε, και γι' αυτό μας επιτέθηκαν επιτέθηκαν σε ψηφοφόρου, μόνο και μόνο γιατί πήγαν να ψηφίσουν, μας επιτέθηκαν γιατί οργανώσαμε ένα ε, δημοψήφισμα και μα αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε εγκληματίες. Εμείς οι Καταλανοί όμως θα ανακαλύπτουν και κάτι άλλο, την υποκρισία της Ευρώπης. Στο μεταξύ, όλε οι επιθέσει εναντίον μα πολλαπλασιάστηκαν. Ε, στο μεταξύ, οι Ισπανοί, που είναι, οι Καταλανοί μάλλον, που είναι υπέρ τη ανεξαρτησία, αποδεσμεύονται λιγάκι από την ε, Ευρώπη. Ποιε είναι οι ευρωπαϊκέ αξίε, θα επανέλθουμε μεγαλύτερη δύναμη για να διεκδικήσουμε από την Ευρώπη ελευθερίε και δικαιώματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να μα τα είχαν αρνηθεί. Μακάρθη. Η Κομισιόν θα δώσει 13 δισεκατομμύρια τα επόμενα 5 χρόνια για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Εφημισμό. Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό στρατό. Τη στιγμή που η δημόσια σε χώρε όπω στην Ιλλανδία έχουν φτάσει στα άκρα. Το ΣΥΝΦΕΙΝ θα αντιδράσει στην αύξηση της συμμετοχή της χώρας στον Ευρωπαϊκό Προπολισμό, αν είναι να χρηματοδοτήσουμε μια πολεμική μηχανή. Θέλουμε να είμαστε ουδέτεροι, να κρατήσουμε τα χρήματά μας, να είμαστε ασφαλείς, να διασφαλίσουμε την διεθνή μας φήμη. Θέλουμε να διαδραματίσουμε θετικό ρόλο για την ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Το Φίνα και το Φίνα Γκέιλ μια πρόταση, η οποία θα επέτρεπαν στον ελληνικό λαό να παραμείνει ουδέτερος. Χάσαμε μια ευκαιρία να υπερμηνθούμε της αξιοπρέπειάς μας. Και αντί αυτού χρηματοδοτούμε έναν Ευρωπαϊκό στρατό. Το Σινφέιν δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτά τα σχέδια κατά τη ουδετερότητα τη Ιρλανδία και θα το κάνουμε αυτό κάθε μέρα, για πάντα. Κύριε Φλάνναγκεν. Κύριε Πρόεδρε, ψηφίσαμε για τις ενισχύσεις στην Επιτροπή Γεωργίας δώσουμε 150 εκατομμύρια για μια περιοχή στο κέντρο της Ιρλανδίας. Ως το 2026 θα έχουμε δώσει διάφορα εκατομμύρια σε επιμέρους περιοχές στην ε, Ιρλανδία. Μοιράζουμε δεκάδες εκατομμύρια αριστερά και δεξιά και παρά τα νούμερα αυτά, παρά τις χρηματοδοτήσεις, δύο πράγματα βλέπουμε εν τέλει δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση για τις περιοχές που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να σας συστήσω ένα action film. Έχει τον τίτλο Collateral Murder και μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Ε, η παραγωγή είναι ο Αμερικανικός στρατός ε, και δημοσιεύτηκε από το Wikileaks ε, του Assange. Βλέπουμε λοιπόν εκεί Αμερικανούς στρατιώτες οι οποίοι από ελικόπτερα ε, πυροβολούν κατά των αμάχων παιδιά, αθώοι πολίτες και το χειρότερο από όλα το διασκεδάζουν. Υπάρχει λοιπόν ένα έγκλημα και ο άνθρωπος που το δημοσιοποίησε κινδυνεύει να εκδοθεί τώρα στους ανθρώπους οι οποίοι συγκαλύπτουν όλα αυτά τα γεγονότα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγο καιρό συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο σχετικά με τους καταγγέλλοντες, τους whistleblowers. Κατά τη δική μου άποψη αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο το να ταπεινώνει κανείς ανθρώπους και να διασκεδάζει. Και να πω κάτι άλλο στους Βρετανούς. Αν εσείς τελικά εκδώσετε τον Julian Assange στις ΗΠΑ, να ξέρετε ότι θα έχετε το σκληρότερο Brexit που μπορείτε να φανταστείτε. Κιού μόνο μόνον αυτό, αλλά και χωρίς καμία καθυστέρηση. Σωσνίτς, κύριε Πρόεδρε, το πιο δύναμο σημείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η νομοθετική διάρκεια. Εκδίδουμε 500 κείμενα το χρόνο, πάνω από ένα την ημέρα, τα οποία δεν διαβάζει κανείς. κανείς δεν μπορεί να τα διαβάσει, γιατί οι άνθρωποι έχουν τις δουλειές τους. Δεν ενδιαφέρονται να διαβάσουν αυτά τα οποία εκδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ψηφίζουμε, επί τροχάδιν, πολλές φορές ε, οι ψηφοφορίες μας γίνονται με τέτοια ταχύτητα. Έχουμε καμιά φορά λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα ανατροπολογία. Πολλές φορές ο πρόεδρος δεν κοιτάζει καν ποιος ψηφίζει τι κοιτάζει μόνο τα χέρια των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων και πολλές φορές άλλοι ψηφίζουν για λογαριασμό άλλων συναδέλφων, κάτι το οποίο είναι απολύτως απαράδεκτο. Εν ώψη αυτών των παρατυπιών ζήτησα από εμπειρογνώμονες να εκδώσουν έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν ε, ετοιμαστεί αυτή η έκθεση, θα σταλεί σε όλου, θα μεταφραστεί και ελπίζω ότι θα βάλουμε τα πράγματα κάποια στιγμή στη θέση του. Κύριε Κοράτσα Κύριε Πρόεδρε, τα δικαιώματα των παιδιών δεν είναι αμεληταίο θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Η μεικτή ομάδα για τα δικαιώματα των, παιδιού, των παιδιών κάνει ό,τι μπορεί για να τεθεί το θέμα στο κέντρο της δράσης μας. Ένα μόνιμο σώμα, μια μόνιμη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Η δική μου προτεραιότητα ήταν να πατάξουμε κάθε μορφή βίας κατά των παιδιών, κατά των παιδιών μεταναστών. Κάναμε πολλά πράγματα σε συνεργασία με το Συμβουλίο της Ευρώπης. Ενισχύσαμε τη συνεργασία μας για να προστατεύσουμε τα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ, στο Κοινοβούλιο, δημιουργήσαμε έναν δίκτυ σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών σε ζώνες πολέμου Πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα. Την επόμενη θητεία, Καλό την Επιτροπή να εγκρίνει ένα νέο θεματολόγιο για τα δικαιώματα των παιδιών, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, στο πλαίσιο του GDPR, μια οδηγία για την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Γιατί ποτέ δεν θα έχουμε κάνει αρκετά για τα παιδιά. Καλό όλου του υποψηφίου, να συνταχθούν με τη δεσμευσή μα Και ε, ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, να δεσμευτούμε όλοι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Κ. Μαυρίδης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η τουρκική κατοχή της Κύπρου συνεχίζεται και είναι ένα έγκλημα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όμως το προβάλαμε πριν πέντε χρόνια σε αυτή εδώ την αίθουσα, ελάχιστη έδινα σημασία. Όταν ο Ερτογάν προχώρησε και συνέτριψε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ίδια την Τουρκία, όταν φυλάκιζε όποιον διαφωνούσε μαζί του αυξάνονταν όσοι έδιναν σημασία αλλά κάποιοι έβρισκαν λόγους να τον υποστηρίζουν. καθώς μιλάμε όμως στην ανατολική μεσόγειο η κυπριακή δημοκρατία επιχειρεί να αξιοποιήσει τα ενεργειακά της αποθέματα προς όφελος της ευρωπαϊκής ένωσης. νομίζω έφτασε η ώρα και θα κριθούμε όλοι μας στην πράξη θα στηρίξουμε την κυπριακή δημοκρατία και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας ή θα βρούμε πάλι λόγους να στηρίξουμε την τουρκία. ενώ η τουρκική κατοχή στην κύπρο συνεχίζεται η ευρώπη παραμένει ακροτηριασμένη και στην πολιτική κρινόμαστε για τη διορατικότητά μας. ας βάλουμε επιτέλους μπροστά απ' όλα την ίδια την ευρώπη και όχι οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ που μου δίνουν το λόγο. Σε, σε δύο μήνες, από 1η Μαρτίου που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μίλησα για πολλά θέματα. Τώρα θα μιλήσω για ένα δικαίωμα, το δικαίωμα να πεθάνει κανείς με αξιοπρέπεια. Στην Ισπανική Δημοκρατία έγινε μια πολύ ε, σημαντική συζήτηση για την ευθανασία μια συζήτηση όπου το, ένα άτομο, ο άντρα μιας κυρίας με μια πολύ σοβαρή αναπηρία, θέλει να τη βοηθήσει για να πεθάνει με αξιοπρέπεια. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δικάζεται αντιμετωπίζει μια σοβαρή κατηγορία. Το άτομο αυτό ζούσε στο Βέλγιο. Ε, αν το άτομο αυτό μάλλον ζούσε στο Βέλγιο, θα είχε τελείω διαφορετικά δικαιώματα. Γιατί το Βέλγιο αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ευθανασία. Θα ήθελα να πω λοιπόν στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο ότι πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση στην Ευρώπη για την ευθανασία σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι ευρωπαϊκό θέμα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ευχαριστώ ξάκι. Κυρία Πρόεδρε, οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι πρώτον πυλών και συζητάμε ε, πολύ συχνά για τα ακραία κόμματα και εγώ νομίζω ότι δεν αρκεί απλά να συζητάμε για τα κόμματα αυτά γιατί και κόμματα που εκπροσωπούνται εδώ στηρίζουν ακραίες απόψεις δυστυχώς και στη δική μου την πατρίδα την Τσεχοσλοβακία το κόμμα Most Hit και το κόμμα Smer αυτά έχουν συστήσει συμμαχία με ένα εθνικιστικό σλοβακικό κόμμα. Ε, το βρίσκω πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό, γιατί αυτό το ε, επίπεδο των εθνικιστών είναι πολύ χαμηλό και έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ το κράτος δικαίου, ήδη δολοφονήθηκε ένας δημοσιογράφος και τώρα πια δεν επιτρέπεται να ανακρούονται οι ύμνοι άλλων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιο ανακρούει τον ύμνο ε, άλλου κράτου μέλους τη Ευρωπαϊκή Ένωση. καλύτερα να πληρώσει πρόστιμο 7.000 ευρώ. Ο Τανουσέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι παρά τις ε, διαφορετικές πολιτικές απόψεις, ε, το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωράει και είμαστε κοντά στην Ευρώπη της συνοχής. Είναι η πρώτη φορά όπου η πολιτική συνοχή είναι το σημαντικότερο. Για την περιοδο 2021 2021-2027 το θέμα της συνοχής το ε, συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ε, θα χρηματοδοτηθεί με 317 δις ευρώ. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα έλαβαν περισσότερα κονδύλια και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, για χώρες οι οποίες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι καλές ε, ενδείξεις. Ε, η συζήτηση που είχαμε τα τελευταία χρόνια για το μέλλον της Ευρώπης, παρόλα αυτά είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε, να συμβιώσουμε, γιατί μια ενωμένη Ευρώπη είναι ο τελικός μας στόχος. Ο κύριος Πολτσακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ε, υποστήριξή μου στο λαό της Γαλλίας λόγω της ε, τραγωδίας ε, που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή η Notre Dame, η Παναγία των Παρισίων, αποτελεί μέρος της ε, πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ελπίζω οι πυροσβέστες να μπορέσουν να σώσουν αυτό τον καθεδρικό ναό. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Μετανάστευση, ρήπανση του περιβάλλοντος. Κατά τη δική μου όψη το σημαντικότερο όλων είναι η κλιματική αλλαγή οφείλουμε να το λάβουμε αυτό υπόψη μας ε, γιατί η αδυναμία μας να το αντιμετωπίσουμε μπορεί να αποβεί μοιραία. Καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε την ξηρασία. Ε, εξάλλου πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ύπεθρο, ε, να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Ε, η ρήπανση είναι καθοριστική σημασίας. Ε, μόνο από κοινού θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις και ελπίζω τελικά να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η τελευταία περίοδος αυτών των σύντομων παρεμβάσεων σε αυτή τη θητεία. Ε, εγώ προσπάθησα να εκπροσωπώ καλύτερα μπορούσα τη χώρα μου. Εδώ πέρασα πάρα πολλές ώρες και είμαι πολύ περήφανος που μπόρεσα να είμαι ένας από τους πιο παραγωγικούς και παρόντες βουλευτές. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην εκλογική μου περιφέρεια ε, για να μπορέσω να μεταφέρω την ιδέα ότι η Ευρώπη ε, ο ιδέα έχει οριμάσει. Μια Ευρώπη της ειρήνης για, του, για όλους, αλλά και η φιλοδοξία να είμαστε τα ενωμένα κράτη της Ευρώπης. Ε, είναι μια πολύ δύσκολη όλη αυτή η περιοχή. Είναι μια περιοχή η οποία δεν ξέρω αν τους αξίζει πραγματικά αυτό το όνομα, γιατί πάρα πολλοί δυστυχώς ε, παραπλανούν τους πολίτες. Εγώ απευθύνομαι λοιπόν στους ψηφοφόρους. Ας σεβαστούμε στην περιοχή μα, α μπορέσουμε να σταθούμε στο ύψο των περιστάσεων τη προεκλογική εκστρατεία, ε, α θελήσουμε να βασιστούμε στην ε, ιδέα ότι ζήτω η Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτω η Ιταλία, ζήτω η Νότιο Ιταλία. országom polgáraként fájdalommal élem meg κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω με μεγάλη ανησυχία ε, διαπιστώνω ότι ε, για τρίτη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι το θέμα της Ρουμανίας στη μέση διάταξη. Εγώ είμαι Ούγγρος, ανήκω στην Ουγγρική μειονότητα της Ρουμανίας και γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας υπενθυμίσω την εχθρότητα της Ρουμανίας έναντι των μειονοτήτων. Αυτό είναι και παραβίαση του κράτους δικαίου. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σιωπά. Εγώ λοιπόν συγκεκριμένα απαιτώ να αφαιθούν ελεύθεροι δύο Ούγγροι, οι οποίοι συνελήφθησαν από το μετακομμουνιστικό καθεστώς, απλά και μόνο λόγω της εθνοτικής τους προέλευσης. Ο Μπέκε και ο Σέλτς, ο δήμαρχος του Κορούν, λόγω του ότι χρησιμοποιεί την ουγγρική γλώσσα, του επευλήθη πρόστιμο 100.000 ευρώ. Θα ήθελε λοιπόν να αρθεί και αυτό το πρόστιμο. Και για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδου περιπτώσει, ζητώ την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Αν και είναι η τελευταία μου ομιλία ενός λεπτού κατά τη διάρκεια της πρέπει να αλλάξω θέμα. Θα μιλήσω για την πυρκαγιά στο Παρίσι. Εν ώψη της πυρκαγιάς στην Νότερνταμ, στον Καθεδρικό των Παρισίων, θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου. Γνωρίζω πολύ καλά το σύμβολο αυτό της χριστιανικής πίστης στο Παρίσι. Ένα σύμβολο της ιστορίας μας, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ελπίζω ότι το μνημείο αυτό θα επισκευαστεί σύντομα Ελπίζω επίσης ότι θα είμαστε σε αυτό όλοι ενωμένοι, ότι θα επιδείξουμε καλή θέληση. Ελπίζω το φως της Dame να μας ε, εξηγείρει να συνεγερθούμε και να ξαναδούμε σύντομα την η υπερήφανη όπως ήταν πάντα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα λόγια που μόλις τώρα απευθύνατε στην Ολομέλεια. Πραγματικά αυτό που διαδραματίζει αυτή τη στιγμή είναι τραγωδία. Εγώ έχω μεγαλώσει στο Παρίσι και έχω επισκεφτεί αυτόν τον καθεδρικό ναό επανειλημμένα. Ο ναός αυτός είναι θησαυρό και θέλω να ελπίζω ότι θα καταστεί δυνατόν να διαφυλαχθεί αυτός ο θησαυρό και θα καταστεί επίσης δυνατόν να σβήσει όσο το δυνατόν συντομότερα η επόμενη συνεδρίαση λαμβάνει χώρα αύριο το πρωί, Τρίτη. Ε, το πρωί ξεκινάμε στις 9 η ώρα. Έχει δημοσιευτεί η μερίσια διάταξη. Μπορείτε και να την βρείτε και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν λοιπόν κλείσουμε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παριστάμενους που παρέμειναν εδώ μέχρι αυτή την τόσο προκεχωρημένη ώρα. Ευχαριστώ τους και τις διερμηνείς, ε, τους συναδέλφους και τους ε, συνεργάτες μας, ε, τους ΟΙΣΧΕ, γιατί είναι πολύ σημαντικοί γιατί είναι πολύ σημαντικοί για να μπορούμε και εμείς